and emissions in the automotive sector in the EU. Αφορά την, ε, ε, τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ένωση. Έχουμε στείλει γραπτές ερωτήσεις στον κύριο Φάλκενμπεργκ, πράγμα που μπορούμε να, ερωτήσεις που μπορούμε να βρούμε μαζί με τις απαντήσεις του κύριου Φάλκενμπεργκ στο ντοσιέ το ηλεκτρονικό που σας έχει σταλεί. Έχουμε μια μισή ώρα για την συζήτηση. Θα σας δώσω κύριε Φάρκε, με το λόγο για να κάνετε την εισήγησή σας και έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και αγαπητά μέλη της Επιτροπής εμείς σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να διευκρινίσω το ρόλο μου και το ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η θητεία μου ως Γενικό Διευθυντή σε μεγάλο βαθμό συμπίπτει με τη θητεία του Γιάννη Σποτότσνη ως Επιτρόπου που ήδη είδατε. Ξεκίνησα την υπηρεσία με το Σταυροδήμα με πρώτο θέμα ενδιαφέροντος το, τις κλιματικές αλλαγές και με τον Επίτροπο Βέλα το 2015 έληξε η θητεία μου. Δεν θα σας καθυστερήσω περισσότερο Θα ήθελα να αναφερθώ περισσότερο στις πολύ σημαντικές πολιτικές τοποθετήσεις του Επιτρόπου Ποτότσνικ, γιατί εργαστήκαμε στενά για να ε, βρούμε ένα καλύτερο, μια καλύτερη λύση για τη βελτίωση της ατμοσφαιρικής ε, Τη ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και να αντιμετωπίσουμε ορισμένα από τα ζητήματα ω προ την υλοποίηση τη περιβαλλοντική νομοθεσία Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υλοποίηση λοιπόν ξεκινά με την ποιότητα και την ευκρίνεια τη ίδια τη νομοθεσία, πράγμα το οποίο αποτελεί πάντοτε βέβαια πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και για του δύο συνομοθέτε, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Δεύτερον, απαιτεί μια ξεκάθαρη αντίληψη του πόσο η κοινή νομοθεσία που δεσμεύει όλα τα κράτη-μέλη για το καλό των 500 εκατομμυρίων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιείται και από ποιον. Η αρχή της επικορικότητας είναι μια πολύ θετική αρχή, αλλά προκειμένου να μπορούν 28, οι αρχές 28 κρατών μελών να εφαρμόζουν με την ίδια ένταση ε, την νομοθεσία αυτή, χρειάζονται κοινοί κανόνες και αναθεώρηση. Βλέπουμε πολλές φορές ότι δεν υπάρχει λύση για τον πολίτη παρά να ενημερώσει την Επιτροπή σε σχέση με ελλείμματα ή προβλήματα ως προς την υλοποίηση από τα επιμέρους κράτη-μέλη των ε, διατάξεων των σχετικών με την περιβάλλον. Έχει έτσι δεχθεί πάρα πολλές ε, προσφυγές από πολίτες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα το δικαστήριο βεβαίως κυρίως ε, από παράπονα των πολιτών. Έχουν διατυπωθεί βέβαια προτάσεις για τη βελτίωση, την ενίσχυση της υλοποίησης και έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα παρακολούθησης κατάστασης μαζί με μια καλύτερη πρόσβαση για τον πολίτη σε εθνικά δικαστήρια, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Το θέμα που σας απασχολεί ε, σήμερα κινείται γύρω από αυτά τα ζητήματα. Γνωρίζω λοιπόν ότι υπάρχουν αποκλήσεις μεταξύ των δοκιμών σε εργαστήριο και των πραγματικών εκπομπών. Έχω ακούσει τριών διαφορετικών τύπων εξηγήσει. Καταρχά ότι οι εκπομπέ του ιδιωτικού οχήματο μπορεί να εξαρτώνται από τη συμπεριφορά του οδηγού. Μέχρι 30% τη κατανάλωση σε καύσιμα και ω κρούτου και τη μόλυνση μπορούν να εξηγηθούν από την ε, οικολογική ημί. Ε, οδήγηση, δεύτερον ε, σε εργαστηριακές συνθήκες όπως ορίζεται με, την, ε, με το τεστ NEDC μπορεί να υπάρξει δυνατότητα για περαιτέρω βελτίωσης των εκπομπών και τρίτον μπορεί να υπάρχουν και κάποιες εξηγήσει για το πώς μπορούν να καταστούν τα ιδιωτικά οχήματα πιο καθαρά εάν αλλά, αλλά μπορεί να οφείλεται η, εξακολουθ... η διαρκή κακή κατάσταση του ατμοσφαιρικού αέρα σε μεγάλε πόλει Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να οφείλεται λοιπόν στον όλο και μεγαλύτερο αριθμό οχημάτων που κινούνται στου δρόμου των πόλεων μα. Για μένα η απουσία πραγματικής βελτίωσης σχέση με τι εκπομπέ ε, οξυδίου του αζότου και μικροσωματιδίων στον ατμοσφαιρικό αέρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν το κύριο ζήτημα, το κύριο μέλημα με το οποίο ασχολήθηκα και εγώ κατά τη θητεία μου. Ο τομέα των μεταφόρων συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό κατά το 1 τρίτο συγκεκριμένα στην ναι. συμβάλλει λοιπόν κατά το 1 τρίτο στην ε, ε, μόλυνση του ατμοσφαιρικού αέρα και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη Γενική Διεύθυνση για το Περιβάλλον πίεσε για πιο αυστηρία όρια ιδιαίτερα από τους κινητήρες με πετρέλαιο. Σημειώσαμε ότι η ανακοίνωση CARS 2020 ε, έχει ιδιαίτερα επιμείνει ως προς το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Έχουμε πιέσει για την ε, υιοθέτηση ε, συστημάτων ελέγχου σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Το ΚΑΡΣ 2020 όρισε ένα χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή του νέου συστήματος σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης με την εφαρμογή με την παράλληλη εφαρμογή τη προδιαγραφής Euro 6, δηλαδή το Σεπτέμβριο του 2014, θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια, πρόταση έως τα τέλη του 2013, προκειμένου να τηρηθούν αυτές οι ε, προθεσμίες, υποκανονικές συνθήκες. Η τεχνολογική, η τεχνική δουλειά χρειάστηκε περισσότερο και αυτό εξηγεί και γιατί ε, η επιστολή μου επισήμανε το κατεπήγον της υπόθεσης προς τον ε, Γενικό Διευθυντή Καλέχα. Η ανάγκη αυτή λοιπόν για κατεπήγουσα δράση ιδιαίτερα επιτάθηκε και από τη μελέτη ICCT που σημειώνει ακόμη ψηλότερες αποκλίσεις. Έτσι λοιπόν, εάν ε, μπορεί ακόμη να είναι τεχνικά δυνατό με την επιστολή εφαρμοστικής πράξης να, καταστεί, να καλυφθούν οι προδιαγραφές του Euro 6, αλλά παραμένει το ζήτημα εάν η ερμηνεία της ε, εφαρμοστικής πράξης μπορεί να δικαιολογήσει η κοσαπλάσια υπέρβαση προδιαγραφών που ορίζει ο νόμος. Οι αρμόδιε αρχέ λοιπόν των κρατών μελών θα έπρεπε να έχουν αξιοποιήσει τα μέτρα επιτήρηση αγορά και να αμφισβητήσουν την ε, ε, αιτιολογία τέτοιου είδου ε, εγκρίσεων τύπου. Ελπίζω όλοι οι φορείς να καταλήξουν, τόσο τα κρατημέρια δηλαδή όσο και τα θεσμικά όργανα, να καταλήξουν τα κατάλληλα συμπεράσματα σε σχέση με αυτό το σκάνδαλο εκπομπών από πετρελαιοκινητήρε. Το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι δεν αρκεί μόνη η νομοθεσία, χρειάζεται σαφής μηχανισμός ανεξάρτητης επιτήρησης και παρακολούθησης της πραγματικής υλοποίησης νομοθεσίας και έγκαιρη συντονισμένη δράση όταν διαπιστώνονται αποκλήσεις σχέση με τους όρους της νομοθεσίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε θα ξεκινήσουμε τον πρώτο γύρο ερωτήσεων και θα ξεκινήσουμε με τους εισηγητές και στη συνέχεια θα έχουμε έναν εκπρόσωπο από κάθε πολιτική ομάδα με ε, δικαίωμα ομιλία για πέντε λεπτά για την ερώτηση και την απάντηση. Ο κύριος Μπράντε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ κύριε Φάλκεμπερ. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω εδώ. Ε, η ερώτησή μου είναι η εξή. Όταν ε, κανεί εξετάσει την, την, τα ανακοινοθέντα τη Επιτροπή, είτε πρόκειται για γραπτέ απαντήσει ή για άλλου είδου δηλώσει εδώ, ε, φαίνονται όλα να είναι συνεπή ή είναι η ίδια απάντηση κάθε φορά. Όμω γνωρίζουμε ταυτόχρονα ότι για χρόνια συνεπει η ειναι η ιδια απαντηση καθε φορα τμήματα τη ε, Επιτροπή έχουν ε, έρθει σε αντιπαράθεση για αυτό το θέμα. Είδαμε ανταλλαγές επιστολών από εσά, α πούμε, προς τον συνάδελφό σας ε, Καλέχα, ε, επιστολή του Επιτρόπου Ποτότσνικ προς τον Επίτροπο Ταγιάννη. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε κάποια περισσότερα πράγματα για το τι γινόταν εσωτερικά και το τι ακριβώς ήταν γνωστό. Γιατί τώρα παίρνουμε ανταλλαγές email από την DG Enterprise, την DG Κλίμα, την DG Περιβάλλον με το JRC, το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο, ήδη από το 2008, όπου υπήρχαν ισχυρές υποψίες, έντονες υποψίες για τη χρήση συσκευών αναστολής και έτσι γίνεται, καθίσατε δύσκολο να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στις συσκευές αναστολής και το cycle beating, την υπέρβαση του κύκλου. Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν τι, συνέβαν, τι συνέβαινε. Η ερώτησή σας αφορά χρόνο που ήταν πριν από τη δική μου άφηξη ως Γενικού Διευθυντή, γιατί στην προετοιμασία αυτής της ακρόασης κατέστη σαφές για πολλούς συναδέλφους στην ε, ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ περιβάλλον ότι υπήρχε πρόβλημα ανάμεσα στις εργαστηριακές δοκιμές και τις ε, πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Επανήλθαμε στις προδιαγραφές Euro 5 για την περίοδο μάλλον μέχρι το 2005. Αυτό το οποίο νομίζω δεν ήταν σαφές ήταν ο βαθμός στον οποίο ε, υπάρχουν αυτές οι διαφορές, υπήρχαν μάλλον αυτές οι διαφορές και υπήρχαν ε, ίσως εξηγήσεις για το τι, γιατί συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ένα αυτοκίνητο εκπέμπει διαφορετικά ρήπους ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιείται. Οπότε δεν ε, είναι λες και οποιοδήποτε αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε οδηγητική συνθήκη θα συμπεριφερθεί ακριβώ με τον ίδιο τρόπο. Μικρέ αποκλήσει δηλαδή είναι φυσιολογικό να υπάρχουν. Ανέφερα ότι μέχρι 30% μπορούσε να εξηγηθεί και έχει εξηγηθεί από την στάση την οικολογική, δηλαδή δεν πατάς και τόσο τον γκάζι, προσπαθείς να είσαι λίγο πιο λογικός ως οδηγός. Εκεί μπορεί να υπάρξουν μικροαποκλήσεις. Μετά αρχίσαμε στην DG Περιβάλλον να κάνουμε μια μελέτη μαζί με το JRC για να έχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια για το ποιες ακριβώς είναι αυτές οι διαφορές και για, σε τι οφείλονται. Να τις καταλάβουμε καλύτερα. Και νομίζω ότι εξ αρχής το είδαμε αυτό γιατί είδαμε στο τέλος ότι η ποιότητα του αέρα για την οποία εμείς είμαστε υπεύθυνοι δεν βελτιωνόταν στις πόλεις μας. Οπότε Κάναμε αυτή τη μελέτη και η μελέτη μας έδωσε περισσότερες ενδείξεις ότι υπήρχαν ε, αποκλήσεις, διαφορές και μάλιστα διαφορές δυσεξήγητες. Εγώ ο ίδιος όμως όλο αυτό το διάστημα, το χρονικό, δεν είχα σκεφτεί ότι μπορεί να υπάρχουν παράνομες πρακτικές. Εγώ η καλύτερη αναλογία παρομοίαση που μπορώ να σας δώσω είναι η φορολογική νομοθεσία όπου έχει κάνει τη τάση για φορολογική βελτιστοποίηση. Δηλαδή οι διάφοροι ε, ε υπόλογοι, φορολογούμενοι, προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν κάθε δυνατή εξήγηση για να μειώσουν τους φόρους που θα πληρώσουν. Και νομίζω πως έτσι χρησιμοποιήθηκε. Δηλαδή νομικός ορθή αλλά ηθικός λάθος. Εντάξει, τώρα το <laughs> ηθική τώρα αιτιολόγηση, επειδή μιλάμε για νομική επιβολή, επιβολή μάλλον του νόμου, δεν νομίζω πως είχαμε πραγματικά εδώ νομική ε, στοιχειοθέτηση υπόθεση εδώ. Ε, αλλά έπρεπε να καλύψουμε οποιασδήποτε κενά παραθυράκια υπήρχαν. Να κοιτάξτε, τα πέντε μας λεφτά είναι σχεδόν, ε, έχουν σχεδόν τελειώσει, αλλά θα πρέπει να ήταν πολύ δύσκολη η θέση σας στην DGNG, και κατά κάποιο τρόπο, γιατί θέλατε να βελτιωθούν τα πράγματα, αλλά δεν ε, λειτουργούσε το σύστημα. Το JRC ε, είχε ήδη αποφασίσει από το 2011 ότι οι φορητές συσκευέ ελέγχου μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, αλλά και κάποια χρόνια ακόμα συνεχίστηκε η χρήση των παλιών τεστ να Ενώ υπήρχαν εναλλακτικέ, πράγμα το οποίο καθυστέρησε τη διαδικασία. Είχατε ποτέ την αίσθηση ότι υπήρχαν κάποιε δυνάμει, α πούμε, η κακή κατάσταση της αυτοκινητοβιομηχανίας εκείνα τα χρόνια που πίστευαν ότι οι οικονομικές συνέπειες ήταν πολύ πιο σημαντικές από ότι οι συνέπειες της κακής ποιότητας του αέρα και τα νομικά όρια που είχαμε θεσπίσει παλιότερα. Κοιτάξτε, είναι σαφώς μια περίοδος όπου υπήρχαν πολλές, πολλοί οικονομικοί προβληματισμοί. Είναι επίσης αλήθεια και μάλλον πολλά μέλη εδώ θα θυμάστε ότι όταν υποβάλαμε την πρόταση για την ποιότητα του αέρα, έπρεπε να προσπαθήσουμε πολύ για να πείσουμε ότι το θέμα της ποιότητας του αέρα είναι σοβαρό και ότι έπρεπε να αντιμετωπιστεί ακόμα και σε χαλεπούς οικονομικούς καιρούς. Πιστεύω πως ναι, υπήρχαν στιγμές όπου επικρατούσε σύγχυση, απόγνωση. Από την άλλη πλευρά γίνονταν και βήματα, ας πούμε η ανακοίνωση ΚΑΡ 2020 μας έδωσε ένα πρόγραμμα δράσης και εγώ έχω εργαστεί πολύ ώστε να πιέσω για την εφαρμογή αυτού του σχεδίου δράσης. Τελικά δεν καταφέραμε να το κλείσουμε θα έπρεπε να είχαμε το, τη δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες το RDE ε, εγκαίρος. θα έπρεπε να το είχαμε από το Σεπτέμβριο του 2014 και δυστυχώς περάσαμε σε αυτό μόνο το 2015. Ε, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι το επιανελειμμένο εργαζόμουν και θυμίζα συνέχεια στον Επίτροπο Ποτότσνικ, αλλά και με τους συναδέλφους ολόκληρη την Κομισιόν και επιμείναμε ότι έπρεπε να, να επιταχυνθεί η διαδικασία και αυτό ήταν όλο ένα και μεγαλύτερη ανησυχία. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερος μας εισηγητής δεν έχει φτάσει ακόμα, οπότε θα περάσουμε στον κύριο... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς κύριε Γενική Διευθυντά. Ο η συγκεκριτή μα ε, βρίσκεται ακόμα στο αεροπλάνο, αλλά θα μπορέσει νομίζω να υποβάλει μετά ερωτήσεις. Σχεδόν δεύτερο, κάθε δεύτερο, κάθε ένα αυτοκίνητο στα δύο δηλαδή, είναι αυτοκίνητο diesel. Αλλού είναι αλλιώ. μόνο 3%. Ε, πώς εξηγείται αυτή η διαφορά. Φάλκενμπερκ. Νομίζω ότι αυτό έχει μεγάλη σχέση με το γεγονός ότι στην Ευρώπη αντιμετωπίσαμε πιο συνειδητά την αλλαγή στο κλίμα, την αλλαγή της αλλαγής του κλίματος δηλαδή. Το δε καύσιμο ντίζελ θεωρούνταν το πιο αποδοτικό καύσιμο και επομένως αυτό το οποίο εκλείει και λιγότερο διοξίδιο του άνθρακου στην ατμόσφαιρα. Νομίζω μάλιστα ότι έχουν δοθεί και φορολογικά κίνητρα υπέρ του καυσίμου ντίζελ κάτι που οδήγησε στα τελευταία 25-30 χρόνια ο ευρωπαϊκός στόλος αυτοκινήτων όλο και περισσότερο να κατευθυνθεί προς το καύσιμο δίζελ. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε με τον τρόπο αυτό στις αλλαγές του κλίματος και ότι ίσως θα έπρεπε να είχαμε προσέξει περισσότερο το γεγονός ότι στον ατμοσφαιρικό αέρα που όλοι αναπνέουμε και στις πόλεις και στην Ήπεθρο ότι οι ε, εκπομπές ε, καυσαερίων του ντίζελ ε, σημαίνει και σωματίδια, σημαίνουν και άλλες ρηπογόνες ουσίες και ούτω καθεξής. Εύα το είχαμε προσέξει περισσότερο αυτό. Συμφωνώ μαζί σας. Νομίζω ότι η ευρωπαϊκή πολιτική στόχευσε στην μείωση των διοξιδίων του άνθρακος και ίσως παραμέρισε κάπως τα οξύδια του αζότου. Και η αυτοκινητοβιομηχανία έπραξε το ίδιο. Όντως, όπως είπατε και εσεί, το ντίζελ είναι καλύτερο στο να εκπέμπει μειωμένα διοξίδια του άνθρακο. Με την ευρωπαϊκή πολιτική περιβάλλοντος, εν μέρη, ας βγάλουμε τα δημοσιονομικά κίνητρα, ε, φέρουμε ωστόσο πολιτικά ένα μέρος τη ευθύνη. Απάντηση δεν γνωρίζω αν θα πρέπει να μιλήσει κανείς για ένα μερίδιο συνευθύνης. Ωστόσο, θεωρώ ότι θα έπρεπε ευκρινέστερα από ό,τι το πράξαμε να είχαμε επισημάνει ότι η κινητικότητα με βάση το καύσιμο συνεπάγεται και συγκεκριμένα μειονεκτήματα και σημαντικά μειονεκτήματα. Αν διαβάσετε την ανακοίνωση ΚΑΡ 2020 θα δείτε πρόγραμμα δράσεων που αναφέρεται σε αυτές τις αρνητικές εκπομπές οξυδίων του αζότου και επισωματιδίων και λέει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν. Νομίζω δηλαδή ότι δεν ταχθήκαμε απαραίτητα υπέρ μιας τεχνολογίας ή κατά μιας άλλης. Αλλά όντως στα μάτια της κοινή γνώμης η αντίληψη που κρατεί και λόγω των φορολογικών ελαφρύνσεων που δώσαμε στις χώρες μέλη, προκλήθηκαν τελικώς, δόθηκαν τελικώς κίνητρα υπέρ της αγοράς αυτοκινήτων δίζελ. Ίσως τώρα, ε, ερώτηση καινούρια, βρισκόμαστε στη σημείο καμπής, όπου η κινητικότητα θα αλλάξει πάλι πρόσωπο. Προ δύο εβδομάδων είχαμε κοντά μας τον ε, Οραβείο Υπουργό και στην Ομοσπονδιακή Γερμανία έχει ανατεθεί μελέτη για να ε, μην χρησιμοποιούνται πλέον μηχανές καύσεως από το 2030 και μετά. Πράγματι στο σχέδιο, ανεξαρτήτως τώρα της εφικτότητας, δόθηκε η εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το μελετήσει. Θέλω λοιπόν τώρα να θέσω υπόψη σας κάτι που είπε ο Φρίτς Ίντρα, από την ε, καθηγητής από τη Βιέννη, που είπε ότι η, ο κινητήρας εσωτερικής καύσεως θα παραμείνει εκτός ανταγωνισμού για τα επόμενα 100 μέχρι 300 χρόνια. πιο 2030. Χρειάζεται λοιπόν προσπάθεια να βελτιωθεί και άλλο ο κινητήρας εσωτερικής καύσεως. Μιλούμε εδώ για κάποιον ο οποίος ε, βεβαίως είναι άνθρωπος ειδικό, δεν είναι ε, κάτι από το πρόγραμμα των πράσινων. Φάλκενμπερκ, κοιτάξτε δεν είμαι τεχνικός, είμαι οικονομολόγος. Γι' αυτό δεν θα αντίπω σε αυτά που λέει ο καθηγητής σας, αλλά νομίζω ότι και για τις ηλεκτρομηχανές, τους ηλεκτρικούς κινητήρες, δηλαδή θα πρέπει να σκεφτεί κανείς, μα από πού προέρχεται το ρεύμα το οποίο χρησιμοποιούν, πώς παράγεται αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα. Και από αυτή τη διαφορά θα φανεί τελικώς ποιο τρόπος είναι ο καλύτερος κίνησης δηλαδή των οχημάτων. Ε, ο κ. Ντάνς, ευχαριστώ ε, κύριε Φαλκενμπερκ. Πολύ σύντομα, μετά από αυτές τις ερωτήσεις που μόλις ακούσαμε, σας είπαν διάφοροι, ο ΙΕΜ, ε, περιβαλλοντικές ομάδες κλπ, ότι υπάρχει τεχνολογία για να μειωθούν και το διοξείδιο του άνθρακος και τα οξύδια του αζότου. Υπάρχουν τεχνολογίες αυτές. Πώς το βλέπετε? Απάντηση Φάλκενμπερκ. Ε, αυτό που κατανοώ εγώ είναι ότι όντως υπάρχει η τεχνολογία. Κατ' επανάληψη έχω ειδή... επιδείξεις από πλευράς επιχειρήσεων που μου δείχνουν ότι μπορούν να κατασκευάσουν ε, καθαρά αυτοκίνητα και στη μελέτη SCT δύο τουλάχιστον από τα αυτοκίνητα που εξετάστηκαν ανταποκρίνοντα τις προδιαγραφές αυτές. Λοιπόν, η δική μου αξιολόγηση είναι ότι όντως υπάρχει η τεχνολογία. Ευχαριστώ, λέει ο κ. Ντάνη. Ήθελα, βέβαια και ε, γνωρίζετε ότι η Επιτροπή μας, εξετάζει πού βρίσκονται τα νομικά παράθυρα, πόρτες κλπ. Και πού μπορεί να βελτιωθεί η υφιστάμενη νομοθεσία. Και πώς φτάσαμε εδώ που μπορει να βελτιωθει η υφισταμενη νομοθεσια και προστασαμε εδω που φτασαμε στην νομοθεσία. Δώσατε ένα καθαρόρισμο για το τι πιστεύετε ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό το cycle beating, η αντιστροφή του κύκλου. Η υπέρβαση του κύκλου, αν θέλετε. Φάλκενμπεκ, δεν έχω βρεθεί ποτέ σε εργαστήριο δοκιμών, αλλά οι ιστορίες που μου έχουν διηγηθεί κινούνται από ειδικά λάστιχα, τα οποία έχουν καλύτερη, ευκολότερη κύληση από τα λάστιχα που φορεί ένα αυτοκίνητο στην πραγματική ζωή, μέχρι μια προσπάθεια λεπτομερούς προγραμματισμού, ώστε οι διαδικασίες κινήσεως του αυτοκινήτου να είναι πέραν και από ιδέατες ή από ιδεώδεις. Αυτά τα παραδείγματα έχω ακούσει dance. Ίσως μερικοί από εμά να μπορούν όντω να οδηγούν έτσι, τι να πω. Με ενδιαφέρει ο ορισμός της διατάξεως αναστολής, του συστήματος αναστολής στην νομοθεσία. Κάθε, δηλαδή, το οποίο μπορεί να ανακόψει ή να τροποποιήσει ή να καθυστερήσει μέρος του συστήματος ελέγχου των καυσαέριων. Εάν τώρα αυτό το tuning, δηλαδή η ρύθμιση του κινητήρα, ε, οδηγεί σε, ε, σε υπέρβαση του κύκλου. Ε, Χωρί αυτό στον ορισμό σας. Δηλαδή δυσκολεύομαι να βρω διαφορά ανάμεσα στις δύο εκδοχές. Φάλκενμπεργκ. Νομίζω πολλοί θα δυσκολευτούν. Διάβασα και ξαναδιάβασα το νομοθέτημα πολλές φορές τα τελευταία ένα-δύο χρόνια και δεν νομίζω ότι μπορώ να σου προσφέρω ξεκάθαρες απαντήσεις. Ε, νομίζω ότι ο τρόπος που εξετάζει το θέμα και ο Γκερμπράντι προσπαθεί δηλαδή να καταλήξει στο αν υπάρχουν ενδεχομένω διαφορές ανάμεσα στην στάση μιας επιχείρησης απέναντι στον νόμο και στη στάση απέναντι στην ηθική. Σε αυτόν εξηγεί κάπως περισσότερο τις διαφορές. Από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, υπό την εποπτεία και την ευθύνη των εθνικών εργαστηρίων δοκιμών και των εθνικών αρχών που δίνουν, παρέχουν τις εγκρίσεις τύπων, θα γίνεται ο έλεγχος ότι γίνεται σεβαστή η νομιμότητα των δοκιμασιών, των τεστ. Δεν θεωρώ ότι μιλούμε για παράνομες δοκιμές και δεν το γνωρίζαμε μέχρι ότου που μάθαμε από τους Αμερικανούς ότι όντως υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Βουλευτής Ντάνης. έχει ζητηθεί, έχουν ζητηθεί τα στοιχεία αυτά από τις χώρες μέλη. Υποτίθεται λοιπόν όμως ότι τότε τα έχετε. Σας ρωτώ και για την απάντηση σας στην ερώτηση 4. Ε, λέτε ότι υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες καθυστέρησαν αδικαιολόγητα και ότι τέσσερις χώρες μέλη διαμαρτυρήθηκαν για τις καθυστερήσεις στην DCMV. Ποιες ήταν οι χώρες αυτές και ποιες είναι οι συγκεκριμένες ενστάσεις τους. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη ένσταση, απαντά ο κ. Φαρκενμπερκ, ήταν ότι τον Ιούνιο του 2014 ανεμένεται ότι στη συνάντηση του Οκτωβρίου θα κατετίθετο πρόταση για δοκιμές RBE και όταν εμφανίστηκε τελικώς η ατζέντα το θέμα δεν περιλαμβανόταν καν και οι τέσσερις χώρες μέλη αν θυμούμε καλά ήταν η Γερμανία, Ολλανδία, Δανία και μια τέταρτη που διαφεύγει. Μήπως το Ενωμένο Βασίλειο? Όχι, δεν νομίζω ήταν το Ενωμένο Βασίλειο. Καλή προσπάθεια πάντως, λέει ο Πρόεδρος. Και να ακολουθήσει ο κ. Φέντερ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας. Πρώτη ερώτηση. Όταν περνούσε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η νομοθεσία, υπήρχε η διάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανεξαρτήτως Γενικής Διευθύνσεως η θέση της Κομισιόν να είναι ότι θα πρέπει να περνά τις ε, δοκιμές εργαστηρίων που απαιτεί η νομοθεσία στον δρόμο. Αυτό έχει συστηθεί κατά επανάληψη. Διότι αυτά που βλέπουμε είναι ότι η βιομηχανία θεωρεί ότι οι δοκιμές γίνονται στο εργαστήριο. Ζητούμε καθίσματα ασφαλείας για τα παιδιά στα αυτοκίνητα, τα οποία να λειτουργούν σε ε, μια ενδεχόμενη σύγκρουση, αλλά θέλουμε να γίνονται και πραγματικές, ε, ε, να γίνονται και δοκιμές σε πραγματικές συγκρούσεις, σε πραγματικές συνθήκες. Γιατί αν αγοράσετε ένα λεξίπτο, θέλετε να ξέρετε ότι λειτουργεί και όχι μόνο στο εργαστήριο. Αυτά, αυτέ οι δοκιμέ λοιπόν θα λειτουργούσαν και στον δρόμο, Φάρκενμπεργκ. Αν καταλαβαίνω καλά την ερώτησή σα, αναφέρεστε σε ένα χρονικό σημείο που προηγείται της αφήξεώ μου στα θέματα ε, του περιβάλλοντος. Ρωτάτε δηλαδή όταν αυτή η εκτελεστική πράξη ε, βρισκόταν στη φάση της εξελίξεως, τι γινόταν. Δεν μπορώ να σας το πω. Αυτό που κατανοώ εγώ πάντως είναι ότι ο στόχος αυτή της ε, εκτελεστικής πράξης για την θέσπιση των απαιτήσεων για τις δοκιμές εργαστηριών ήταν να μπορέσει η βιομηχανία να αποδείξει ότι μια προδιαγραφή ευρώ 4, ευρώ 5, ότι σε αυτήν ανταποκρίνονται τα οχήματά τους, έτσι ώστε να τους χορηγηθεί έγκριση τύπου. Όμως δεν ήμουν εδώ τότε και δεν έχω γνώση για τις συζητήσεις που λάμβαναν χώρα τότε. και ο εισηγητής κ. Γκερμπράντι έχει επανέλθει στις εντάσεις μεταξύ DG Envy, DG Enterprise κλπ. Για την διαδικασία WLTP που είχε αρχίσει το 2008 και που εγκρίθηκε πρόσφατα. Αυτός, ας πούμε, ο αγώνας εξουσίας ανάμεσα στις διάφορες γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μήπως οδήγησε στην καθυστέρηση ολόκληρου του έργου, διότι προωθούσαν νομοθεσία αλλά τελικώς πέρασε πολλής χρόνος. Μήπως μπορεί αυτό να ε, είναι μία εξήγηση. Απάντηση Φάρκεντρικ. Δεν νομίζω ότι οι συζητήσεις μεταξύ γενικών διευθύνσεων απορροφούσαν την περισσότερη ενέργεια. Η, Γενική Διεύθυνση Enterprise τότε, το οποίο, το οποίο λέγεται Grow τώρα, ήταν η επί της ουσίας αρμόδια με συμμετοχή στις τεχνικές της Επιτροπές Εθνικών Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων. Αυτή η διαδικασία χρειάστηκε πολύ περισσότερο χρόνο και προσπάθεια από την διευκρίνηση των θέσεων των ιδιογενικών γενικών διευθύνσεων στις οποίες αναφερθήκατε εσείς. Υπήρξαν διαφορετικές απόψεις, υπήρξαν και διαφορετικά επίπεδα συνειδητοποιήσεως, υποθέτω, Γι' αυτό έκανα εγώ συζητήσεις ξανά και ξανά με τις αρμόδιε γενικές διευθύνσεις για να καταστήσω σαφές ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Προσπαθούσαμε να προχωρήσουμε στη διαδικασία αυτή μέσα ωστόσο στο χρονοδιάγραμμα του σχεδίου δράσεως και αυτά μας οδηγούσαν στον Σεπτέμβριο του 2014 μαζί με την εφαρμογή της πιο πρόσφατης προδιαγραφής της Ευρώ 6. Αυτά το 2012-2013 όπου είχε γίνει μεγάλη προσπάθεια για να γίνει συνείδηση η ανάγκη ε, επιτάχυνσης. Ερώτηση. Από τα τέλη δεκαετία του 90 και μέχρι τώρα όπου μάθαμε για, αυτές τις, για ε, αυτά τα συστήματα αναστολής. Έχουμε δει διάφορες εκθέσεις από μη κρατικούς οργανισμούς κλπ. Ότι υπάρχουν τεράστιες αποκλήσεις ανάμεσα στις μετρήσεις που γίνονται στα εργαστήρια και στον δρόμο. Δεν υπάρχει κάποιος αυτόματα λειτουργών μηχανισμός μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε όταν υποβάλλονται τέτοιες εκθέσεις να αρχίσουν να λειτουργούν, να αρχίσουν να δουλεύουν οι γενικές διευθύνσεις πάνω στον φάκελο αυτό ή απλώς συνεχίζεται η δουλειά ως συνήθως πάνω σε όλα αυτά τα θέματα. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, απάντηση τώρα, άρχισε μια μελέτη το με το JRC, με το Κοινό Κέντρο Ερευνών, ε, μετά από τα πρώτα δεδομένα που μας υποβλήθηκαν. Δηλαδή έγιναν δοκιμές με πραγματικές συνθήκες οδηγήσεως και αυτά τα αποτελέσματα των δοκιμών τα θέσαμε υπόψη και των άλλων συνεργαζόμενων γενικών διευθύνσεων. Τον Οκτώβριο 2014 έμαθα για τις δραματικά μεγαλύτερες αποκλίσεις σε σύγκριση με τη μελέτη του Γενικού Κοινού Κέντρου ε, Έρευνων από αυτά που είχε ε, σημειώσει η Γενική Διεύθυνση. Και αυτό έδωσε μια όθηση να πιέσουμε ακόμη περισσότερο. Όταν άρχισα να αντιλαμβάνομαι τις μεγάλες αυτές διαφορές, προχωρήσαμε σε διπλούς ελέγχους και σε μια προσπάθεια να ε, εξασφαλίσουμε ότι θα γίνονται δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες. Ευχαριστώ κύριε Λόπης Μπενέχο. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Φάλκεμπερ που είστε σήμερα εδώ κοντά μας. Από τις απαντήσεις σας στις γραπτές ερωτήσεις της Επιτροπής μας καταλαβαίνω ότι θεωρείτε πως η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος γνώριζε πριν από την άφηξή σας, στις αρχές δηλαδή του 2009, την ύπαρξη παρεκκλήσεων ανάμεσα στις εκπομπές σε εργαστήριο και τις πραγματικές εκπομπές των κινητήρων ε, diesel και εσείς ο ίδιος ενημερωθήκατε γι' αυτό το 2010. Επαληθεύθηκαν δύο φορές, ε, δύο ε, μάλλον στις μελέτη του ε, Κοινού Κέντρου Ερευνών το 2011 οι δε συσκευέ αυτές απαγορεύονταν για όλα τα αυτοκίνητα από το 1999. Αυτές επιβεβαιώνουν ένα μεγάλο κομμάτι της εργασίας αυτής εδώ της επιτροπή και είναι πολύ σοβαρέ παραλήψεις. Η υπηρεσία σα, επανειλημμένα ενημέρωσε τι αρμόδιε ε, αρχέ της Επιτροπής για αυτές τις σημαντικέ παρεκκλήσει και συγκεκριμένα τον κύριο Καγέχα. Γι' αυτό και θέλουμε να σα ρωτήσουμε και Έχω τα εξή τρία ερωτήματα να σας υποβάλω. Το πρώτο αφορά την νομιμότητα των ε, συσκευών αναστολής defeat device και Σύμφωνα με την ε, νομοθεσία του 1998 ε, απαγορεύονταν αυτοί οι συσκευές και αρκούσε αυτή η νομοθεσία για να απαγορεύονται και στις διαδοχικές μετέπειτα νομοθεσίες. Εσείς γνωρίζετε ότι υπήρχαν και χρησιμοποιούνταν αυτοί οι μηχανισμοί που παραβίαζαν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Πρέπει να σας επαναλάβω ότι δεν ήμουν υπεύθυνο για αυτήν την νομοθεσία, την παρακολούθησα. Δεν γνώριζα την χρήση συσκευών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παραβίαση των ορίων εκπομπών. Μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι σε καμία ε, περίπτωση δεν γνώριζα τέτοιες ε, πληροφορίες όπως αυτές που φαίνεται εσείς να λέτε. Ε, τώρα, σε ποιο βαθμό αυτές οι συσκευές είναι νόμιμες ή παράνομες, θα πρέπει να το δούμε και να οριστεί από τα δικαστήρια. Και είμαι βεβαίως ότι θα υπάρξει νομική δράση, θα ακολουθήσει νομική απόφαση ε, εγώ εργαζόμουν ε, υπό την υπόθεση ότι τα οι εργαστηριακές δοκιμές όπως είχαν σχεδιαστεί και όπως είχαν την νομικό εφαρμοστεί θα επέτρεπαν, θα, θα επέτρεπαν μεγάλες παρεκκλήσεις. Γι' αυτό και εγώ εστίασα στο ότι έπρεπε να κινηθούμε από αυτές τις δοκιμές τις εργαστηριακέ σε δοκιμές υπό πραγματικέ συνθήκες οδήγησης, διότι έτσι θα είχαμε μεγαλύτερο έλεγχο επί των πραγματικών εκπομπών των αυτοκινήτων. Δεύτερη μου ερώτηση με τις ε, νέες, ε, τα νέα όρια των 80 μιλιγκράμμα ανά χιλιόμετρο για τα οξύδια του αζότου που εγκρίθηκαν το 2007 δεν θα έχουμε φτάσει τα όρια αυτά ούτε το 2021. Εσείς όμως μιλήσατε για πιο φιλόδοξη πορεία. Πότε νομίζετε πως θα είναι δυνατόν να, τηρηθούν, να τηρηθούν τα στάνταρ του Ευρώ 6. Εγώ νόμιζα ότι θα ήταν τεχνικά δυνατόν τώρα. Είχα μια ερώτηση προς την ίδια κατεύθυνση. Υπάρχουν οχήματα που τηρούν αυτές τις εκπομπές ήδη. Εγώ δεν ορίζω να υπάρχουν, να είναι αδύνατο τεχνικά αυτό. Άλλη ερώτηση. Αλλά θα ήθελα να την αφήσω για το δεύτερο γύρο των ερωτήσεων, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Μάλιστα. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Η επόμενη μου είναι η κυρία Ντέλη. Ντάλη, μάλλον. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Γενική Διευθυντά, καλώς ήρθατε. Διάβασα προσεκτικά τις ερωτήσεις σας στο ρυθματολόγιο. Το μικρόφωνο της ομιλήτρης έχει κλείσει. Can you use your microphone, please? Thank you. ήρθατε λοιπόν στην ε, Επιτροπή Μα διάβασα με προσοχή τι απαντήσει σα, στι οποίε μα λέτε ότι δεν μπορούσατε ποτέ να διανοηθείτε ότι θα ε, κορόιδευαν οι ε, κατασκευαστές αυτοκινήτων και ακόμη περισσότερο με απατηλά συστήματα. Ταυτόχρονα μας λέτε στις απαντήσεις σας πάντα ότι από ορισμένε ε, πιστοποιημένες και από το Κοινό Κέντρο Ερευνών ε, μεθόδους ε, για την αναστολή, με συσκευέ αναστολής που μπορεί να μετριέται σε χαμηλή θερμοκρασία ή όταν έχει ανάγκη από πρόσθετη ισχύ το όχημα. Μάλιστα μας λέτε ότι ξεπερνούν οι πρακτικές αυτές ακόμα και τα επιτρεπόμενα από τη Euro 5 από την νομοθεσία αυτή. Εδώ θέλω να μου διευκρινίσετε σε τι αναφέρεστε κύριε Γενική Διευθυντά. Δεν είναι αυτά λογισμικά απατηλά. Και αν μου απαντήσετε αρνητικά, είναι όντως απολύτως παράνομο ένα απατηλό λογισμικό. Φάλκεμπεργκ. Στα γαλλικά από τα όσα άκουσα και κατάλαβα αυτά τα πέντε χρόνια που υπηρέτησα στη, από τη θέση αυτή είναι ότι αντελήφθην ότι υπάρχουν δυνατότητες μέσα από το κείμενο αυτής της νομοθεσίας για προστασία του κινητήρα και σε αυτό αναφέρεστε με την ε, παράθεση από τις απαντήσεις μου. Υπάρχει δηλαδή μια νόμιμη βάση από την νομοθεσία που επιτρέπει την εισαγωγή μηχανισμού ή ε, συσκευή που μπορεί να εξασφαλίσει τον έλεγχο των εκπομπών προκειμένου να προστατέψει την βιωσιμότητα, τον ίδιο τον κινητήρα ουσιαστικά. Τώρα, το μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό και από ποιο σημείο και μετά αναιρεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, είναι δύσκολο να το κρίνω από τις γνώσεις που έχω. Και δεν είδα ειδικό από αυτούς που συνάντησα τακτικά και συνομίλησα για τα θέματα αυτά, να ε, επισημαίνει ότι είναι εν γνώση απατηλών πρακτικών που ενδεχομένως να χρησιμοποιούνταν πέραν των όσων προβλεπόταν στην εφαρμοστική πράξη, δηλαδή πρακτικών που να ξεπερνούσαν τα όρια του νόμου και όσο και ήταν παράνομες. Κύριε Αντελή, θα επανέλθω και στο, ε, στην ερώτηση παριθμών 8 του ερωτηματολογίου, στην οποία δεν έχετε δώσει καμία απάντηση. Ερωτώ λοιπόν, ένα αυτοκίνητο, το οποίο ξεπερνά κατά πολύ τις οριακές τιμές, ενώ εντάσσεται στον κύκλο του νέου του συστήματος του νέου κύκλου, ευρωπαϊκού κύκλου οδήγηση, το NDED. E ερωτώ λοιπόν, NEDC συγγνώμη, ερωτώ λοιπόν, εάν αυτά τα αυτοκίνητα αυτά δεν ε, τηρούν τον νόμο, γιατί κυκλοφορούν στους δρόμους μας. Κύριος Φάλκενμπεργκ. Πολύ καλή ερώτηση νομίζω. Πρόκειται όμως για μια ερώτηση στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν κατά πρώτο λόγο οι αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την έγκριση και την θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων αυτών επί τη βάση των δοκιμών που έχουν διεξαχθεί. Πρώτες αυτές λοιπόν θα πρέπει να διασφαλίζουν την τήρηση από τα οχήματα αυτά της νομοθεσίας, το σεβασμό της νομοθεσίας και επίσης, αν υπήρξε κάποιο πρόβλημα ως προς την εφαρμογή θα πρέπει να αντλήσουν και τα σχετικά συμπεράσματα. Αυτό νομίζω ότι λέω και με την αρχική μου τοποθέτηση σήμερα, την αρχική μου ομιλία, ότι για μένα εγείρεται ένα πραγματικό νομικό ζήτημα άπαξ και η εφαρμοστική πράξη νομοθετήματος που έχει εγκριθεί επιτρέπει την υπέρβαση, τουλάχιστον κατά τα φαινόμενα επιτρέπει, την υπέρβαση κατά το 20 πλάσιο τιμής την οποία από κοινού το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν ή έχουμε αποφασίσει στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο τεχνικό το ζήτημα δηλαδή, είναι ουσιαστικό νομικό ζήτημα. Κύριε... Τέλειωσα κιόλας κύριε Πρόεδρε. Ναι, ε, εξέπνευσαν τα πέντε σας λεπτά. Κυρία Αίβη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ που είστε εδώ κύριε Φάλκεμπερ. Καλώς ήρθατε. Στην ε, ερώτηση παριθμών 3 κατηγορείται ουσιαστικά από ό,τι καταλαβαίνω τα κράτη-μέλη ότι δεν πραγματοποίησαν επαρκείς ελέγχους στην αγορά και θα αναφερθώ στο παράδειγμα της Σουηδίας, για την οποία διαβάζω ότι διερευνά περί τα ε, επενδύει κατά τα 2 εκατομμύρια ε, το χρόνο για, τις, ε, για τους ελέγχους των κινουμένων αυτοκινήτων. Και αυτό μάλιστα το είχε αποφασίσει πριν να ξεσπάσει το σκάνδαλο της Volkswagen που αποδεικνύει ότι οι εκπομπές ήταν πολύ ψηλότερες από τα όρια. Ε, πάντως βλέπουμε ότι οι διατάξεις προβλέπουν ότι μόνο η πιστοποιούσα αρχή μπορεί να παρέμβει, εάν είναι να παρέμβει κάποιος. Αλλά αυτό δεν συνέβη. Άρα βρισκόμαστε σε μια ε, ούτως υπήν αδράνεια από πλευρά των αρχών πιστοποίησης. Και βέβαια οι σχετικοί δεσμοί και με την αυτοκινητοβιομηχανία δεν επιτρέπουν από ό,τι φαίνεται στις αρχές να ε, παρέμβουν όπως τα όφυλαν. Ερωτώ λοιπόν. Υποβαθμίστηκε λοιπόν η σημασία αυτού του ζητήματος και της υποχρέωσης να αποσυρθούν τελικά αυτά τα ρηπογόνα οχήματα. Ερώτηση. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα αυτό, ένα ερώτημα, το οποίο θα ήταν καλό να συστήσετε με τον Ντανιέλ Καλέχα, ο οποίος έχει ε, ασχοληθεί με το θέμα της εποπτείας της αγοράς. Εγώ έχω μια εξωτερική μόνο εικόνα της κατάστασης και της νομοθεσίας από τη δική μου εμπειρία από την περιβαλλοντική νομοθεσία. Μπορώ να συμπεράνω ότι είναι σημαντικό για να υπάρχει σωστή επιτήρηση της, Ευρωπαϊκ... της εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, να ξέρουμε ξεκάθαρα ποιος έχει την ευθύνη για ποιο θέμα. Και αν αυτό περάσει μέσα από την αρχή της επικουρικότητας και περάσουμε στο στάδιο, στο επίπεδο των κρατών μελών, πρέπει να υπάρχουν σαφείς κανόνες που θα μας επιτρέπουν να βεβαιωνόμαστε κάθε φορά ότι τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν με ομοιόμορφο τρόπο την νομοθεσία και ότι ή μη τι άλλο θα υπάρχει ο έλεγχος το νομοτήμων όπως ονομάζεται το peer control για να βεβαιωνόμαστε ότι υπάρχει ο ουσιαστικός έλεγχος. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω με μια άλλη ερώτηση. Σε πολλές από τις μαρτυρίες που ακούσαμε σε αυτές τις ακροάσεις ε, μας υπόθηκε ότι είναι σχεδόν αδύνατον να εντοπιστεί η ύπαρξη ενός τέτοιου ε, συστήματος αναστολής και μάλιστα εν προκειμένου με το σκάνδαλο της Volkswagen δηλαδή η ίδια η Volkswagen ομολόγησε ότι είχε παρέμβει στις εκπομπές. Ωστόσο μας λέει ταυτόχρονα η Volkswagen ότι αυτό το λογισμικό της δεν παραβιάζει στην πραγματικότητα την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αντίθετα από ό,τι ισχύει στις ΗΠΑ. Πιστεύετε ότι είναι ορθή αυτή η ερμηνεία της νομοθεσίας από πλευράς της Volkswagen και πιστεύετε ότι δεν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να προβλεφθεί μια λύση που δεν θα επέτρεπε στη Volkswagen να ισχυρίζεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή να υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης μέσα από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ότι έχουν εισαχθεί συσκευέ αναστολής ή διατάξεις αναστολής, όπως ορίζεται από τον κανονισμό 715 με το άρθρο 3 για τα ελαφρά οχήματα εν αντιθέσει προς τα βαρέα. Απάντηση. Κοιτάξτε, η στρατηγική της Volkswagen, την οποία παρακολουθώ από τον τύπο, δεν είναι για μένα ε, προορισμένη στην επιτυχία. Γιατί υπάρχουν διαφορές στην νομοθεσία μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης ΜΕΝ και σωστά επισημαίνεται ότι υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης που προβλέπεται στην Αμερικανική νομοθεσία και αυτό άλλωστε ήταν και το κίνητρο για τη Volkswagen να ομολογήσει τις πρακτικές αυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά ο στόχος της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας είναι ο ίδιος ακριβώς. Και άρα η απαγόρευση της εισαγωγής συσκευών αναστολής και για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι σαφώς διατυπωμένη. Δεν βλέπω δηλαδή πώς μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι το να σβήνουν αυτές οι συσκευέ ε, υπό τις κανονικές συνθήκες οδήγησης μπορεί να στηριχθεί σε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι μεταξύ έχει έρθει ο δεύτερο ηγητή μα, ο κύριο Άλμπα. Αλλά για να ολοκληρώσουμε αυτό το γύρο, και για να ολοκληρώσουμε αυτόν τον γύρο, θα ήθελα να του δώσω το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά ε, δυστυχώ ε, υπήρξε καθυστέρηση στο πτήση μου, αν και παρακολουθούσα μέσω streaming τις παρεμβάσει του κυρίου Φάλκεμπεργκ. Έχω διάφορε ερωτήσει. Ε, θα ήθελα καταρχά να γνωρίζω μετά από την ανταλλαγή επιστολών με τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποια ήταν η δική σα αντίδραση στην απάντηση του Γενικού Διευθυντή. Φάλκενμπεργκ. Εγώ συνέχισα να συζητώ με τον Ντανιέλ Καλέχα, αλλά στην απάντησή του βασικά συμφώνησε μαζί μου ότι ήταν επίγον το θέμα και εξήγησε, μου εξήγησε γιατί συνέβησαν κάποιες καθυστερήσεις. Ε, τόνισε ότι χρειάζεται να υπάρχει ε, ε, δυνατότητα πλειοψηφία στην Τεχνική Επιτροπή πριν την υποβολή πραγματική πρόταση. Δηλαδή πριν να τεθεί επιτάπητο και πριν να ψηφιστεί. Εγώ συνεχίζω λοιπόν τη συνεργασία μου μαζί του, ώστε να προσπαθήσω να τον πείσω ότι τα κείμενα επί των οποίων έχουμε εργαστεί ήταν αρκετά όρημα ώστε να τεθούν ε, επιτάπητο και να πιέσουμε για ψήφο. Ωραία. Επίση, είχα συζήτηση με του εκπροσώπου τη αυτοκινητοβιομηχανία για να προσπαθήσουμε, να προσπαθήσω μάλλον να του καταστήσω απόλυτα σαφέ ότι οποιαδήποτε κολυσιεργία, οποιοδήποτε περαιτέρω πρόβλημα προκύψει σε αυτή τη διαδικασία, ώστε να υπάρξει καθυστέρηση, τελικά εκείνου θα επιβαρύνει και θα ε, δημιουργηθεί έτσι ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Προσωπικά λοιπόν, ε, νεπλάκιν ε, ε, πλήρως και με την ομάδα μου προσπαθήσαμε έτσι ώστε να μπορέσει να ψηφιστεί γρήγορα μια πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Είναι αλήθεια ότι συμφωνήσατε με το τελικό αποτέλεσμα που κατάφεραν να, έχουν μερικούς μήνες αργότερα. Μάλιστα. Εν τέλει, συνεχάρει το συνάδελφο για το γεγονός ότι αν και ε, εκτός προθεσμίας είχαμε τελικά ε, στήριξη της πρότασης που υπευλήθη. Χαίρομαι για αυτή τη συνεργασία και για το ότι είχε καρπούς και ότι συμφωνούσατε μεταξύ σας. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία επιτρέπει την έναρξη άμεσων ε, ερευνών για τους ε, στις διάφορες αυτοκινητοβιομηχανίες. ισχύουσα ο... Ναι. Και πάλι νομίζω πως η ερώτηση θα είναι καλύτερο να τεθεί στην ε, Γενική Διεύθυνση που είναι αρμόδια για αυτήν την νομοθεσία για την νομοθεσία για την οποία εγώ είμαι αρμόδιο στον τομέα του περιβάλλοντος. Μπορώ να σα δώσω παραδείγματα όπου υπάρχουν ρητοί τρόποι που προβλέπονται για την παρακολούθηση της εφαρμογής, αλλά υπάρχουν και νομοθεσίε όπου αυτό δεν προβλέπονται και όπου η εφαρμογή, η επιβολή της νομοθεσίας ε, ανατίθεται στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν και δύο περιπτώσει. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να ξεκινήσει κανεί άμεσα έρευνα αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ να το συζητήσετε με τους συναδέλφους που έχουν και ασχολούνται με αυτήν ακριβώς την νομοθεσία. Ναι, αλλά και εσείς θα πρέπει να γνωρίζετε αν είναι δυνατόν ή όχι να ξεκινήσει κανείς άμεσα έρευνα. Κατά τη γνώμη σας είναι δυνατόν ή όχι. να σας πω, είμαστε διαφορετικές γενικές διευθύνσεις και εγώ ως γενικός θητής δεν γνωρίζω απ' έξω κάθε νομοθέτημα που ε, ε, προτείνει και εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε να μπείτε σε λεπτομέρειες για κάθε νομοθέτημα και να δείτε ακριβώς με ποιο τρόπο ερμηνεύεται, νομίζω πως είναι πιο λογικό να θέσετε τα ερωτήματα αυτά σε αυτούς που είναι αρμόδιοι για αυτή την νομοθεσία. Εγώ το έχω συζητήσει μαζί τους, από ό,τι κατάλαβα θεωρούν ότι είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες, αλλά αυτή δεν είναι δική μου κρίση, είναι από αυτά που έχω ακούσει. Εγώ από αυτά που κατάλαβα δεν προβλέπονται η διενέργεια άμεσων ερευνών. Δεν λέω αν είναι καλό ή κακό, αλλά εν πάση περιπτώσει με εντυπωσιάζει που εσείς δεν το ξέρετε αυτό. Εγώ αυτό που προσπαθούσα να κάνω με αυτήν την επιστολή ήταν να τονίσω πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και ότι πρόκειται για πρόβλημα που επηρεάζει ένα τομέα πολιτικής για τον οποίο εγώ είμαι αρμόδιος, δηλαδή η ε, ρήπανση του ατμοσφαιρικού αέρα σε ολόκληρη την Ένωση, κυρίως λόγω του τομέα των μεταφορών. Και γι' αυτό έλεγα στον συνάδελφο παρακαλώ να εξασφαλίσετε ότι οποιαδήποτε δυνατότητα που εσύ, ε, για την οποία εσύ υπεύθυνο νομοθετικά να τη διερευνήσει. έτσι, ε, και χρηματοδοτήσαμε τη μελέτη του Κοινού Κέντρου Έρευνων για να δούμε ε, σε τι οφείλονταν αυτές οι διαφορές, οι αποκλήσεις. Ε, υπάρχουν τρόποι δηλαδή με τους οποίους μπορεί κανείς να ψάξει περισσότερο ε, και αυτό προσπαθούσα να διαβιβάσω σε αυτή μου την επιστολή προς τον συνάδελφο. Μάλιστα. Έτσι ολοκληρώνει το πρώτο γύρο των ερωτήσεων και περνάμε στο δεύτερο γύρο των ερωτήσεων, όπου ο κάθε ερωτών έχει τρία λεπτά για την ερώτηση και την απάντηση. Παρακαλώ λοιπόν να κρατάτε το χρόνο σας, ώστε να υπάρχει χώρος για απάντηση. Πρώτος τώρα λοιπόν, ο μιλητής είναι ο κύριος Γκίζικε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Φάλκενμπερκ, θα επανέλθω στην προηγούμενη μου ερώτηση για το μέλλον του ε, κινητήρια εσωτερικής καύσης. Ε, μπορεί να υπάρχει ένα πράσινο μέλλον στους δρόμους όταν ε, δηλαδή δεν θα υπάρχουν ούτε διοξίδια του άνθρακα ούτε οξίδια του αζότου αρκεί αυτή, αυτό το όραμα η παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπορεί, με όσα μας λέει το το Φράουενχοφ, να έχει επιβάρηση για το περιβάλλον κατά 80% μεγαλύτερη από το κινητήριο στερικής καύσης και λόγω της παραγωγής ε, της ε, ε, μπαταρίας και του αναγκαίου ρεύματος. Έτσι λοιπόν μπορείτε να μας πείτε τι είδους αηφόρο παραγωγή ε, ρεύματος μπορείτε να προβλέψετε ε, πυρηνική ενέργεια, ε, ορυκτά καύσιμα, υδρορογμάτωση, αιωλική ενέργεια κτλ. Απάντηση. Ναι, πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε ολιστικές προσεγγίσεις. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια, έναν απλό διαχωρισμό μεταξύ των ηλεκτρικών κινητήρων και των κινητήρων εσωτερικής κάψεις, ε, δηλαδή ότι ο κινητήρας ο οποίος ε, τροφοδοτείται από μια μπρίζα είναι καθαρός, γιατί πρέπει να δούμε αυτή η πρίζα που, από πού παίρνει το ρεύμα της, με ποιο τρόπο εξασφαλίζει το ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι λοιπόν, στο μείγμα πόσο άνθρακα, πόσο πετρέλαιο και ό,τι άλλο χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε μια δημόρφωση μείγματος καταλληλότερο, θα έχουμε καλύτερο περιβάλλον, καθαρότερο περιβάλλον και εν τέλει τη μικρότερη επιβάρυνση για το περιβάλλον. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πως πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο προς τις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργεια για να έχουμε καθαρότερο περιβάλλον. Καλώς ε, επανέρχομαι λοιπόν. Είπατε νωρίτερα, έχετε μάλλον πει στο παρελθόν ότι δεν, υπήξατε, δεν, δεν μπήκατε ποτέ σε εργαστήριο δοκιμών. Δεν υπάρχει στο κοινό κέντρο ερευνών εργαστήριο δοκιμών. Έχετε πάει εκεί, το έχετε παρακολουθήσει όταν ήσασταν γενικός διευθυντής. Ποτέ δεν πήγατε στην Ίσπρα. Απάντηση. Να διορθώσω τα λόγια μου. Όχι, έχω επισκεφθεί την Ίσπρα. Έχω μπει στο εργαστήριο της Ίσπρα, το έχω επισκεφθεί. Αυτό που είχα πει ήταν ότι δεν έχω μπει, δεν έχω επισκεφθεί κανένα εργαστήριο δοκιμών κράτους μέλους. Στην Ίσπρα βεβαίως και έχω μπει και μάλιστα στο εργαστήριο ελέγχου εκπομπών. Ο πρόεδρος ευχαριστώ. Bon θα μιλήσω γαλλικά. Και ξεκινώ από τα ε, εισαγωγικά σας λόγια. Είπατε ότι θα θέλατε μια πιο σαφή και ακριβή αυστηρή νομοθεσία, ανεξάρτητους ελέγχους, πολύ ωραία και εμείς ε, στα όσα ζητούμε διαρκώς ε, απαιτούμε μια ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Αρχή Ελέγχου και επιβολής κυρώσεων των παραβιάζει την νομοθεσία και συντονισμένε και γρήγορες δράσεις. Πολύ ωραία όλα αυτά τα οποία μας προτείνεται ως συμπεράσματα. Θα επανέλθω όμως στον απολογισμό της θητείας σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την ανταλλαγή επιστολών που είχαμε την ευκαιρία να μελετήσουμε μεταξύ ημών και των συναδέλφων σας και στα όσα μας είπατε και στην απάντηση στην αδελφή κυρία Αντελή, μας είπατε ότι και στο, στο παρελθόν ήταν ο σεβασμός, ο περιορισμός των εκπομπών οξυδίων του αζώτου μέλημα. Γιατί λοιπόν εσείς την εποχή που ήσασταν Γενικό Διευθυντή. Και μιλώ για τη συγκεκριμένη αυτή περίοδο. Δεν κάνατε κάτι, δεν, ε, δεν εισαγαγάτε ένα σύστημα κυρώσεων ή δεν κάνατε κάτι περισσότερο για να ζητήσετε από τα κράτη-μέλη να ε, περιορίσουν ή να ελέγξουν καλύτερα τι εκπομπέ οξυδίων του αζότου. Απολογισμό λοιπόν είναι αυτό που σα ζητάω. Σήμερα, 2016, κάνοντα την αναδρομή στα όσα ε, πράξατε στο παρελθόν, τι συμπεράσματα μπορείτε να βγάλετε, ελπίζοντα βέβαια ότι θα μου δώσετε μια απάντηση σαφή και ειλικρινή. Απάντηση. Αναλύοντας την κατάσταση, διεπίστωνα ότι η εφαρμοστική νομοθεσία δεν ήταν επαρκώς ακριβής και ότι δοκιμές σε ε, εργαστήριο που είχαν προκύψει κατόπιν διαπραγματεύσεων ατέρμονων επί χρόνια με πολύ υψηλό βαθμό τεχνικής λεπτομέρειας, πάλι δεν επέτρεπαν την ε, ε, ασφάλεια ότι θα μπορούσαν να γίνονται οι μετρήσεις σε πραγματικό περιβάλλον των εκπομπών. Επομένως, δική μου πρόθεση ήταν η βελτίωση της νομοθεσίας, η τροποποίηση της νομοθεσίας, η βελτίωση της νομοθεσίας, ώστε να μπορούμε ναι, με συγχωρείτε όμω η βελτίωση τη νομοθεσία αφορά το μέλλον, αλλά στο παρόν υπάρχει η τήρηση τη υφισταμένη νομοθεσία και πολλοί από αυτού του οποίου είδαμε με τι ακροασει μα έλεγαν ότι είναι αρκετά συγκεκριμένη, ακριβή αυτή η νομοθεσία. Γιατί λοιπόν δεν έγινε αυτή η δουλειά, όταν η Επιτροπή το κάνει για τόσα άλλα κείμενα, γιατί για τον κανονισμό 715 του 2007 δεν έγινε η σχετική δουλειά, δηλαδή η εξασφάλιση ότι τηρείται αυτή η νομοθεσία, δεδομένου ότι είχατε στοιχεία και ήδη από το 2009-2010 υπήρχαν κάποιες ανταλλαγές ε, ηλεκτρονικού τουλάχιστον ε, ταχυδρομείου που δείχνουν ότι υπήρχαν υπόνοιες για ε, διατάξεις αναστολής. Απάντηση. Τα στοιχεία τα δικά μας, αυτά που είδα εγώ τουλάχιστον, δεν με οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι υπήρχε στοιχειοθετημένη επαρκώς απόδειξη για παράβαση νομοθεσία. Δηλαδή οι υποθέσεις με τις οποίες εργαζόμασταν μπορούσαν να καλυφθούν από την εξήγηση των δύο πρώτων σημείων προσπάθησα να σας παρουσιάσω, δηλαδή την διαμόρφωση σε ένα εργαστήριο του τρόπου οδήγησης ενός αυτοκινήτου κατά τρόπον ώστε τελικά να εξηγείται η διαφορά εκπομπών μεταξύ διαφόρων οχημάτων. Ε, και από αυτά που είδα εγώ, δεν κατέληξε σε ένα συμπέρασμα σαν αυτό που πονοείται. Μέχρι ότου η μελέτη ICCT μας μίλησε για αποκλήσεις 20 πλάσες μέχρι και 37 φορές περισσότερες εκπομπές φάνηκαν σε ένα συγκεκριμένο όχημα από τις ε, προβλεπόμενες και ακριβώς τότε άρχισα να γύρω εγώ και ερωτήματα και προς τον συνάδελφο Καλέχα ε, για το εάν υπάρχουν νομικά ζητήματα, αν υπάρχει δηλαδή βάση για μια ε, ένομη δράση. Αυτά τα είδα εγώ στο τέλος του 2014, ουσιαστικά τη στιγμή που ερχόταν η ώρα της αντικατάστασης της παλιάς αυτής νομοθεσίας από μια νέα νομοθεσία που μιλούσε πλέον για πραγματικές εκπομπές. Ε, ε, έθεσα λοιπόν το θέμα αυτό στον συνάδελφο που ήταν και υπεύθυνο και συνέχισα εγώ να πιέζω για μια πιο συγκεκριμένη νομοθεσία, πιο κατάλληλη νομοθεσία έτσι ώστε να μετράτε ε, ακριβώς τι εκπέμπουν τα αυτοκίνητα σε πραγματικό περιβάλλον, σε πραγματικές συνθήκες. Αντί να μιλάμε για το αν υπάρχει ε, χειραγώγηση, αναστολή, νόμιμη ή μη. Ούτως ή άλλως επρόκειτο να αντικατασταθεί, δηλαδή όπως θέλαμε όλοι. Άλλωστε η νομοθεσία. Ευχαριστώ κύριο Γκίζικη. Πάλι εγώ κύριε Φάλκενμπεργκ στην εισαγωγική σας ομιλία. Ζητήσατε ευκρίνεια της νομοθεσίας και ομοιόμορφη εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Ξέρετε πολύ καλά βεβαίως ότι δεν μπορεί πάντοτε η πραγματική ζωή να ακολουθεί τη θεωρία. Στην πράξη υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες από τα διαφορετικά κράτη-μέλη. Και το έχουμε δει εμείς ε, εδώ στην Επιτροπή μας από τον Υπουργό των Μεταφορών της Γερμανίας, ε, ο οποίος μάλιστα είχε κάνει μια ένα διάβημα προς τη Βιφίατ προκειμένου να δει εάν ήταν νόμιμο ή μη ένα σύστημα αναστολής. Ενώ στην Ιταλία η ερμηνεία που δινόταν ήταν διαφορετική. Ε, μετά έγινε λόγος για, μια, για ένα clearing, ε, για μια θέση clearing, για μια μονάδα clearing, δηλαδή εξίσωση των θέσεων και ρωτώ εάν αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει λύση και μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί πάντα θα υπάρχουν αποκλήσει και ερμηνείε διαφορετικέ από την κάθε Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα υπάρχει λοιπόν κάπου ένα συντονισμό ώστε να ε, εφαρμόζεται ομοιόμορφα και στην πράξη νομοθεσία. Απάντηση. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό μαζί σα, γιατί πιστεύω ότι η ενιαία υλοποίηση, εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία μπορεί να βελτιωθεί εάν ε, προβλεφθούν περισσότερες δυνατότητες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μια υπηρεσία ενδεχομένως, ανεξάρτητη υπηρεσία, η οποία θα είχε ως έργο να παρακολουθεί τον τρόπο με την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές ε, του δικαίου στα επιμέρους Ανέφερα και νωρίτερα ότι αντιμετωπίσαμε πολλές φορές διαφορές ερμηνείας οι οποίες ε, προκειμένου να διευκρινιστούν έπρεπε να φτάσουν μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ωστόσο, πιστεύω ότι τουλάχιστον ο έλεγχος ε, των ομοτήμων, το peer control, ε, μπορεί να είναι αξιόπιστη μέθοδος. Και έτσι μπορούν οι εθνικές αρχές να συντονιστούν κατά τρόπον ώστε να ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο, με ομοιόμορφο τρόπο την ε, νομοθεσία. Γκίζικε. Ναι. Επιτροπή. Υπηρεσία. Πλατφόρμα. κεντρικά οργανωμένη δηλαδή αρμοδιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτό που μας λέτε. Και αν υπήρχαν όλα αυτά θα είχαμε αποφύγει το σκάνδαλο Volkswagen. Οι υποθετικές ερωτήσεις ε, δύσκολα βρίσκουν απάντηση. Από ό,τι βλέπω εγώ, και από τα παραδείγματα που έχω υπόψη, όπου είχε δυνατότητες για ελέγχους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Φερρυπίνη στον χώρο των φαρμάκων, όπου έχουμε σαφείς μηχανισμούς εποπτείας στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βλέπω ότι τα συστήματα φέρνουν αποτελέσματα και καλύτερα αποτελέσματα από ότι μια χαλαρή ε, σχέση. Ευχαριστώ κυρία Ανταλή. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Φάλκεμπερκ που είστε εδώ. Ε, θα ανατρέξω στην επιστολή σας προς τον κύριο Καγιέχας όπου λέτε ότι υπάρχει περιθώριο για τροποποιήσεις ε, που θα επιτρέψουν ε, δράση εις βάρος των ξεκάθαρα παράνομων πράξεων. Υποθέτω ότι ε, υπονοούσατε έτσι από αυτό που διαβάζω ότι η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων, η Enterprise, ήταν δεκτική σε τροποποίησεις από την αυτοκινητοβιομηχανία, τροπολογίες μάλλον από την αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτό εννοούσατε και σε ποιο βαθμό υπήρχαν τέτοιου είδους πρακτικές. Απάντηση. Η παράθεση αφορά και σωστά συζητήσεις εντός και περί την TCMV. Εκεί δηλαδή όπου είχα την εντύπωση ότι οι εκπρόσωποι της αυτοκινητοβιομηχανίας προσπαθούσαν ξεκάθαρα να υποβαθμίσουν ε, την νομοθεσία, να υπονομεύσουν την ε, νομοθεσία για τους ε, μηχανισμούς ελέγχου εκπομπών. Και μάλιστα σε μία περίσταση, σε μία τεχνική ομάδα, είχαμε την εντύπωση ότι οι συνάδελφοι έτειναν πιο ευήκον ους στα επιχειρήματα της αυτοκινητοβιομηχανίας από ό,τι θα είχαμε εμείς τίνει. Και μάλιστα είχα επισημάνει στον συνάδελφο συγκεκριμένο ότι πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερως για να έχουμε μια σωστή και ξεκάθαρη νομοθεσία απάντηση. Δηλαδή μας λέτε ότι αυτή τη διαδικασία την επηρέασε σε, περισσότερο από, μεγαλύτερο από το δέοντα βαθμό η αυτοκινητοβιομηχανία. Δεν ξέρω αν είναι περισσότερο από το δέον ή υπερβολικά. Πάντως η αυτοκινητοβιομηχανία προσπαθούσε να εισαγάγει ορολογία ε, τυπώσεις οι οποίες θα αποδυνάμωναν την νομοθεσία. Και εγώ δεν έχω αντίρρηση ω προς το ότι υπάρχει βέβαια και ανάγκη για την πραγματογνωμοσύνη των ε, ε, του φορέα. Αλλά υπήρξε, όπως σας είπα, περίπτωση όπου θεώρησα ότι δεν ήταν χρήσιμες οι υποδείξεις και ότι θα έπρεπε να αντισταθούμε σε αυτές. Μάλιστα. Από εκείνο το σημείο και για να γυρίσουμε στα όσα έχουμε εντωμεταξύ δει, Και αφού μας λέτε ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε πολλές ομάδες εμπειρογνωμόνων ε, συμμετέχει η αυτοκινητοβιομηχανία και δίνει και την πραγματογνωμοσύνη κτλ. Βλέπετε κάποιες αντιφάσεις, ε, μπορεί να επηρεάσει ενδεχομένω την διατυπούμενη νομοθεσία. Απάντηση. Κοιτάξτε, στο βαθμό που λαμβάνεται υπόψη, οι, ε, λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές τους γνώσεις και αυτές αντισταθμίζονται από τη δική μας αξιολόγηση, την ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη, τεχνική πραγματογνωμοσύνη των ε, ερευνητικών Ινστιτούτων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων ή άλλων φορέων. Δεν έχω πρόβλημα σε αυτό, δεν έχω αντίρρηση, γιατί έτσι έχουμε μια ευρύτερη βάση πάνω στην οποία θα στηρίξουμε ε, επιστημονικά βάσιμες αποφάσεις. τελευταία ερώτηση. Την ισορροπία αυτή βλέπετε να την επιτυγχάνουν αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το αποτέλεσμα και η νομοθεσία RD που έχουμε τώρα για το νέο σύστημα είναι νομίζω ισορροπημένη, ναι. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Α, ο κύριος Γκίζικε. Φαίνεται πως ε, συμμετέχω σε σειρά. Καλά τα πήγατε κύριε Φάλκενμπερκ. Έχω ωστόσο τώρα λίγο πιο κριτικές ερωτήσεις. Αυτή η περίφημη επιστολή του 2014. Εξ όσων γνωρίζω, η επιστολή αυτή προς την Γενική Διεύθυνση Enterprise περίχει και ένα παράρτημα. Αυτά τα γνωρίζουμε από την ταχεία επικοινωνία με ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, αν δηλαδή δεν λάβω ένα ε, παράδειγμα, ένα συνημένο θέλω να πω, τότε αμέσως με ειδοποιεί το σύστημα. Φαίνεται τώρα πως την ε, Κομισιόν, και βεβαίως μιλούμε πάντοτε για καλύτερη νομοθεσία, χρειάστηκαν λοιπόν δέκα μήνες. Είτε εσείς στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος γράψατε ένα email χωρίς το συνημένο ή στην ε, GD Enterprise είδαν ότι έλειπε ένα συνημένο Πώς, εν πάση περιπτώσει, επί ένα δεκάμινο ε, δεν έγινε αντιληπτό ότι παρόλο που αναφερόταν ε, συνημένο, τελικώς δεν είχε ληφθεί το συνημένο. Απάντηση Φάλκενμπερκ. Νομίζω ότι η μοναδική εξήγηση είναι ότι θεωρούμε ότι τα πράγματα έγιναν όπως είχαμε φανταστεί. Και στις συζητήσεις που έκανα μετά με τον συνάδελφο Καλέχα, ε, συζητήσαμε για αυτά τα πράγματα. Εξ αρχής δηλαδή δεν είχα ειδοποίηση ότι αυτά που είχαν εξέλθει τελικώς, δηλαδή το, τα εξερχόμενο mail δεν είχε το συνημένο αυτό, διότι μιλήσαμε και για το συνημένο. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα feedback, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Δηλαδή, σε έλεγχο εκ των υστέρων έγινε αντιληπτό ότι είχε ανακοινωθεί ότι θα έρχεται και συνημένο, τελικό όμως το συνημένο δεν είχε φτάσει. Άρα μιλήσατε για ένα συνημένο το οποίο δεν είχε αποσταλεί καν. 9 Ενδεκάτου 2014. Και μετά από την δημοσιοποίηση του σκανδάλου Volkswagen, τότε δημοσιεύσατε το συνημένο ή το ανακαλύψατε. Είναι παράξενο αυτό. Ελπίζω πάντως στις τωρινές εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην χρειάζεται ένα δεκάμινο για να στείλει ένα συνημένο. Συμφωνώ μαζί σας, ε, λέει ο ε, Γενικός Διευθυντής Φάρκενμπερκ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπλάνκο Λόπεθ. Ευχαριστώ. Όλα αυτά που ακούμε εδώ και εσείς συμμετείχατε στην ε, συνεδριάση της τεχνικής ε, ομάδας για το ε, RDE. Εσείς θέσατε αυτές τις ανησυχίες σας υπόψη των κρατών μελών. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν συμμετείχα σε DCMV, την ε, Τεχνική Επιτροπή για τα ε, οχήματα με κινητήρε, αλλά οι εκπρόσωποι της ε, Γενικής μου Διεύθυνσης συμμετείχαν και έθεσαν τις ανησυχίες μας. Ο μιλητής χωρίς μικρόφωνο. Δεν είναι αναμένο. Ναι, με συγχωρείτε. Έθεσαν λοιπόν τις ανησυχίες προς τα κρατημέλη. Ποιες ήταν οι απαντήσεις τους, εφόσον έθεσαν αυτές οι ερωτήσεις. Υπήρξαν πολλές αντιδράσεις, τόσο εντός της Επιτροπής, και αυτά όλα θα έχουν καταγραφεί στα πρακτικά. Υπήρξαν διμερείς συζητήσει που ξέρω τι έγιναν γιατί οι συνάδελφοι μου διαβίβασαν τα όσα διαμήθησαν εκεί στη διάρκεια όλων αυτών των ετών. Υπήρξε ανταλλαγή ε, γραπτών γράφων, τηλεφωνήματα, συζητήσεις για τα θέματα εντός και εκτός αυτών των συνεδριάσεων. Οπότε ναι, υπάρχει τακτική ανταλλαγή απόψεων. Υπήρχε μάλλον τακτική ανταλλαγή απόψεων. Εσείς είπατε ότι Υπήρχε μια ε, εντατική συνεργασία με τον κύριο Καγέχα στη διάρκεια όλη αυτή τη διαδικασία. Υπήρχε επικοινωνία ανάμεσα στι γενικέ διευθύνσει. Όμω, σε ποιο βαθμό υπήρχε αποτελεσματική συνεργασία ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που εσεί ανακαλύπτατε στην πορεία. Again, uh, we, we did it on, on several... Και πάλι, επανειλημμένα, ε, βλεπόμαστε, είμαστε συνάδελφοι, επαν, ε, έχουμε επαφές. Το ξεκινήσαμε με τον κύριο Σούρικ, αλλά όταν ήρθε και ανέλαβε ο Ντανιέλ Καλέχα αυτή την ε, θέση, Είχαμε τακτικές ε, συνεδριάσεις των γενικών μας διευθύνσεων μεταξύ μας και εκεί ο καθένας μας έβαζε τα θέματα που θεωρούσαμε ότι ήταν απαραίτητο να συζητηθούν. Και επανελειμμένα Μιλήσαμε για την ανάγκη να προχωρήσουμε από τα εργαστηριακά τεστ στις, δοκιμές, στις δοκιμές πραγματικής οδήγησης. Και ο Ντανιέλ και εγώ δεν είχαμε ποτέ αποκλίνουσες απόψεις ότι όντως αυτή ήταν η κατεύθυνση που έπρεπε να ακολουθήσουμε και ότι έπρεπε αυτό να γίνει επιγόντως ώστε να ενταχθεί στην, στο πρόγραμμα δράσης CAR 2020. Τελευταία ερώτηση το περιθώριο των ανακοινώσεων που εσείς είπατε ότι ότι δεν υπήρχαν διαφορές στη στιγμή που έπρεπε να δοθούν απαντήσεις από πλευρά των γενικών διευθύνσεων, ότι είχα την ίδια άποψη. Αυτό μας επιβεβαιώσατε, έτσι. Κοιτάξτε, οποτεδήποτε είχα συζητήσεις με, με τον συνάδελφο, συμφωνούσαμε ότι έπρεπε να προχωρήσουμε αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιες φορές δεν ήταν πιο αργή η διαδικασία πόσο θα το επιθυμούσα εγώ, αλλά και εκείνος θα ήθελε να έχει προχωρήσει γρηγορότερα η διαδικασία. Ωστόσο δεν καταφέραμε γρηγορότερα ε, να τα ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ. Κυρία Ιτικ, τα επόμενα τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Φάλκενμπεργκ. Θεωρείτε ότι αυτή η υπέρβαση του κύκλου μπορεί να οριστεί με τρόπο ακριβή και αν ναι, θεωρείτε ότι τέτοιες πρακτικές είναι εκτός νόμου ή βρίσκονται σε μια θεά ζώνη. Και ποιος θεωρείτε ότι θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνο να εξετάσει την θεά αυτή ζώνη και γιατί δεν ανελήφθη άμεσα δράση. Φάλκενμπρικ. Επανέρχομαι στην αναλογία που χρησιμοποίησα, χρησιμοποίησα προηγουμένως. Είναι δύσκολο να πει κανείς πότε η φοροαποφυγή είναι νόμιμη μεν, ανήθικη δε. Και νομίζω η αναλογία αυτή ταιριάζει και στην κατάσταση που συζητούμε. Έχουμε δει κατασκευαστές που προσπάθησαν να βελτιστοποιήσουν τα οχήματά τους σε δοκιμές εργαστηρίων ώστε αυτά να αποδίδουν τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το έπραξαν εντός των ορίων της νομοθεσίας ή τουλάχιστον αυτό νόμιζα. Μετά κατανοήσαμε ότι τουλάχιστον σε μια θεμελιωμένη, αποδειγμένα δηλαδή περίπτωση της Volkswagen, ότι είχαν υπερβεί τα όρια. Εγώ θεωρούσα πάντως αρχικά ότι βρίσκονταν μέσα στα όρια και γι' αυτό η αντίδρασή μας ήταν α βελτιωθεί η νομοθεσία. Βελτίωση τη νομοθεσία θα σήμαινε να φύγουμε πλέον από τα εργαστήρια και να γίνουν οι μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες, καθώς το αυτοκίνητο θα κινείται μέσα σε πόλεις ε, ή στην Ήπεθρο ή ανεβαίνοντας ε, στο βουνό και Άρα ε, για σας δεν υπήρχε ε, θεά ζώνη. εγώ νομίζω ότι υπάρχει, αυτό είναι το νόημα της απαντήσεώς μου. Σε κάθε νομοθεσία που καθορίζεται, έχετε τον κίνδυνο να ε, συμπεριλάβετε και μια θεά ζώνη και να προκληθούν διαφορετικές ερμηνείες. Και γι' αυτό είπα στην αρχή της ομιλίας μου ότι το θέμα εξαρτάται πρωτίστως από τις αφήνες νομοθεσίας. Εμείς συλλογικά, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο Συνομοθέτες οφείλουν να διασφαλίσουν ότι η νομοθεσία θα είναι σαφής, ακριβής, ώστε να αποφύγει οποιαδήποτε θεά ζώνη. Και στο παρελθόν, αλλά και στην προκείμενη υπόθεση, νομίζω ότι έχουμε θεές ζώνες. Και νομίζω ότι οι κατασκευαστές προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν αυτές τις θεές ζώνες. Ευχαριστώ. Σάλβα Μπιλικάινεν. Στα αγγλικά. Ο κύριο Σάλβα. Ευχαριστώ. Κύριε Φάλκενμπεργκ, επιθυμώ να σας ρωτήσω πώς αξιολογείτε τις ικανότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξέταση έρευνα των τεχνολογιών γύρω από το αυτοκίνητο για τη θέσπιση σχετικής νομοθεσίας. Απάντηση Φάλκενμπεργκ. Εγώ θα έλεγα να κάνετε την ερώτηση σας αυτή στην επόμενη συνεδρία. Δεν ήμουν εγώ, ε, δεν υπεύθυνο για αυτά τα πράγματα. Αυτό που μπορώ να σας πω ως παράδειγμα είναι το εξή. Ε, έμαθα μια ε, πληροφορήθηκα για μια αξιολόγηση της μελέτης της ICCT. Δύο εβδομάδες μετά από, την δυνατότητα, από τη στιγμή που είχαμε τη δυνατότητα να προσλάβουμε έναν έξτρα εμπειρογνώμονα στην εκεί μας διεύθυνση. Οι αριθμή του προσωπικού μας είναι ιδιαίτερα περιορισμένη και έχουμε και σημαντικές άλλες υποχρώσεις, συναντήσεις κλπ. Όλοι λοιπόν αντιμετωπίζουμε σημαντικό πρόβλημα χρόνου. Μπορώ λοιπόν μόνο να μιλήσω για τη Γενική Διεύθυνση για την οποία είμαι υπεύθυνο. Είμαστε αρκετά αραιοί, α το πω έτσι, σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό μας. Θα πρέπει να συζητήσετε ε, την στελέχωση της Γενικής διεύθυνση GROW με τον Γενικό Διευθυντή. Ευχαριστώ, λέει ο κ. Σάλβα, για την απάντησή σα. Παρακαλώ, ποια είναι η γνώμη σα σχετικά με το πλήθος εγκρίσεων τύπων που χορηγούνται από χώρες όπου δεν υπάρχει καν κατασκευή ε, αυτοκινήτων, όπως Λουξεμβούργο και Μάλτα. Απάντηση Φαλκενμπεργκ. Και αυτή η ερώτησή σας διαφεύγει τουλάχιστον των γνώσεών μου σχετικά με την νομοθεσία αυτή. Είμαι πεπισμένος ότι ο επόμενος που θα καθίσει εδώ στην θέση μου θα μπορέσει να σας δώσει μια στέρεα θεμελιωμένη απάντηση. Είδα στην νομοθεσία πάντως ότι την νομοθεσία για την χορήγηση εγκρίσεως τύπου την φέρουν οι χώρες μέλη. Τώρα, γιατί γίνεται και πώς γίνεται αυτό στις λεπτομέρειες διαφεύγει των γνώσεών μου. Σάλβα, είναι φυσιολογικό για σας σε τέτοιες χώρες να υπάρχουν τόσες πολλές εγκρίσεις τύπων, επαναλαμβάνω για από χώρε οι οποίε δεν κατασκευάζουν ούτε ένα αυτοκίνητο όχημα. Ε, ε, ε, Πετε μου τη γνώμη σα. Εγώ καταρχήν εμπιστεύομαι όλες τις ε, αρχές των χωρών μελών με τον ίδιο τρόπο. Έχω συζητήσει σε πολλά μέρη τις διαδικασίες επαλήθευσης συμμορφώσεως με ε, προδιαγραφές, ελέγχους κλπ. Και νομίζω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις που υπέπεσαν στην αντίληψή μου, οι περισσότερες χώρες μέλη έχουν κάποιους peer controls, δηλαδή ελέγχουν σωμοτήμων. Και ότι οι διαδικασίες αυτές είναι της ίδιας ποιότητας σε όλες τις χώρες μέλη. Θα έλεγα πάντως ότι ακόμη και αν δεν υπάρχει απευθείας κατασκευή οχημάτων ίσως τότε η Εθνική Αρχή να είναι πιο ανεξάρτητη από αρχή άλλης χώρας μέλους όπου υπάρχει κατασκευή αυτοκινήτων. Πάντως όλοι λειτουργούμε και κινούμεθα μέσα σε ένα ευρωπαϊκό δικαιοίκο σύστημα το οποίο αναγνωρίζει ότι είναι ισότιμες οι αρχές αυτές και ότι διέπει το έργο τους η ίδια ποιότητα. Ευχαριστώ Κάλμπαχ. Τι κάνετε κύριε Φάρκενπερκ Δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι από την αρχή μαζί σας. Έχασα άλλωστε και ένα μέρος της ανταλλαγής απόψεων. Άκουσα όμως την κυρία Ντάλη να σας ρωτά για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων και για την εμπειρογνωμοσύνη. Δεν νομίζετε ότι για λόγους διαφανείας οι εκπρόσωποι της αυτοκινητοβιομηχανίας θα πρέπει να ακούονται μόνο στις αρχικές φάσεις της διαδικασίας και ότι από εκεί και πέρα θα πρέπει να απαγορεύεται η αδίποτε επαφή. Δεν ζητούμε υπερβολικά πολλά από την αυτοκινητοβιομηχανία, αν δεν το πράξουμε αυτό δηλαδή. Δηλαδή να στραφεί κατά των ίδιων των συμφερόντων της. Φάλκενμπεργκ καπαντά. Δεν είναι βέβαιος ότι είναι κατά των συμφερόντων της αυτοκινητοβιομηχανίας η υπόθεση να καταλήξει σε κατασκευή περιβαλλοντικά ε, ενάρετων, να το πω έτσι, προϊόντων. Αντίθετα, μάλιστα, ακριβώς αυτό είναι το θέμα, γιατί έχουν παραχθεί και αυτοκίνητα τα οποία δεν σέβονταν τις προδιαγραφές αυτές. Δεν είμαι βέβαιος, λοιπόν, ότι θα συμφωνούσα εξ ορισμού ότι κάποια βιομηχανία έχει αυτομάτως συμφέρον να καταστρατηγεί περιβαλλοντικούς κανόνες, προδιαγραφές ή προδιαγραφές υγείας κλπ. Ωστόσο, δέχομαι την άποψή σας ότι θα πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός σε ό,τι αφορά την ε, επίκριση εμπειρογνωμοσύνης, αλλά ταυτόχρονα να καταστά απόλυτα σαφές και ποιος λαμβάνει την τελική απόφαση. Και αυτές είναι βεβαίως στην περίπτωση αυτέ οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτέ δηλαδή που έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν πρόταση. Βλέπετε τέτοια ανεξαρτησία, επιμένει η κυρία Κάλενμπαχ. Κοιτάξτε, 40 χρόνια υπηρετώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι τομεί όπου έχω υπηρετήσει, κοιτάξτε, νομίζω ότι στην πολύ μεγάλη ε, ε, πλειονότητα των υποθέσεων, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να θυμηθώ καμία υπόθεση όπου το να ακούσω την εμπειρογνωμοσύνη ή την άποψη αν θέλετε κάποιου τομέα της οικονομίας με οδήγησε ή μας οδήγησε να κινηθούμε προς μια κατεύθυνση. Διότι αν είχαμε ακούσει ε, τη βιομηχανία θα είχαμε ακούσει και ε, ταυτόχρονα και επιστημονικές ε, συμβουλές των ερευνητικών ιδρυμάτων, τις απόψεις της ε, κοινωνία των πολιτών και ούτω καθεξής και των υπολοιπών φορέων. Και μόνο υπό το φως όλων αυτών των απόψεων μπορεί κανείς να καταλήξει σε ε, λογικές αποφάσεις. Λόγος Βερμέχο. Όπως ε, ξέρουμε, η χρήση των ε, συσκευών αναστολής αυτών των συστημάτων δηλαδή που χρησιμοποιούνται απαγορεύεται από το 1998 για όλα τα οχήματα. Από αυτή την άποψη για την έγκριση νέων αυτοκινήτων θα ήθελα να ρωτήσω αν εσείς υποψιαζόσασταν τη χρήση συσκευών αναστολής. Πώς αιτιολογείτε ότι επιτράπηκε η κυκλοφορία αυτοκινήτων με εκπομπές πολύ ψηλότερες από το όριο. Δεν υποψιαστήκατε ότι οι εθνικές αρχές στη Γερμανία, την Αγγλία, τη Γαλλία, τις κατοχώρες στο Λουξεμβούργο, την Ισπανία, την Ιταλία, το Βέλγιο ενέκριναν την κυκλοφορία αυτοκινήτων που παραβίαζαν το ε, όρια. Και σε αυτή την περίπτωση, γιατί νομίζετε ότι δεν ξεκίνησε καμία διαδικασία κατά παράβαση ε, για αυτές τις υποθέσεις. Τέλος, θεωρείτε ότι είναι απαραίτητη μια νομοθεσία για την έγκριση οχημάτων αντί για μια οδηγία πλαίσιο. Falkenberg. Σε καμία φάση, δεν, σε καμία στιγμή μάλλον, δεν ε, σκέφτηκα ούτε μου είπε κανείς ότι υπήρχαν πρακτικές στα κρατημέλη παραβατικές. Και το είπα νομίζω και στις απαντήσεις μου τις γραπτές ότι δυσκολεύομαι να φανταστώ ότι οι αρμόδιες αρχές στα κρατημέλη έχουν ενεργήσει αντίθετα με τις νομοθετικές απαιτήσεις. Ισχύει το κράτος δικαίου στην Ευρώπη, η Ευρώπη σημαίνει σεβασμός του δικαίου και πραγματικά δυσκολεύομαι πάρα πολύ θα, να, το πιστέψω κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό να πω ακόμα μια φορά ότι πιστεύω ότι προφανώς υπήρχε πρόβλημα στην ερμηνεία, δηλαδή σε ποιο βαθμό ήταν δυνατόν να τραβήξουμε τα όρια αυτής της νομοθεσίας και το, αν τα κρατημέλη έπρεπε να είναι πιο προσεκτικά, πιο επιφυλακτικά, θα έπρεπε να θέσουν περισσότερες ερωτήσεις όταν συνειδητοποίησαν ότι υπήρχαν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις εργαστηριακές δοκιμές και τις ε, πραγματικές εκπομπές σε πραγματική οδήγηση. Ναι, θα έπρεπε να το έχουν κάνει, αλλά δεν πιστεύω πως ε, υπήρχαν ε, υποψίες για παράνομες πρακτικές τις οποίες στις οποίες εμέσως ή ε, αμέσως συμμετείχαν αμεσως συμμετειχαν τα κρατη μελη οι Ντέλη. Θέλω να επανέλθω σε αυτά που είπαμε πριν από λίγο, στην τελευταία μου ερώτηση και πάλι εσείς υποδεικνύετε την αδυναμία των εθνικών αρχών. Ξέρω πως αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους μας ξεπερνούν πέντε, κατά πέντε φορές τα επιτρεπόμενα όρια στις εκπομπές τους και ωστόσο πέρασαν επιτυχώς την περίφημη δοκιμή NEDC την εργαστηριακό κύκλο δοκιμισό. Για όλα αυτά συμφωνούμε μαζί σας. Τώρα όμως πρέπει να προβλέψουμε το μέλλον. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω τι μας προτείνετε για αυτό το περίφημο νέο σύστημα έγκρισης τύπου για τα οχήματα. Πιστεύετε, όπως πολλοί από μας ε, πιστεύουμε σε αυτή την Επιτροπή, ότι είναι η ώρα να θεσπιστεί μια πραγματική ευρωπαϊκή ανεξάρτητη αρχή που θα εποπτεύει ακριβώς αυτό που είπατε προηγουμένως, δηλαδή το θέμα της των αγορών, εποπτεία των αγορών, αλλά και το θέμα της έγκρισης τύπου για τα αυτοκίνητα. Είναι αυτή η γνώμη σας ότι πρέπει κάτι τέτοιο να γίνει. Πιστεύω ότι τα συστήματα που έχει συστηθεί μια ευρωπαϊκή αρχή έχουν δείξει την αξία τους. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε. Όμως αυτό εξαρτάται από τον ε, νομοθέτη, τους νομοθέτες, τα κράτη-μέλη, αλλά και ε, Συμβούλιο, Κομισιόν, Ευρωκοινοβούλιο να θεσπίσουν, να, να ορίσουν σε ποιο βαθμό είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Είμαι βέβαιος ότι ε, έχουμε προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε περισσότερες διαβεβαιώσεις ότι ερμηνεύουμε και εφαρμόζουμε την νομοθεσία που υιοθετείται εδώ με τρόπο συγκρίσιμο και ισότιμο για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Επικρότεια. Μάλιστα, συμφωνούμε απόλυτα. Εσείς έχετε κάποιο κάποια πορεία για την εργασία σας, πώς θα θεσπιστεί αύριο μεθαύριο αυτός ο νέος οργανισμός, γιατί μιλάμε για ανεξαρτησία, γιατί βεβαίως βλέπουμε ότι ο καθένας προσπαθεί κάπως να κάτι να υποφεληθεί από αυτή την νομοθεσία. Θα πρέπει να βασιστούμε στο αμερικανικό πρότυπο, δηλαδή αυτό τον οργανισμό περιβάλλοντος και υγείας ή πιστεύετε ότι πρέπει σταδιακά να προχωρήσουμε, να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό που θα εποπτεύει τις εθνικές αρχές ένα πρώτο χρόνο, ώστε αύριο μεθαύριο να, μπορούμε, να μπορεί να είναι τελείω ανεξάρτητη και να επιβάλλει και στις εθνικές αρχές τα δέοντα. Φάλκενμπεργκ. Πιστεύω ότι το πρώτο βήμα είναι η σωστή και ξεκαθαρή νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και επίτα ε, θα πρέπει να ασχοληθούμε με την εφαρμογή αυτής. Ε, και νομίζω ότι αυτό κάνουμε με την νομοθεσία για τις ε, δοκιμές, για τις πραγματικές εκπομπές. Θα έχουμε πολύ καλύτερη βάση κατά αυτόν τον τρόπο. Το επόμενο στάδιο θα είναι να αποφασίσουμε πώς θα επιβάλλουμε την συνεργασία είτε αποκεντρωμένα ανάμεσα στις αρχές των κρατών μελών ή θα πρέπει να φτιάξουμε κάτι πιο κεντρικό και πώς θα το ορίσουμε. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα ε, που θα μας απασχολήσει στο μέλλον και θα απασχολήσει τους διαδόχους μου. Ωραία ερώτηση αυτή για το μέλλον, για να κλείσουμε την ε, ακρόαση αυτή και πάλι να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ. Οι συνάδελφοι που θέλουν μπορούν να υποβάλουν και γραπτές ερωτήσεις πριν τις 18 του μηνός. Έχουμε ένα σύντομο διάλειμμα τώρα πριν να προχωρήσουμε στην επόμενη μας ακρόαση. Σας ευχαριστώ. Okay, colleagues, we can uh, move on Ας συνεχίσουμε τώρα με την δεύτερη ακούρασή μας. Έχουμε κοντά μας τον ε, κύριο Καλέχα Κρέσπο, πρώην Γενικό Διευθυντής, Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης GROW. Σας ευχαριστώ πολύ ε, κύριε που ε, δεχθήκα την πρόσκληση. Σας προσκαλέσαμε στην Επιτροπή μας, εμείς, υπό την ιδιότητά σας του πρώην Προέδρου, ε, συγγνώμη, του πρώην Γενικού Διευθυντού της ε, Γενικής Διευθύνσεως ε, ε, ε, ε ενιαίας αγοράς μικρομεσαίων επιχειρήσεων κλπ. μέχρι το 2015, διότι η Επιτροπή μας επιθυμεί να αντλήσει περισσότερες πληροφορίες για τα ε, ζητήματα που την απασχολούν. Έχουμε λάβει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τις απαντήσεις σας ενός πρώτου ερωτηματολογίου Έχουμε στη διάθεσή μας μία ώρα και 40 λεπτά για την συζήτηση μαζί σας και πολύ ευχαριστώ, θα σας δώσω το λόγο για να τοποθετηθείτε προφορικός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ντεμεσμάκερ, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Να ξαναέρθω ενώπιον τη Επιτροπή σα, γιατί ήμουν και στο πρώτο στην πρώτη ακρόαση ως Γενικός Διευθυντής της ε, Γενικής Διευθυντής Περιβάλλοντος ε, για να περιγράψω την κατάσταση. Με μεγάλη χαρά λοιπόν ξαναέρχομαι να σας δω και να σας μιλήσω ε, για τη θητεία μου στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων έως το 2015 και επιτρέψτε μου να κάνω και κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με την εμπειρία μου από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος από το Σεπτέμβριο του 2015. Ξεκινώ λοιπόν από την πρώτη περίοδο τα χρόνια της δράσης θα το ονομάσω και γιατί. Διότι όταν άρχισα ως Γενικός Διευθυντής, όταν έλαβα καθήκοντα στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων Enterprise και μετά Grow Ανάπτυξης, καθήκον μου ήταν να ε, ετοιμάσω την ανακοίνωση CARS 2020 και να προετοιμάσω την ε, εφαρμογή της. Η CARS 2020 ήταν ένα εγχείρημα άνευ προηγουμένου με την ε, κατάθεση μιας στρατηγικής συνολική για την αυτοκινητοβιομηχανία που θα επέτρεπε την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τη, τις δυνατότητες της για καινοτομία, της ασφάλειας αλλά και, πολύ σημαντικό, τη συμβολή της στην αηφορία. Ας, ξαναθυμηθούμε την κατάσταση που αντιμετωπίζαμε τότε. Βαθιά οικονομική κρίση, ανάγκη για ένα κατεπήγον σχέδιο για ένα τομέα που απασχολούσε 12 εκατομμύρια εργαζομένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεγαλύτερο βέβαια ιδιωτικό επενδυτή για την έρευνα και την καινοτομία που όμως ταυτόχρονα είχε κέρυες ευθύνες και για, την ε, βέλτιστη, για τις βέλτιστες συνθήκες ασφαλείας αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Και ξέρετε τι μεσολάβησε. Υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανακοίνωσή της τον Νοέμβριο του 2012 κατόπιν ε, ε, εκτεταμένων συζητήσεων με κράτη-μέλη, 7 επιτρόπους, 9 υπουργούς, ε, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Επιτροπή των Περιφερειών, 18 εμπλεκόμενους φορείς από τη βιομηχανία, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, με μια διαφανή, ανοιχτή και ε, χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία. Το Δεκέμβριο του 2012 εγκρίθηκε το σχέδιο και ένα χρόνο αργότερα, το Δεκέμβριο του 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, με τη σειρά του ενέκρινε το σχέδιο με τη συμφωνία της Επιτροπής Εμπορίου, Μεταφορών, Εσωτερικής Αγοράς και Απασχόλησης των τεσσάρων των επιτροπών. Ε, ένα κύριο ζήτημα λοιπόν ήταν οι, οι εκπομπέ σε πραγματικέ συνθήκε οδήγηση, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι συμφώνησαν με τη διάγνωση και παραθέτω αυτό που είχε υποθεί συγκεκριμένα, τα ισχύοντα μέτρα για τον υπολογισμό των ρήπων δεν αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης και υπόθηκε συγκεκριμένα οι εκπομπές οξυδίων του αζότου είναι σημαντικά υψηλότερες πραγματικές συνθήκες οδήγησης από ό,τι προβλέπεται στα όρια εκπομπών κατά την μέτρηση σε ε, συνθήκες εργαστηριακές. Ήταν σαφής η διάγνωση λοιπόν ότι το σύστημά μας δεν λειτουργούσε, το σύστημα είχε αποτύχει. Επιπλέον αυτού, πολλά κράτη-μέλη δεν τηρούν ακόμη την νομοθεσία ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Ξέρετε τα στοιχεία, 400.000 πρόωροι θάνατοι στην Ευρώπη, 70.000 εκ των οποίων συνδέονται με τον τομέα των μεταφορών. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε σχέδιο για την ανάπτυξη μιας νέας και πρωτοπόρου διαδικασίας μετρήσεων σε δοκιμές για τις εκπομπές των αυτοκίνητο σε πραγματικέ συνθήκε οδήγηση, αλλά και βελτίωση των εργαστηριακών δοκιμών. Και ορίστηκε ένα χρονοδιάγραμμα πολιτικό για, τις, ε, για τη δουλειά για τι πραγματικέ συνθήκε οδήγηση έω το τέλο, ε, έω την ώρα τη εισαγωγή του Euro 6, με την, μέχρι την πλήρη ε, εφαρμογή του συστήματος. Όλοι ήταν εν γνώση των μεγάλων αποκλήσεων ε, μεταξύ των εργαστηριακών δοκιμών και του RD. Κανείς δεν ε, αμφισβήτησε την προσέγγιση ή το χρονοδιάγραμμα. Όλοι συμφώνησαν ότι αυτό ήταν ο καλύτερο τρόπος να προχωρήσουμε. Όλοι επίσης συμφωνήσαμε ότι για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση έπρεπε να δώσουμε έμφαση σε δύο τομείς εργασίας. Καταρχάς μεταρρύθμιση τη διαδικασία έγκρισης τύπου και δεύτερον ενίσχυση της εποπτείας. Οι διαδικασίες λοιπόν Έγκριση τύπου και η εποπτεία της αγοράς αποτελούν δύο του ίδιου νομίσματος. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή επέτυχε και εγώ κατά την ε, θητεία μου ως Γενικός Διευθυντής να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, να την ολοκληρώσουμε, να εξασφαλίσουμε μέχρι το Μάιο του 2014 την έγκριση του ε, συστήματος μέτρησης με το ΠΕΠΣ ως σύστημα υποχρεωτικό για την έγκριση τύπου ήταν μια πραγματική λοιπόν σημαντική και ριζική αλλαγή αυτή την οποία επιτύχαμε. Και επίσης ετοιμάσαμε το έδαφος για το δεύτερο ε, τεστ ε, πραγματικών συνθήκων οδήγησης που εντελειοθετήθηκε και το WLTP, το παγκόσμιο δηλαδή σύστημα, το οποίο στη συνέχεια υιοθετήθηκε προκειμένου να αντικαταστήσει το νέο ευρωπαϊκό ε, σύστημα οδήγησης η κύκλο οδήγησης. Και φεύγοντας από το, θέση ως Γενικού Διευθυντή της Enterprise, είχα ήδη έτοιμο το σύστημα αποπτίας της αγοράς, το οποίο στη συνέχεια ε, με κάποιες μικροαλλαγές ε, κατετέθη για να ε, δημοσιευθεί τον Ιανουάριο του 2016. Ξέρω ότι ιδιαίτερα μεριμνά λοιπόν η Επιτροπή σας για τη διερεύνηση του κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβράδυνε τη διαδικασία για την εισαγωγή των νέων δοκιμών. Είναι από τα ζητήματα που σας απασχολούν. Επιτρέψτε μου λοιπόν να μιλήσω περίφραστη. Ο κανονισμό 715 του 2007 έδινε στην Επιτροπή την εντολή, τη δυνατότητα για την ανάπτυξη νέων δοκιμών. Ξεκινήσαμε αμέσω τη δουλειά. Η DG Enterprise ήταν πρωτοπόρο σε στενή συνεργασία με άλλε γενικέ διευθύνσει, μεταξύ των οποίων και η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντο. Συνεργαστήκαμε στενά με το Κοινό Κέντρο Ερευνών, για να, το οποίο ανέπτυξε δύο, ε, δύο μελέτε και αναπτύξαμε επίση την ομάδα εργασία πραγματικών συνθήκων οδήγηση ω ένα χώρο συζήτηση αυτών των πραγματικών συνθήκων οδήγηση. Και δεν ήθελα εδώ να αποτίσω φόρο τιμή σε όλου του εμπλεκόμενου συναδέλφου, γιατί είχαμε περιορισμένου πόρου. Αναφέρθηκε νωρίτερα και από τον κύριο Φάλκεμπεργκ το πρόβλημα αυτό. Ωστόσο, κάναμε πολλή δουλειά το Κοινό Κέντρο Ερευνών και εμεί και σε στενή συνεργασία με όλε τι υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπής καταφέραμε αυτό το αποτέλεσμα. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών στην έκθεση ε, που διατύπωσε ανέλυε δύο διαφορετικούς τύπους ε, μελέτης εκπομπών. Έπρεπε να αλλάξει το σύστημα λοιπόν, το να αναντηθεί. Καταρχάς είχαμε τους ε, τυχαίους κύκλους και δεύτερον είχαμε τα φορητά συστήματα μέτρησης, τα PEPS δηλαδή. Ε, δύο συστήματα τα οποία ήταν και τα δύο εφικτά. Ωστόσο, το Κοινό Κέντρο Ερευνών κατέληξε ότι τα ΠΕΠ, e στα φορητά συστήματα, ήταν πολύ πιο αποτελεσματικά για την καταγραφή των πραγματικών των εκπομπών σε πραγματικέ συνθήκε οδήγηση, αλλά και για να αντιμετωπίσει τα συστήματα αναστολή. Ταυτόχρονα το 2014 το Κοινό Κέντρο Ερευνών με την έκθεση αυτή μα είπε ότι δεν υπήρχε επάρκεια ε, φορητών συστημάτων, ότι υπήρχαν γεωγραφικοί, κλιματολογικοί ε, περιορισμοί, περιορισμοί σχετικοί με τη θερμοκρασία, ότι θα σήμαινε αυτό, αυτή η εισαγωγή επιπλέον κόστος και ότι έπρεπε να αξιολογήσουμε τους γενικότερους όρους και για τις θερμοκρασίες ε, δοκιμών, παραδείγματι, τι είδου επίδραση θα μπορούσαμε να έχουμε στα αποτελέσματα. Χρειαζόταν λοιπόν περισσότερη δουλειά και γι' αυτό εκλήθη το Κοινό Κέντρο Ερευνών αναπτύξει μια διαδικασία PEPS και θα ήθελα εδώ να υπενθυμίσω υπενθυμίσω ότι η αυτοκινητοβιομηχανία προτιμούσε τον τυχαίο κύκλο, δεν ε, προτιμούσε την ιδέα των ΠΕΠΣ, της άρεσε η ιδέα των ΠΕΠΣ, αλλά δεν ακολουθήσαμε τη θέση της. Επίσης, συμφωνήθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστήριξε αυτά τα συστήματα σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης ως μια συμπληρωματική διαδικασία για το παγκόσμιο σύστημα, το οποίο εν τέλει υιοθετήθηκε στο συγγνώμη που αναφέρομαι συνέχεια σε ακρονίμια, αλλά εάν χρειαστεί να πω αναλυτικά τα ονόματα όλων αυτών των συστημάτων, χάνω πολύ χρόνο. Συμφωνήθηκε λοιπόν ότι το το νέο σύστημα δοκιμών θα υιοθετούνταν μέχρι το 2017 ε, ο χρόνος έπαιζε σημαντικό ρόλο, πολλά ήταν τα διαφορετικά συστήματα, τα συμφέροντα, τα πολιτικά περίπλοκο το ζήτημα, μια μεγάλη πρόκληση λοιπόν. Καμία άλλη περιοχή στον κόσμο δεν είχε και δεν έχει αποδειχθεί σε αντίστοιχο εγχείρημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για άλλη μια φορά ήταν πρωτοπόρο στον χώρο τη αυτοκινητοβιομηχανία, στον τομέα αυτών. Ξέρετε ότι οι προδιαγραφέ μα σε μεγάλο βαθμό ε, είναι ε, παγκόσμια εμβέλεια. Ολοκληρώθηκε λοιπόν τον Απρίλιο του 2014 η δουλειά με την παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της αρχιτεκτονικής του συστήματος πραγματικών συνθήκων οδήγησης, συνεννόηση με τις ε, υπηρεσίες, με τέσσερα νομοθετήματα πάνω στα οποία είχαμε συμφωνήσει ότι θα πρέπει να κατευθούν για να διευκολυνθεί και η έγκριση και πολύ σωστά επιλέξαμε αυτή την ε, λύση, παρότι θεωρήθηκε ότι μπορεί να αποδυναμώνει το CARS 2020, όμως το νέο σύστημα, η νέα δοκιμή, συζητήθηκε το 2014 στην Επιτροπή Αυτοκινήτων, Οχημάτων με Κινητήρα και συζητήθηκε σε όλε τι συνεδριάσει τη σχετική επιτροπή. Αυτό, όμω ω επιτροπή δεν μπορούσαμε να περάσουμε στην έγκριση αυτού του συστήματο, γιατί χρειαζόταν η επιτροπολογία και η ειδική, πλειονό... η... ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών. Εν προκειμένου, ο συνάδελφο και φίλο Καρλ Φάλκεμπεργκ όντω μου απέστειλε επιστολή λέγοντα ότι ε, τρέφει ανησυχίε για την καθυστέρηση του σχετικού ζητήματο. Η απάντησή μου, την οποία έχω και διαβιβάσει στην επιτροπή σα, ήταν σαφέστατη και ε, έλεγε ότι δεν είμαστε ε, δεκτική εναντιασδήποτε καθυστέρησης ή υποβάθμισης των ορών ε, της νομοθεσίας, αλλά Έλεγα, ε, του εξηγούσα ότι οι συζητήσει ήταν ε, μακροχρόνιε και έρχονταν προτάσει τελευταία στιγμή, οι οποίε ήμασταν υποχρεωμένοι να εξετάσουμε. Ήταν η πρώτη φορά που κάποιο προέβαινε στην εισαγωγή συστήματο πραγματικών συνθηκών οδήγηση για τι δοκιμέ σε ολόκληρο τον κόσμο. Άρα ήταν ένα νέο σύστημα και έπρεπε να κάνουμε το καλύτερο για να το επαληθεύσουμε. Έτσι λοιπόν το Μάιο του 2015 υιοθετήθηκε. Βεβαίω θέλαμε να έχουμε την υιοθέτηση τον Σεπτέμβριο του 2014. Μια μικρή καθυστέρηση μερικών μηνών έω το Μάιο του 2015 όντω ε, έλαβε χώρα με μια νέα επιτροπή το 2014, με νέα δομή, με νέα διαδικασία έγκριση και από, ε, από την Επιτροπή Συλλογικό Όργανο, μην το ξεχνάμε αυτό, και βέβαια την ειδική πλειοψηφία για το Μάρτιο του 2015 και εν τέλει την έγκριση μετά την έγκριση από το Συμβούλιο από την ε, Επιτροπολογία το Μάιο του 2015. Όλες αυτές οι διαδικασίες με τις ε, υπηρεσίε Επιτροπής, την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, ε, και τη δική μας κλπ. Και ο κύριος Φάλκενμπεργκ ε, συμφώνησε το Μάρτιο του 2015 για το νέο αυτό σύστημα. Ξέρω ότι η Επιτροπή σας μελετά επίσης και τα συστήματα αναστολής, συσκευές αναστολής. Ξέρω ότι είναι ακαθόδεστο το ζήτημα, συναρπαστικό κιόλα και το να ορίσουμε τι ακριβώς συζητούμε. Θα πρέπει να αναφέρω ότι οι συσκευές αναστολής είναι παράνομες, απαγορεύονται το 1998 από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Εσδήποτε αυτοκίνητο κατασκευές της αυτοκίνητο χρησιμοποιεί πρέπει να ε, τιμωρείται και πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να τηρηθεί αυτή η νομοθεσία και να, να επιβληθούν οι απαγορεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σε θέση να διαγνώσει αποκλήσει ε, οφειλόμενε στο γεγονό ότι ήταν πεπαλαιωμένα τα συστήματα των δοκιμών. Ωστόσο, η εισαγωγή των πραγματικών ε, συνθηκών οδήγηση του νέου αυτού τεστ ξέραμε ότι θα μειώσει τι αποκλήσει και ω εκ τούτου τον κίνδυνο τη παρέμβαση των συσκευών αναστολή, όπω άλλωστε μα είχαν διαβεβαιώσει. Για να ολοκληρώσω λοιπόν για τα δύο τελευταία χρόνια στην Επιτροπή Περιβάλλοντο, αν μου επιτρέπει ο Πρόεδρο, πολύ σύντομα, αναλαμβάνοντα καθήκοντα στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντο, ε, βλέπω να ε, ξεσπάει το σκάνδαλο Volkswagen με σημαντική ε, βλάβη για την φήμη της ε, αυτοκινητοβιομηχανία τη Ευρώπη. Εξεπλάγημεν. Και εγώ προσωπικώ εξοργίστηκα κιόλα, γιατί ω πρώην Γενικό Διευθυντή της Επιτροπή τη Γενική Διεύθυνση για την για, το, για, την, ε, για τις επιχειρήσεις, για την ανάπτυξη, θα έπρεπε να είμαι εν γνώση αυτών. λοιπόν, ζήτησα πρώτα απ' όλα ως Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος να έχω κάθε στοιχείο στη θέση μου, να ζητήσω από τα κράτη-μέλη να ε, μου δώσουν κάθε στοιχείο και από τις Εθνικές Δικαστικές Αρχές, οι ανακριτικές αρχές. Δεύτερον, ήθελα να επαληθεύσω εάν υπάρχει περίπτωση να ε, χωρεί εδώ εφαρμογή τη νομοθεσία τη οδηγία συγκεκριμένα τη σχετική με το περιβάλλον, γιατί δηλαδή οι Αμερικανοί να μπορούν να επιβάλλουν κυρώσει και όχι εμεί. Δυστυχώ όμω από την νομική ανάλυση διαπιστώσαμε ότι αυτή η οδηγία δεν καλύπτει εκπομπέ, καλύπτει μόνο βιοπικιλότητα, ύδατα ε, και ω εκ τούτου δεν είχαμε τη δυνατότητα να ε, προξενήσουμε ε, επιβολή κυρώσεων δυνάμει αυτή τη οδηγία. Ζητήσαμε λοιπόν ανάληψη δράσεω, ε, αλλαγή διαδικασιών δεν θα αρκούσε μόνο, θα χρειάζονταν και πολλά άλλα μέτρα και φορολογικά ακόμη και επιτύχαμε και θα ήθελα επί τη ευκαιρία να προσφέρω φόρο τιμή ε, στου ευρωβουλευτέ που είναι εδώ παρόντε, γιατί καταφέραμε να εξασφαλίσουμε ανώτατα επίπεδα σε εθνικό επίπεδο που θα μειώσουν σημαντικά τα προβλήματα και τις συνέπειες της μόλυνσης ω το 2030. Παρακολουθούμε και διώκουμε όποιες παραβιάσεις έχουμε ε, τις ε, προσφυγές που έχουμε κατά των κρατών μελών για τις παραβιάσεις ε, της νομοθεσίας, 29 το σύνολο, τις οποίες παραπέμπουμε για δίκη και στόχο μα είναι να αποκαταστήσουμε και την εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην αυτοκινητοβιομηχανία τη Ευρώπη και για να ολοκληρώσω θα ήθελα να αναφέρω την εξή σκέψη ότι η κρίση τη Volkswagen αποδεικνύει ότι είναι πολύ απαραίτητο να γίνει σωστή διάγνωση του ότι συνέβη και ασφαλώ αυτό το ρόλο θα διαρμετήσει τη Δική Επιτροπή. Πρέπει να αντλήσουμε τα διδάγματα για να αποφύγουμε στο μέλλον αντίστοιχε κατα... καταστάσει, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει και να ολοκληρώσουμε την ε, μεταρρύθμισή μα για τι πραγματικέ συνθήκε οδήγηση γιατί εδώ ακριβώς έχουμε τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων. Δεύτερον, πρέπει να ενισχύσουμε το σύστημα έγκρισης τύπου και της εποπτείας της αγοράς ταυτόχρονα, αλλά πρέπει επίσης να βελτιωθεί και η διακυβέρνηση των συστημάτων μας. Ένα από τα διδάγματα από την κρίση αυτή είναι ότι η Ευρώπη πληρώνει βαρύτα το τίμημα της κατακαιρματισμένης της προσέγγισης και από την εμπειρία που έχω συλλέξει όλα αυτά τα χρόνια στην Επιτροπή διαπιστώνω ότι αυτό σημαίνει έναν ισχυρό μηχανισμό εποπτείας και των φορέων και των εθνικών αρχών για το αυτοκίνητο. Γιατί δεν υπάρχει άλλο το μέσο μεταφορών αυτή τη στιγμή και αυτό προτείνουμε άλλωστε και κατά την έγκριση του ε, και κατά τη μεταρρύθμιση του, της έγκρισης τύπου. Χωρίς να θέλουμε να, θέσουμε, να βάλουμε στο δόλιο του κατηγορουμένου κανέναν, πρέπει να βρούμε τα κατάλληλε λύσει. Είναι καθοριστική στιγμή. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που μας προσφέρετε. Θα είναι κρίσιμη η προσπάθεια που θα καταβάλουμε όλοι, το δικό σας το έργο ιδιαίτερος, για να βελτιώσουμε το, την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και την υγεία όλων των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη που μακρηγόρησα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ε, και τώρα θα προχωρήσουμε στον πρώτο γύρο ε, ερωτήσεων. Θα ξεκινήσουμε με τους εισηγητές ε, και στη συνέχεια θα έχουμε έναν εκπρόσωπο από κάθε πολιτική ομάδα. Για αυτό τον πρώτο γύρο θα έχουν ο καθένας πέντε λεπτά. Παρακαλώ λοιπόν να κρατήσετε το χρόνο, να τηρήσετε το χρόνο αυτό. Οι ευρωβουλευτέ έχουν τη δυνατότητα να σας διακόψουν στις απαντήσεις σας και να θέσουν επερωτήσεις, αλλά φυσικά χωρίς να ξεπερνούν το σύνολο των 5 λεπτών. Ξεκινάμε με τον κύριο Γκερμπράντι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς και Κρέσπο που επανέρχεστε ενώπιόν μας. Και πρώτα το Κοινοβούλιο έχει ψηφίσει ψήφισμα για το ΚΑΡ 2020, έχει όμως ασκήσει κριτική στην καθυστέρηση ε, των ε, δοκιμών. Και ζητήσαμε να εφαρμοστούν αυτές χωρίς καμία καθυστέρηση. Τώρα, η ερώτησή μου όπως έχει κάποιο άλλο νόημα. Είδαμε εσωτερικές επικοινωνίες μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Enterprise επίσης ε, ε, άλλων γενικών διευθύνσεων και του Κοινού Κέντρου Ερευνών και από τότε που μπήκατε ε, εσείς στη Γενική Διεύθυνση της Διεύθυνσης Crow όπου εκφράζεται υποψία οι υποψίες για την χρήση διατάξεων αναστολής. Είχατε εσείς κάποια γνώση. Σας ευχαριστώ, απαντά κύριο κ. Κρέσπο. Υπενθυμίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναφέρομαι στο πρώτο σας ε, θέμα, αναφέρ, ε, ε, ζητεί μάλλον χωρίς καμία καθυστέρηση την εφαρμογή των, των δοκιμών. Αλλά βεβαίω έχουμε κάποια τεχνικά θέματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά email, δεν είχα καμία γνώση. Αυτό όμως είναι ανησυχητικό, επιμένει ο κ. Γκέρμπραντι, διότι πρόκειται για πάρα πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα του Κοινού Κέντρου Ερευνών και οι άνθρωποι σας θα έπρεπε να σας είχαν ενημερώσει και εσείς με τη σειρά σας θα έπρεπε να είχατε ενημερώσει τον πολιτικά υπεύθυνο επίτροπο. Τέλος πάντων, το ψάχνουμε ακόμη. Η δεύτερη ερώτησή μου αναφέρεται στην δήλωσή σας. Είπατε δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή αναλάβατε τη Γενική Διεύθυνση ε, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Έχετε κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για διάφορε παραβιάσεις κλπ. Όμως, ως Γενικός Διευθυντής στοχεύεται περισσότερο στα μακροπρόθεσμα. Ταυτόχρονα είχατε ισχυρές ενδείξεις και μετά από ενημέρωση των συναδέλφων σας της DG Envy ότι η εφαρμογή δηλαδή της υφιστάμενης νομοθεσίας πόρο απήχε από το να είναι τέλεια. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι γιατί ποτέ δεν ενημερώσατε ή δεν ζητήσατε από τις χώρες μέλη πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για την εφαρμογή της ε, υφιστάμενης νομοθεσίας. Και επίσης αυτό που μας είπε ο κ. Φάλκενμπεργκ προηγουμένως, απόλυτη έλλειψη εποπτείας των αγορών από πλευράς Γιατί δεν μας είπατε τίποτα, γιατί ε, ε, δεν είπατε τίποτα, ενώ ήταν, σας ήταν γνωστά. Καγέχα ή Κρέσπο, απαντά. Στην Γενική Διεύθυνση Enterprise βασική, βασικός μας στόχος ήταν να αλλάξουμε το σύστημα δοκιμών, το οποίο δεν απέριδε επαρκώς δεν ήταν αντιπροσωπευτικό. Να ε, φτιάξουμε λοιπόν τις Real Driving Emissions. Κάθε φορά που είχαμε ε, πληροφορίες για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό στις χώρες μέλη, αντιδρούσαμε. Θυμούμε ε, για παράδειγμα την διαδικασία MAC. Σε ό,τι αφορά την νομοθεσία εγκρίσεως τύπων, υπάρχει οδηγία, η οποία εφαρμόζεται από τις χώρες μέλη, αλλά το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο προβαίνει σε καταμερισμό των ευθυνών ρυθμιστής είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι χώρες μέλη εφαρμόζουν την νομοθεσία και η αυτοκινητοβιομηχανία συμμορφώνεται. Οι χώρες μέλη λοιπόν είναι οι αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή. Κάθε φορά που έχουμε στοιχεία ότι μια χώρα μέλος δεν ασκεί τον ρόλο της, της επιβολής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να προσφύγει κατά τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ναι, αλλά υπάρχει μια διαδικασία πριν από το δικαστήριο, λέει ο κ. Κερμπράντη, πριν να ξεκινήσετε την διαδικασία για παράληψη. Να ζητήσετε πληροφορίε. Η ΔΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πολλέ πληροφορίε ότι οι χώρε μέλη δεν εφαρμόζουν ή δεν επιβάλλουν την εφαρμογή τη υφιστάμενη νομοθεσία. Και δεν τέθηκε ποτέ κανένα θέμα προ τι χώρε μέλη για τα πράγματα αυτά. Κρέσπο. Ποτέ δεν είχαμε πληροφορίε σε ό,τι αφορά την παράληψη των χωρών μελών εφαρμογή νομοθεσία. Αυτό που γνωρίζαμε ήταν ότι τα αυτοκίνητα υπερεύαιναν τα όρια και εμεί το αποδίδαμε αυτό στην έλλειψη αντιπροσωπευτικότητα των ε, κύκλων δοκιμών. Κύριε Μπράντι, μία ακόμη ερώτηση. Μίλησα με ανθρώπους που ήταν αναμειγμένοι στη διαδικασία αυτή και μου είπαν ότι υπήρχαν τόσοι πολλοί εκπρόσωποι από την αυτοκινητοβιομηχανία και τόσο λίγοι εκπρόσωποι των χωρών μελών. Δεν συντάσσονται πρακτικά των συναντήσεων και αυτά για την ανάπτυξη των νέων RDE, Road Driving Emissions δηλαδή. Εάν είχατε προσπαθήσει να οργανώσετε μια θεσμική απάντηση, διότι όλοι τελικώ δυσαρεστούνταν επειδή δεν λαμβάνονταν απαντήσει, δεν λαμβάνονταν αποφάσεις μάλλον και υπήρχε καθυστέρηση στη διαδικασία. Γιατί δεν φροντίζεται να υπάρχουν δύο, τρει, τέσσερι εκπρόσωποι τη βιομηχανία και όχι 30-40. Κρέσπο. Επιθυμώ να τονίσω ότι υπήρχαν πρακτικά όλων των συναντήσεων που γίνονταν στην Τεχνική Επιτροπή Αυτοκινήτων Οχημάτων και μάλιστα τα έχω εδώ, δείχνω το φάκελο, Είχαμε και την ομάδα εργασίας Real Driving Emissions των ε, ελαφρών οχημάτων, ανοιχτή σε όλους και με εκπροσώπηση από το ICCT κλπ. Δεν είναι κλειστά τα πράγματα αυτά, οι συναντήσεις αυτές. Λογικό είναι βέβαια όταν προχωρείτε σε μεταρρυθμίσει στην νομοθεσία που διέπει ένα τομέα, ο τομέας να την παρακολουθεί προσεκτικά. Αλλά μπορώ να σας δώσω τα πρακτικά της Τεχνικής Επιτροπής Αυτοκινήτων Οχημάτων. Επίσης τα όσα έχει κάνει η Τεχνική Επιτροπή για τις RDE. Ο κύριος Σάλβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ κύριε Καγιέχα που είστε εκ νέου σήμερα εδώ για την διάθεσή σας να εργαστείτε με την ερευνητική μας αυτή επιτροπή. Θα ήθελα να επανέλθω στο ερώτημα του κατά πόσο κάποια στιγμή εσείς είχατε απόδειξη για υπόθεση παραβίασης της νομοθεσίας ε, περί εκπομπών από πλευράς κάποιου κατασκευαστή αυτοκινήτων και τι κάνατε σχετικά. Να σας πω μια υπόθεση που είχα στη διάρκεια της εντολής μου και μπορώ να σας μιλήσω για το τι έκανα. Μέσω ενός ανακοινοθέντος τύπου το Σεπτέμβριο του 2012 μια εταιρεία, η Daimler-Benz, Benz ανακοινώνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το ψυκτικό που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία γιατί πιστεύει πως υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας με το συγκεκριμένο και θα θέσει στην αγορά ε, αυτοκίνητα που θα ξεπερνούσαν τις επιτρεπόμενες εκπομπές. Τι έκανα εκείνη τη στιγμή. Κάναμε μια συνεδρίαση με την επιχείρηση. Ε, άμεσα ενημερώσαμε το τις ε, εποπτικές αρχές της Γερμανίας. Mm, οι ε, γερμανικές αρχές μας είπαν ότι υπήρχαν αμφιβολίες όσον αφορά την ασφάλεια αυτού του νέου ψυκτικού υγρού και άμεσα ζητήσαμε από το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο να λάβει θέση για το κατά πόσο ήταν σωστή ή όχι η ανάλυση ασφάλειας. Ε, το GRC μας είπε πως αυτό το ψυκτικό υγρό δεν ε, παρουσιάζει προβλήματα ασφαλείας. Εγώ προσωπικά πήγα στην Τεχνική Επιτροπή των Αυτοκινήτων για να θέσω το ζήτημα σε όλα τα κράτη-μέλη ανακαλύψαμε πως υπήρχαν ε, αυτοκίνητα που είχαν τεθεί στην αγορά με ένα παλαιο, παλιό, ε, παλιά έγκριση τύπου. Ξεκινήσαμε τις κατάλληλες διαδικασίες, ανακαλύψαμε ότι υπήρχε πρόβλημα με την νομοθεσία Type Approval, έγκριση τύπου και όχι μόνο με τη Γερμανία αλλά και με το Ηνωμένο Βασίλειο, το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο. Οι τέσσερις ε, ε, ήταν, έγιναν μάλλον αντικείμενο νομικής διαδικασίας και μετά αφού πήραμε εξηγήσει, ε, η υπόθεση έφτασε στην, σε απόφαση της Επιτροπής να παστραφούμε στο 10 μετά από την καταπαράβαση διαδικασία και μετά από την αιτιολογημένη έκθεση. Η σταμάτησε όλα τα αυτοκίνητα στα σύνορα με τη Γερμανία και ε, στράφει στο δικατιστικό της σύστημα. Ήθελα να σας πω ότι η Κομισιόν ε, άσκησε τα καθήκοντά της ως θεματοφύλακα των συνθήκων εφόσον ε, είδαμε ότι υπήρχε πρόβλημα και αδράνεια του κράτους μέλους για να εφαρμόσει το κοινοτικό δίκαιο και η Κομισιόν προέβησε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να τηρηθεί το ευρωπαϊκό δίκαιο και μάλιστα Υπό το φως όλων αυτών αποφασίσαμε να αναμορφώσουμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί της έγκρισης τύπου γιατί προφανώς υπήρχε πρόβλημα γιατί τα κράτη μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν επιστοποιητικά έγκρισης τύπου παλιά για νέα οχήματα. Ε, αυτή η πρόταση ετέθη και είναι ένα σημαντικό στοιχείο για το ότι αυτή η η Επιτροπή παρακολουθεί τα τεκτενόμενα και είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο να το εγκρίνουν. Γιατί τόσο σημαντικό όσο η αλλαγή τη δοκιμή είναι και η εποπτεία τη αγορά. Άρα λοιπόν όλα αυτά ήταν ε, επιβεβαιωμένα και γνωρίζετε ότι ξέρουμε πως λάβατε μια ανεπιστολή ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές, που έλεγε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δοκιμές στο εργαστήριο και στις δοκιμές σε συνθήκες πραγματικής οδήγησης. Γιατί δεν έγινε μια τέτοια συνεδρίαση ανάμεσα στους κατασκευαστές, με τους κατασκευαστές όταν σας έστειλε την επιστολή ο κ. Φάλκενμπεργκ. Κοιτάξτε, ο κ. Φάλκενμπεργκ μου επεξήγησε την ανησυχία του για την καθυστέρηση στην έγκριση του νέου τεστ της μεταρρύθμισης δηλαδή του, ε, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του Real Diving Emissions, του RDE. Και εγώ το απάντησα και νομίζω ότι η απάντησή μου είναι πολύ σαφής. Και έλεγα ότι ήταν η προσωπική μου δέσμευση και ότι δουλεύουμε για να επιτύχουμε να εγκριθεί όσο γίνεται πιο σύντομα αλλά δυστυχώ έλειπε η ειδική πλειοψηφία. Και μάλιστα του είπα ότι δεν θα καταφέρουμε διατάξει αυτέ. δεν θα επιτρέψουμε μάλλον να αποδυναμωθούν αυτέ οι διατάξεις. Ε, το κοινοτικό δίκαιο εμένα δεν μου επιτρέπει να ξεκινήσω διαδικασία έρευνας κατά κάποιου κατασκευαστή. Αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και τα κράτη-μέλη, αφού έμαθαν αυτή την έκθεση που είχε παρουσιαστεί στην ομάδα περί Real Driving Emissions, RD, έπρεπε να δράσουν. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να τους καταγράψουμε, να, τους, να, να ανοίξουμε έρευνες για τις επιχειρήσεις κτλ. Πάντως η νομοθεσία δεν μας επιτρέπει να πάμε να ε, ερευνήσουμε ή να ε, τιμωρήσουμε τους κατασκευαστές. Τα κράτη-μέλη πρέπει να το κάνουν. Μας επιτρέπει να ενημερώσουμε τα κράτη-μέλη και να τα καλέσουμε να λάβουν δράση. Αυτά. Ευχαριστώ κύριο Σκάριντς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούω με πολύ ενδιαφέρον. Ε, καλό που ήρθατε πάλι. Θα σας ε, κάνω μια ευθεία ερώτηση. Ε, κατά τη γνώμη σας, στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ανάπτυξης του RDE, υπήρξε κάποια ισχυρή και επιτυχής προσπάθεια είτε από πλευρά τη Επιτροπή ή κάποιου επιτρόπου είτε από τη βιομηχανία που προσπαθούσε να σταματήσει, να καθυστερήσει την ανάπτυξη της δοκιμής αρδί. Υπήρχε κανείς που κρατούσε αντίσταση ή που έβαζε εμπόδια ε, στην διαδικασία. Από πλευρά τη Κομισιόν όχι, σε καμία περίπτωση το αντίθετο μάλιστα. Είχαμε την υποχρέωση να το ολοκληρώσουμε όσο γινόταν πιο σύντομα. Όλα τα κράτη-μέλη ε, ήταν ε, διαθέσιμα, δεν ήταν ε, αντίθετα, αλλά θέλανε να είναι βέβαια ότι θα λειτουργήσει το σύστημα και από πλευρά τη βιομηχανία είναι γνωστό τη σπάσει, ότι δεν του άρεσε το σύστημα του ΠΕΜΣ, των φορητών ε, συσκευών ελέγχου, αλλά ότι προχωρούσαν ένα, προτιμούσαν έναν κύκλο τυχαίο, όχι όμω αυτό που τελικά εγκρίναμε για τι συνθήκε πραγματική οδήγηση. Και αυτό φαίνεται και το 2013 στην έκθεση που λέει ότι εδώ έχουμε δύο συστήματα. Υπάρχει ένα το οποίο προτιμάει η Κομισιόν και τα Κράτη-Μέλη γιατί πιο πολύ αυτό προσαρμόζεται στην πραγματική οδήγηση. Και υπάρχει και το, η άλλη δοκιμή που είναι ενό τυχαίου κύκλου ε, τη στιγμή επαλήθευση ελέγχου του αυτοκινήτου. Τελικά εγκρίθηκε αυτό που θέλανε τα Κράτη-Μέλη και η Κομισιόν και η αυτοκινητοβιομηχανία χρειάστηκε να προσαρμοστεί σε αυτό. Okay, so Μάλιστα. Αυτό που είπατε τώρα και αυτό που είπατε και στην προηγούμενη σας δήλωση είναι ότι η διαδικασία πήρε χρόνο, αλλά κανείς δεν την παρεμπόδιζε. Όχι επειδή κάποιος την παρεμπόδιζε. Κατά τη γνώμη σας, τι θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον, γιατί εφόσον κανείς δεν την καθυστερούσε η διαδικασία, θα μπορούσε να πει ότι τα 7 ή τα 10 χρόνια είναι πολύ μεγάλο, μακρύ χρονικό διάστημα για την ανάπτυξη τέτοια νομοθεσία ή διαδικασία δοκιμών που έχει άμεση επίπτωση στην δημόσια υγεία. Τι πρέπει να αλλάξει στο σύστημα ώστε την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να αλλάξει η νομοθεσία να μην πάρει τόσο πολύ χρόνο. Ή, είναι... ή δεν υπάρχει τρόπος να ε, επιταχυνθεί η διαδικασία στο μέλλον. Να πω τα δύο, δύο. Πρώτα απ' όλα καταφέραμε να το ολοκληρώσουμε στη δική μου θητεία ως ε, Γενικού Διευθυντή σε μια τριετία. Γιατί δεν τα καταφέραμε νωρίτερα, γιατί νωρίτερα δεν είχαμε τη στήριξη και την πολιτική εντολή όλων των θεσμών, όλων των αυτοκινητοβιομήχανων, όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. Αυτό έγινε το Νοέμβριο του 2012. Όταν λάβαμε την φούλη εντολή το Νοέμβριο, μπορούσαμε και είχαμε ήδη ξεκινήσει το, το, από το 2011 εμείς με το GRC. Αλλά αν δείτε, το χρόνο που μας πήρε να τα καταφέρουμε ήταν τελικά σύντομος. Μέσα σε τρία χρόνια έγινε η δουλειά. Η δική μου θητεία ως Γενικού Διευθυντή δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και μάλιστα σεβόμαστε την ημερομηνία, τηρούμε την ημερομηνία του 17. Είναι αλήθεια, δεν τα καταφέραμε για το Σεπτέμβριο του 14, αλλά τα καταφέραμε για τον Μάιο του 15 και η προθεσμία του 17 τηρείται. Γιατί δεν τα καταφέραμε νωρίτερα, δεν ξέρω. Ήταν πολιτική η απόφαση. Όταν εγώ εργαζόμουν με τον Αντιπρόεδρο Ταγιάννη που ξεκίνησε την ομάδα, πιστεύω πως ήταν μια πολύ σημαντική απόφαση, η οποία Στη συνέχεια στηρίχθηκε από όλα τα κρατημέλη, τους, υπουργού, τους υπουργούς, τους ε, διευθυντές των αυτοκινητοβιομηχανιών κτλ. κτλ. Και έτσι και πέρασε. Το να έχουμε λοιπόν ε, συνενετική, ε, ανοιχτή, καθολική διαδικασία που συμμετέχουν η πολιτική συνιστόσα, η βιομηχανική συνιστότα, όλοι οι φορείς, οι ΟΚΕ, οι περιφέρειες κτλ. Όλα αυτά συνέβαλαν στην υλοποίηση. Ευχαριστώ. Κύριος Ντάνς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καϊέχα, μας δώσατε κάποια στοιχεία για κάποιους πρόρους θανάτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το επαναλαμβάνετε, σας παρακαλώ. 400.000. Α, μου φάνηκε ότι άκουσα 300. Ε, όχι, δεν είναι καλά τα αγγλικά μου γι' αυτό. Και είπα 70.000 σχετιζόμενες με τις μεταφορές. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Αλλά αυτά είναι μόνο τα ε, στοιχεία θανάτων από μικροσωματίδια, όχι από οξύδια του αζότου. Και είπατε ότι θα πρέπει να γίνει και μια περαιτέρω προσπάθεια, γιατί για τα διζελοκίνητα αυτοκίνητα δεν αντιμετωπίζουμε όπως πρέπει τα ζητήματα των εκπομπών μικροσωματιδίων όπως θα έπρεπε. Μάλιστα. Επίσης, είπατε ότι υπάρχουν προβλήματα προς την ερμηνεία της υπέρβασης κύκλου και της ε, συσκευής ε, αναστολής ε, και ότι αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αλλά δεν θα πρέπει να έχετε επαφέ με τα κράτη-μέλη. Και επαφέ με τα κράτη-μέλη χωρί στοιχεία αυτά δεν μπορείτε να έχετε βεβαίω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνο εξωτερικά στοιχεία μπορεί να συλλέξει. Αυτά τα οποία υποπίπτουν στην αντίληψή τη ότι κάτι πάει στραβά. Και αν γυρίσουμε πάλι στα email που έγινε λόγος νωρίτερα, από το 2002, 2010, 2012 και σε σχέση βέβαια με τα βαρέα οχήματα και το σκάνδαλο των ΗΠΑ. Τίποτα από όλα αυτά που είχε συμβεί μέχρι τότε δεν έκρουσε καμπανάκι κινδύνου για να ασχοληθούν οι υπηρεσίες σας. Και αν ναι, Απάντηση. Βεβαίω έχετε απόλυτο δίκιο σχέση με τι ΗΠΑ. Το λέω αυτό ξεκινώντα. Με κατέπληξε το γεγονό ότι έχουν πολύ πιο αυστηρά δεδομένα για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στι ΗΠΑ από ότι η Ευρώπη. Δεν περίμεθα αυτό ότι θα συνέβαινε αυτό. Είναι πολύ πιο αυστηρή λοιπόν στι ΗΠΑ και παραμένουν ακόμη δυσκολίε για μα και σε σχέση με τα στοιχεία τη Παγκόσμια Οργάνωση ε, Υγεία. Σε σχέση με τι συσκευέ αναστολή, νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει και πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση και πόσο δύσκολο να διαγνωστεί ότι υπάρχουν. Ακόμη και το Κοινό Κέντρο Ερευνών, το οποίο έχει κάνει καταπληκτική δουλειά για μα και πρέπει να επενέσω την ποιότητα και τι ικανότητε των τεχνικών του και πραγματογνωμών του, ε, μα έλεγαν ότι είναι αδύνατο ουσιαστικά να διαγνωστεί ότι υπάρχει η συσκευή αναστολή. Γιατί εξ ορισμού αυτή η συσκευή είναι ένα μηχάνημα ή ένα τρόπο που χρησιμοποιείται εσκεμμένα για να αλλάξει τη συμπεριφορά ενό οχήματο. Ε, ναι, αλλά και η υπέρβαση κύκλου θα μπορούσε να είναι μια λύση. Μα υπόθηκε νωρίτερα ότι ε, διάκριση σαφή δεν μπορεί να γίνει, ότι δηλαδή δεν μπορεί να γίνει ακριβώς διάκριση μεταξύ της υπέρβασης κύκλου ή της χρήσης συσκευή αναστολή. Άρα, και επειδή δεν είναι κάτι το απτό, δεν είναι δηλαδή ένα μηχάνημα, πάντοτε υλικό δηλαδή το οποίο μπορεί να διαγνωστεί. Ακριβώς και γι' αυτό δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχερός να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Εγώ έχω 30 υπαλλήλους οι οποίοι διαπραγματεύονται και για τη συμφωνία. Ναι, πολύ καλή δουλειά κάνουν για το FDA, αλλά μια και τελειώνει ο χρόνος μας. Ω, με συγχωρείτε. Από τις πληροφορίες που έχετε συλλέξει από τα email αυτά, σταμάτησαν στο γραφείο σας ή δεν έφτασαν σε σας ποτέ. Ναι, μα υπάρχει μια σειρά από email που λέει «Α, να κοιτάξτε τι συμβαίνει στον έξω κόσμο», υπάρχει κάποια, κάποιο είδος ε, μνήμης. Είναι τα email μεταξύ του Κοινοκέντρου ε, Ερευνών και του Μελετών και της Γενικής Διεύθυνσης για την Ανάπτυξη της Enterprise. Ναι, δεν είχα υπόψη όμω αυτά τα email. Νομίζω ότι πέραν κάποιε ανταλλαγέ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να έχουμε πιο απτά στοιχεία, να γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Δεν μπορούσαμε να έχουμε έτσι τα στοιχεία αυτά. Μα ακριβώ εκεί έγκυται και το ζήτημα, έτσι δεν είναι, λέει ο κ. Στάντ, αφού δεν μπορούσατε να ξεκινήσετε τι έρευνε σα πριν να λάβετε κάποιε πληροφορίε. Δουλειά τη Επιτροπή και το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει η Επιτροπή εν προκειμένου, τη στηρίζει ακριβώ την ενημέρωση από τα κράτη-μέλη, εάν λάβετε κάποια πληροφορία, να αναλάβετε δράση. Εδώ αυτό που μου λέτε είναι ότι δεν έφτασε ποτέ στα χέρια σας αυτή η πληροφορία. Άρα πρέπει να διαρευνηθεί το γιατί δεν έγινε τίποτε. Γιατί ήταν η μόνη πηγή για να ξεκινήσετε τις έρευνες και τις συλλογές στοιχείων. Απάντηση, κοιτάξτε κατά την θητεία μου. Υπενθυμίζαμε με ιδιαίτερη έμφαση τα κράτη-μέλη τις υποχρεώσεις τους, ε, τις ευθύνες τους με επιστολές σε διάφορες χώρες, τους καλούσαμε να δείχνουν επαγρύπνηση για την εποπτεία της αγοράς, ότι τηρούνται οι προδιαγραφές για το περιβάλλον. Επίσης τα κράτη-μέλη έχουν και την αστυνόμευση και την επιβολή και όλα αυτά. Και είναι πολύ σημαντικό να τηρείται η αρχή της επικουρικότητας. Έχουμε ένα αριθμιστικό πλαίσιο. Τα κράτη-μέλη έχουν την ευθύνη της εποπτείας, ε, αν αρχίζουμε να ανακατεύουμε ρόλους κτλ. Όχι, όχι, μα το θέμα είναι ότι ένα πράγμα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήταν να ξεκινήσει μια έρευνα. Αφού είχατε στοιχεία που έλεγαν ότι κάτι συμβαίνει, γιατί δεν κάνατε ποτέ την έρευνα. Εσείς μου λέτε ότι δεν λάβατε γνώση ποτέ. Πολύ καλά. Αλλά γιατί δεν λάβατε γνώση δεν μου λέτε. Καλιέχα. Κοιτάξτε, όταν εγώ πια στα χέρια μου στοιχεία ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ανέφερα την ε, υπόθεση Daimler, αναλάβαμε αμέσω δράση. Δεν είχαμε κανένα λόγο να λάβουμε δράση στη μία περίπτωση και όχι στην άλλη. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτό ο σωστό τρόπο να εξετάζετε το ζήτημα. Δεν είναι η υποχρέωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά των κρατών μελών που επιβάλλουν, που έχουν καθήκον να επιβάλλουν το δίκαιο. Έχω 29 προσφυγές επί παραβάση κατά κρατών μελών. Ούτε είναι και αυτό βέβαια λύση να ξεκινούμε μακροχρόνιες ε, διαδικασίες προσφυγής. Πρέπει να τηρούνται οι ε, διατάξει τη νομοθεσία από το κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας και τι απαντήσει μέχρι τώρα για την εποπτεία στην αγορά, γιατί έχουμε δει μια επιστολή του Επιτρόπου Ταγιάννη, ο οποίο ύστερα από μια άτυπη συνεδρία απευθυνόμενο από την Μέλη έλεγε ότι έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εποπτεία τη αγορά και θυμάμαι αυτή την επιστολή πολύ καλά. Και μάλιστα θυμάμαι πίσω ο ίδιο ο Επίτροπο μου είχε επισημάνει πω την επιστολή αυτή τη συνέταξε κατόπιν μια ε, μιας εισαγωγή ελαστικών από την Κίνα. Άρα πάλι δεν ήταν θέμα εκπομπών. Η επιστολή, λέει ο κ. Καγιέχα, ήταν μια υπενθύμηση προς τις χώρες ότι πρέπει να τηρείται η νομοθεσία. 25 Ιουλίου του 2012 απεστάλησε 28 κράτη-μέλη και δηλώνει, παραθέτω, τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν τις απαραίτητες δομές και πόρους στη διάθεσή τους για να εντοπίζουν στην επικράτειά τους και να αναλαμβάνουν διορθωτική δράση σε περίπτωση όπου τα προϊόντα δεν τηρούν τις προδιαγραφές έγκρισης Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σημαίνουν σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών και το περιβάλλον και επί παραδείγματι η παραποίηση ή ε, τροποποίηση αυτών των προϊόντων. Μια ε, γενική υπενθύμανση και σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Ντάντς, ακόμη και ελλείψη στοιχείων αποδεικνύεται ότι εμείς δεν δηλιάζαμε και υπενθυμίζαμε στα κράτη-μέλη ποιες είναι οι ευθύνες τους. Μάλιστα, δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά τα λόγια σας, μας λέτε ότι τα κράτη-μέλη είχαν τις ευθύνες και αυτά έπρεπε να ανταποκριθούν στα όσα τους έλεγε η Επιτροπή ΜΕΝ, αλλά η Επιτροπή δεν είχε καθήκον να ε, λάβει δράση με βάση τα email που του επεστάλησαν. Όχι εμεί υπενθυμίσαμε στα κράτη-μέλη τα καθήκοντά του. Ο κανονισμό του δίνει ε, εντολή και εξουσίε να αναλάβουν δράση. Μια επιστολή από την GRC δεν δίνει εντολή ή εξουσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διερεύνηση. Εμεί δεν έχουμε τέτοια εντολή. Μπορούμε να ζητήσουμε από τη χώρα που εμπλέκεται, εάν τυχόν, ε, για να ρωτήσουμε αν έχει τηρήσει τη σχετική νομοθεσία. Αυτό είναι το σύστημά μα και είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε το νόμο. Όπω είπε και ο κύριο Φάλκεμπεργκ. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, να βελτιώσουμε το σύστημα, να βελτιώσουμε την εποπτεία της αγοράς, να κάνουμε αυτά τα πράγματα καλύτερα. Και ύστερα από το σκάνδαλο Volkswagen, που είναι και ο στόχος αυτής της ε, έγκρισης τύπου Πρέπει να κάνουμε το σύστημα πιο αποτελεσματικό και σε αυτό έκλεισα την τοποθέτησή μου, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρξει γενικότερη διακυβέρνηση του συστήματος και εποπτεία. Στην προηγούμενη μου θέση στις μεταφορές ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχα τη σχετική ευθύνη τα αυτοκίνητα, άλλωστε είναι ο μόνος τρόπος μεταφορών για τα οποία δεν έχουμε εποπτεύουσα αρχή. Υπάρχει για τις θαλάσσιες μεταφορές. Ναι, με την Ευρωπαϊκή Αρχή ε, θαλασσίων μεταφορών κατόπιν του σκανδάλου Έρικα. Έχουμε για τι αεροπορικέ μεταφορέ, για τι αεροδρομικέ μεταφορέ. Αλλά για τα οχήματα, για τα αυτοκίνητα δεν έχουμε εποπτεία τη αγορά. Αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε για να ενισχυθεί και πρέπει για να συνδυάσω και αυτό που λέγατε εσείς, να υπάρξει εποπτεία και της δράσεως των αρχών, των εθνικών αρχών, αλλά και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ναι, αλλά για να συνεχίσω πριν εξαντληθεί ο χρόνος μου, αναφερθήκατε στην ερώτηση 1 σε πιθανό, πιθανές δράσεις που θα μπορούσαν να αναλάβουν τα κράτη-μέλη με κίνητρα και ε, περιορισμό ή απαγόρευση εισόδου στις, στα κέντρα των πόλεων, φορολογικά κίνητρα και το καθεξής. Ήταν αυτά μια, κάποιες από τις λύσεις που παρουσιάζατε εσείς στα κράτη-μέλη όσο ήταν ε, στη θέση αυτή πριν να ξεσπάσει το σκάνδαλο Volkswagen να επιτρέψετε μου να διευκρινίσω την, την επιστολή αυτή την απέστειλα στην, ε, από τη θέση μου την τωρινή, δηλαδή Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης για το Περιβάλλον. Γιατί το έκανα αυτό γιατί κατάλαβα ότι δεν έχουμε επαρκείς δυνατότητες δράσης και άρα μία από τις προσεγγίσεις που θα να έχουμε, γιατί αυτό ξεκινάει από τις πόλεις, θα ήταν αυτή η λύση. Οι ευρωπαϊκές πόλεις αναλαμβάνουν δράση, περιορίζοντας την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, με ζητήματα που έχουν να κάνουν όλο και περισσότερο με φορολογικά κίνητρα ή αντικίνητρα. Τεχνολογία που μπορεί επίσης να βοηθήσει τα, ηλεκτρονικά, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και την, και την καινοτομία γενικά. Μια σειρά από μέτρα λοιπόν που μπορούν να αξιοποιηθούν όλα αυτά αλλά και άλλα μέτρα τα κατέγραψα σε μια επιστολή που πολύ ευχαριστώ μπορώ να σας ε, διαβιβάσω από την απέστειλα στα 28 κράτη-μέλη για να συζητήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξεπεράσουμε το τεχνικό ζήτημα της έγκρισης τύπου ή των δοκιμών και να κοιτάξουμε με μια πιο γενική προσέγγιση το ζήτημα. Κύριος Λόπες Βερμέχο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καγιέχα, στις απαντήσεις σας φαίνεται με μεγάλη σαφήνεια ότι εσείς γνωρίζατε πως οι πραγματικές εκπομπές δεν αντιστοιχούσαν με τις μετρήσεις στη διάρκεια δοκιμών, ότι αυτές οι αποκλήσεις ήταν γνωστές από διάφορες υπηρεσίες της Κομισιόν και μάλιστα υψηλού επίπεδου συμπεριλαμβανομένων ε, πολιτικών διαλόγων και με τον Επίτροπο κ. Ταγιάννη. Επίσης ε, είχατε θίξει το θέμα και στις αυτοκινητοβιομηχανίες, στους κατασκευαστές και φαίνεται πως αυτό ήταν απολύτως νόμιμο. Εγώ, εμένα μου φαίνεται αυτό ότι είναι το πιο σκανδαλώδες από όλα, γιατί ή υποψιαζόσασταν ότι οι κατασκευαστές χρησιμοποιούσαν τις συσκευές αναστολή, πράγμα το οποίο αρνήθηκαν ε, ε, συστηματικά, ή υποψιάζεσταν ότι τα κράτη-μέλη δεν χρησιμοποιούσαν, δεν εφήρμοζαν σωστά τα δοκιμές για τις εκπομπές. Πάντως αυτό που προκύπτει χωρίς αμφιβολία σημαίνει ότι αυτέ οι παραβάσεις συνέβαιναν ταυτόχρονα και εσεί δεν ενεργήσατε όταν έπρεπε να το έχετε κάνει. Έχω τρεις ερωτήσεις ε, να σας τι υποβάλω όλες μαζί για να κερδίσουμε χρόνο. Δεν θυμάστε σε καμία περίπτωση να συζητήσατε για συσκευέ αναστολή, ε, εφόσον ήταν γνωστέ από όλου του συνομοθέτε ε, όλων των χωρών. Δεν θυμάστε καμία περίπτωση όπου κάποια υπηρεσία έθεσε τη δυνατό... την πιθανότητα οι διαφορέ ανάμεσα στι πραγματικέ και τι καταγεγραμμένε ε, εκπομπέ για ορισμένα μοντέλα, αδιαφορέ και αποκλήσει που εσεί γνωρίζετε μπορεί να οφείλονταν σε παράνομου μηχανισμού. Πραγματικά θα ήταν από τις πρώτες δυνατότητες που θα είχατε ε, και θα έπρεπε να το έχετε σκεφτείτε από τη, σκεφτεί από τη στιγμή που καταλάβατε ότι υπήρχαν τέτοιες ε, αποκλήσεις. Και τέλος, τελευταία από τις τρεις ερωτήσεις. Εσείς ε, ε ξερούσατε τις κατασκευαστικές εταιρείες με, από οποιαδήποτε τέτοια διαφορά και γιατί δεν υποψιαστήκατε πως οι εθνικές αρχές εφήρμοζαν την ευρωπαϊκή νομοθεσία λάθος επιτρέποντας αυτές ε, τις συσκευές. Και εσείς κάνατε συζήτηση με τις εθνικές αρχές ε, πότε, που και σε ποιο επίπεδο αποφασίστηκε να μην ξεκινήσει καμία διαδικασία έρευνας ε, ή παραβάση. Πραγματικά μου φαίνεται κατανόητο να μην το γνωρίζατε. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, όχι μόνο το γνωρίζαμε. Όλοι γνωρίζαμε πως υπήρχαν διαφορές, ξεκινώντα με αυτό και το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο το γνώριζε. Το Συμβούλιο το γνώριζε, τα κάτι μέλη το γνώριζαν. Σας παρέθεσα τι έλεγαν ε, οι ο Καν 40 που είχε μετρήσει ε, πως υπήρχαν μάλλον διαφορές ανάμεσα στις πραγματικές και τις ε, εκπομπές και τις εκπομπές εργαστηρίων. Το γνωρίζαμε όλοι. Το γνω... Ήταν ε, κοινή γνώση. Αυτή το γνώριζαν και οι προβουλευτές. Αυτό που έγινε είναι ότι όλοι πιστεύαμε πως η το αίτιο οφειλόταν σε αυτό το τεστ, το New European Driving Cycle, εκείνο το NEDC, που δεν ήταν αρκετά αντιπροσωπευτικό. Αυτό το, το τεστ θεωρήθηκε λάθος και γι' αυτό το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε το 2013, το Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνισμού, η Κομισιόν, το GRC και όλοι οι θεσμοί είπαν πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Κομισιόν κάνε μας ένα νέο ε, σύστημα που να λειτουργεί. Η λύση ήταν να φτιαχτεί ένα νέο σύστημα το οποίο να λειτουργεί και να μετράει τις εκπομπές σε πραγματικό χρόνο. Κανείς ποτέ δεν μας είπε ότι υπήρχαν τέτοιες συσκευές αναστολής. Είχαμε εκατοντάδες συσκέψεις, συνεδριάσεις με ένα ζωρό επιτροπές, ομάδες κτλ. Κανείς δεν έκανε λόγο για τέτοιες συσκευές αναστολής. Αυτή, έτσι έχει η κατάσταση. Και τέλος, στις σχέσεις μας με τα κράτη-μέλη δεν, ε, δεν δείχνουμε κακή πίστη ποτέ. Ε, οφείλουμε να συνεργαστούμε, αλλά δεν έχουμε κακή πίστη. Εάν υπάρξουν αποδείξεις, μαρτυρίες, ναι, τότε ναι. Αλλά εγώ δεν ξεκινώ ε, θεωρώντας ε, ότι είναι κανείς κακόπιστος. Όχι. Δεν πιστεύω ότι υπήρχε κακή πίστη από πλευρά των κρατών μελών. Ευχαριστώ η κυρία Ντέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας κύριε Καλέχα. Κάτι το φοβερό που είπατε ήταν ότι όλοι το γνώριζαν και κάνει δεν έκανε τίποτα. Και λέτε ότι ε, θα έπρεπε τώρα να βρούμε νέα εργαλεία. Μιλήσατε για ένα εργαλειάκι που είναι σημαντικό και το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε στις διάφορες επιτροπές. Μιλήσατε για το γεγονός ότι πρέπει πλέον να δημιουργηθεί αυτός ο ευρωπαϊκός οργανισμός που να είναι πραγματικά ανεξάρτητος. Ανεξάρτητος για την υποπτήρα των αγορών και για την έγκριση τύπου των οχημάτων. Εσείς λοιπόν τι πιστεύετε, τι θα κάνετε για να μας βοηθήσετε κύριε Καλέχα για να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Η ερώτηση 7. Είστε ένας εκ των πρώτων που είπατε ότι θα πρέπει να γίνει ένας απολογισμός κόστους ωφέλειας πριν από κάθε νομοθετική πράξη σχέδιο. το γεγονό ότι 75.000 άνθρωποι πεθαίνουν πρόωρα ετησίω στην Ευρώπη λόγω των εκπομπών οξυδίων του αζότου, αυτή η απόφαση λήφθη όταν η Επιτροπή αυτή η Επιτροπολογία, εν πάση περιπτώσει, τον Οκτώβριο του 2015 αποφάσισε ότι θα συστήσει νέα νομοθεσία, θα συντάξει νέα νομοθεσία, ένα νέο παράγοντα συμμόρφωση που θα πει στου κατασκευαστέ αυτοκινήτων μη σέβεστε του τύπου. Τα όρια μπορείτε να τα ξεπερνάτε κατά 110% μέχρι το 2020 και μετά κατά 60%. Αυτό το στοιχείο αναφέρθηκε. Δεύτερο, τρίτο μάλλον που θέλω να σας ρωτήσω είναι λέτε ότι η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται παρά μόνο σε περιπτώσεις σε που φτάνει σε βαθμό που έχει αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία. Το τροποποιείτε, το τροποποιείτε πώς προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ντέλη και εδώ θέλω να κάνω μια σύντομη διευκρίνηση για την αρχή των όσων είπατε. Είπατε ότι κανέ, όλοι το ξέρανε και δεν έκανε κανείς τίποτα. Όχι, εγώ πιστεύω ότι κάναμε πολλά. Και αυτό που προσπάθησα να σας εξηγήσω είναι οι προτάσεις μας για την αλλαγή του συστήματος, είναι η τεχνική εργασία του GRC, είναι όλες οι διαφορετικές νομοθετικές πράξεις τις οποίες προτείναμε για να μετατραπούν οι παλιές δοκιμές στο RTE και είναι και η μεταρρύθμιση του έγκριση τύπου. Δεν είναι δίκαιο να λέτε λοιπόν ότι κανεί δεν έκανε τίποτα. Η Κομισιόν έκανε πολλά νομίζω και στηρίχθηκε από τα κρατημέλη, από το από του θεσμού. Ποια είναι η γνώμη μου για μια ανεξάρτητη υπηρεσία, έναν ανεξάρτητο οργανισμό. Εγώ είμαι υπάλληλο τη Επιτροπή και ακολουθώ τι αποφάσει των Επιτρόπων και θα ήθελα να απαντήσω ω εξή. Πιστεύω πω χρειάζεται ένα μηχανισμό εποπτεία ισχυρότερο που θα μας επιτρέπει καλύτερα να επιβλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο ε, εφαρμόζουν ε, τη νομοθεσία οι εθνικές αρχές και για τους οικονομικούς φορείς επίσης. Έθεσα το παράδειγμα της ε, αεροπλοείας. Ο Οργανισμός Ασφάλειας Αεροπλοείας στην Κολονία έχει τη δυνατότητα να εποπτεύει τις δράσεις. Όταν ήμουν διευθυντής της πολιτικής αεροπορίας γίνονταν επιθεωρήσεις στις εθνικές αρχές για να ε, δουν τη λειτουργία. Υπάρχουν νομοθεσίες. Μετά από την 11η Σεπτεμβρίου την επαύριο η Κομισιόν έλαβε την εντολή για κοινοτικοποίηση της ασφάλειας αεροπλοείας. Πράγμα το οποίο έγινε εντός ενός μήνα Υπάρχει μια ομάδα εποπτών επιθεωρητών στην DG Move που ελέγχει τα αεροδρόμια για να επαληθεύει τις, ε, την εφαρμογή των διατάξεων ασφάλειας. Αλλά Χωρί χωρίς να πάμε σαν εξάρτητο οργανισμό, γιατί δεν πιστεύω ότι αυτή ήταν η απόφαση των επιτρόπων, αλλά να μεταρρυθμιστεί το σύστημα εποπτείας των αγορών, όπω προτάθηκε. Και αυτό είναι υποσυζήτηση τώρα στο Κοινοβούλιο. Θέσπιση τη δυνατότητα ε, ε, ελέγχων, ενίσχυση τη ανεξαρτησία των εθνικών αρχών, εναρμόνιση τη επιβολή, τη διευκόλυνση της Κομισιόν ώστε να μπορεί άμεσα να προβαίνει σε ελέγχους και να επιβάλλει κυρώσεις. Ήδη αυτά είναι πολλά και αυτά είναι μέσα στην πρόταση τη Κομισιόν. Συγκεκριμένα μέτρα που είναι επιτάπητο. Εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση μπορούμε να βελτιώσουμε το σύστημα. Ανάλυση κόστους ωφέλεια. Είπατε, ναι, να, απαντήσω, έχετε άλλε δύο ερωτήσει Το έχουμε κάνει. Στην απόφαση του Οκτωβρίου 2015 το κάναμε. Η παράγοντες τη συμμόρφωση τη Κομισιόν δεν εγκρίθηκαν, δυστυχώς, όμως είναι πολύ καλύτερα να υπάρχει αυτή η απόφαση από το να μην υπάρχει τίποτα, να είμαστε στο αδιέξοδο, γιατί έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε στο Real Driving Emissions. Για την οδηγία περί περιβαλλοντικής ευθύνης υπάρχει Γίνεται έλεγχο αυτή τη στιγμή μάλιστα και θα δούμε πώς μπορούμε να το επεκτείνουμε και για άλλε. Βλέπετε ότι υπάρχει αντίφαση εδώ και το κλείνομαι έτσι. Ε, ε, ο, άνθρωπο, ο αριθμός των ανθρώπων που πεθαίνουν λόγω των ε, οξυδίων του αζότου εκρήγνεται, αλλά ε, όμως πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαβουλευθεί, να εγκρίνει. Ναι, μα δεν το εγκρίνει η Κομισιόν, το Συμβούλιο το εγκρίνει, τα κράτη-μέλη. Έληξε ο χρόνος σας τώρα. Παρακαλώ, εσείς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και καλησπέρα σας. Κύριε Καγιέχα, για, τις, ε, για τη χρηματοδότηση που έχει χορηγηθεί στην αυτοκίνητο βιομηχανία. Το άρθρο 12 του κανονισμού 715 με ενδιαφέρει. Εφόσον λοιπόν αυτά τα οχήματα με δίζελ που κυκλοφορούν στην αγορά ξεπερνούν κατά έξι φορές κατά μεσόωρο, τα επιτρεπόμενα όρια και υπάρχει πλέον σαφώς απόδειξη ότι δεν έχουν τηρηθεί τα όρια και ότι υπάρχει μεγάλη απόκληση μεταξύ αυτών που καταγράφονται σε εργαστηριακές δοκιμές και της πραγματικής οδήγησης. Ε, τι πιστεύετε σε σχέση με την χρηματοδότηση που έχει χορηγηθεί ε, στην αυτοκινητοβιομηχανία και αναφέρομαι πάντα στο άρθρο αυτό που ανέφερα νωρίτερα από τον κανονισμό 715. Είναι παράνομη αυτή η χρηματοδότηση ή όχι. Ή εν πάση περιπτώσει τι έχει κάνει η Επιτροπή για να παρακολουθήσει αυτή τη χρηματοδότηση. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Είναι όντως πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση, γιατί όντως το άρθρο 12 του κανονισμού επιτρέπει τα κράτη-μέλη να ε, δημιουργήσουν οικονομικά κίνητρα έτσι ώστε οι κατασκευαστές που προσαρμόζονται στην νομοθεσία να επιβραβευθούν, ώστε να έχουμε αυτοκίνητα που ρηπαίνουν λιγότερο στην αγορά. Αυτά τα κίνητρα θα πρέπει να είναι υποαίρεση τη στήριξη των ορίων που, ορίζονται μέσα στην ε, νομοθεσία, στο πλαίσιο της νομοθεσίας και επίσης συνδέεται με το γεγονός ότι τα ρηπογόνα οχήματα θα μπορούσαν να αποσυρθούν ή μάλλον να αναπροσαρμοστούν ε, είτε απόσυρση είτε μετατροπή ώστε να τηρούν τα όρια. Αυτά τα κίνητρα λοιπόν που δόθηκαν Σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις, όταν γίνεται μια αλλαγή πρέπει να κοινοποιείται στην Κομισιόν ώστε να επαληθεύουμε και εμείς ότι είναι σύμμορφη προς την οδηγία περί κρατικών αυτό το θέμα δεν ετέθη για τους κατασκευαστές. Υπάρχουν όμως κάποιες υποθέσεις όπου οι κατασκευαστές που είχαν κάποια προβλήματα ζητούν περιφερειακά κονδύλια και για την ώρα η Κομισιόν προσπαθεί να ελέγξει εάν όντως αυτά συνάδουν με την εφαρμογή της οδηγίας αυτής. Όμως είναι κάτι που ακόμα το επαληθεύουμε για να δούμε αν έχουμε συγκεκριμένα ε, παραδείγματα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Είναι ανησυχητικό να σκέφτεται κανείς ότι αυτές οι επιδοτήσεις μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν αδιακρίτως και όχι πραγματικά, ώστε να έχουμε καθαρά αυτοκίνητα στους δρόμους. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση σε σχέση με τον ε, κύκλο δοκιμών, το Common Artemis Driving Cycle. Ήθελα να γνωρίζω αν εσείς ε, έχετε υπόψη σε αυτή τη διαδικασία, γιατί συχνά άλλοι ε, προσκεκλημένοι μας και από πλευρά της Κομισιόν φάνηκε να μην γνώριζαν καν ότι υπάρχει αυτός ο κύκλος δοκιμών που ε, μάλιστα υπήρχε ήδη από τότε που ήταν υπό επεξεργασία ο κανονισμός 715 δηλαδή θα μπορούσε να έχει θεωρηθεί έγκυρη εναλλακτική στο δοκιμή NED e NEDC. Δεν έγινε ωστόσο αυτό και εγώ όπως ανακάλυψα αυτό αυτό ο κύκλο δοκιμή χρησιμοποιείται και από του ίδιου τους κατασκευαστές αυτοκινήτων για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν σε με υπορεαλιστικές συνθήκε στο σχεδιασμό αλλά και στον παραγωγή τις εκπομπές των αυτοκινήτων. Γιατί δεν διαλέξατε αυτή την εναλλακτική λοιπόν. Σα ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι αναφέρεστε στη φάση της έγκρισης αυτού του κανονισμού του 715, όπου εγώ δεν ήμουν υπεύθυνο για αυτό το θέμα. Αυτό εγκρίθηκε το 2012. Αυτά τα θέματα σε σχέση με τις διάφορες, ε, τους διάφορα είδη μέτρηση αποτέλεσε αντικείμενο ανάλυσης και μελέτης από το Κοινό Κέντρο Μελετών, το GRC, που επιμένω έχει, έχει παίξει μάλλον σημαντικό ρόλο σε αυτέ τι εργασίε, για να μετρήσει σε ποιο βαθμό α, αυτά, τα, αυτές οι δοκιμές είναι πιο κατάλληλες και αν απαντούν στα προβλήματα που έχουμε. Αφού λοιπόν ανέλησαν όλες τις ε, διαδικασίες και αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν διάφορες επιλογές, το GRC μάλιστα σε κάποια φάση εξέτασε τέσσερις διαφορετικούς κύκλους των ισχύοντα, τους τυχαίους κύκλους, τα διάφορα μοντέλα εκπομπών και τελικά τα φορητά συστήματα μέτρησης εκπομπών, που θεωρήθηκε τελικά το πιο πολλά υποσχόμενο σύστημα που εξασφάλιζε ότι οι εκπομπές σε πραγματικό χρόνο, σε πραγματικές συνθήκες μάλλον, αντιστοιχούσαν με τα όρια που θέσπιζε η κοινοτική νομοθεσία. Αποβεύγοντας τις ε, σημερινές παρεκκλησίες να γνωρίζω ωστόσο ότι δεν είμαι εμπειρογνώμονας ε, για το κύκλο Άρτεμις. Ξέρω πως αναφέρθηκε ως δυνατότητα, αλλά δεν επελέγει τελικά. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ ολοκληρώνουμε τον πρώτο γύρο των ερωτήσεων. Α, δεν τελειώσατε, δεν τελειώσατε. Έχετε και δεύτερος γύρος ερωτήσεων. Εδώ πια όμως θα έχουμε ε, χρόνο τριών λεπτών. Ο κύριος Γκίζικε, μαθαίνω ότι έχετε προσκαλέσει και μια ομάδα επισκεπτών από την Κάτω Σαξονία που είναι η εκλογική σας περιφέρεια. Τους απευθύνω το καλώς ορίσατε, θα σας παρακολουθήσουν να εργάζεστε. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην ειδική εξεταστική επιτροπή για τις μετρήσεις στον ε, ε τομέα των αυτοκινήτων. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και σας κύριε Καγιέχα που είστε παρόν σήμερα για να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Χαίρομαι πολύ βεβαίως για την παρουσία ομάδος επισκεπτών της εκλογικής μου περιφέρειας. Είμαστε απόλυτα διαφανές σώμα. Οι φίλοι και οι φίλοι μου από την Κάτω Σαξονία έφτασαν μέχρι εδώ για να μας παρακολουθήσουν. Πολύ συγκεκριμένα είπατε στην εισαγωγή σας ότι υπάρχουν 400.000 πρώιμοι θάνατοι και 70.000 από τα οξύδια του αζότου. Η κυρία Νταλή έφτασε στις 75.000. Φαίνεται πως προσθέθηκαν λοιπόν μερικές χιλιάδες ακόμη την τελευταία μισή ώρα. Νομίζω ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Θα πρέπει να εμείνει κανείς στα γεγονότα και όχι να λέει ότι οι αριθμοί εκρήγνεται, αλλά οι αριθμοί αυτοί είναι ε, αποτέλεσμα της ιδίας φαντασίας. Θα τις τα πω και μετά γιατί βλέπω τώρα έχει φύγει. Τη συζήτηση αυτή κάναμε και με τον κύριο Φάλκενπεκ. Χρειαζόμαστε ξεκάθαρη νομοθεσία. Χρειαζόμαστε ενιαία επιβολή της νομοθεσίας αυτής σε όλες τις Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Προ δύο εβδομάδων είχαμε εδώ τον κύριο Ντομπριντ, τον Υπουργό ε, Μεταφορών της Ομοσπονδιακής Γερμανίας, όπου λέει ότι σε ένα μοντέλο της Fiat το τεστ ε, ε, κράτησε 22 λεπτά και εφόσον αυτό εκεί χρησιμοποιεί μια διάταξη αναστολής ε, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα. Εδώ όμως είναι αντιφατικά τα ευρήματα. Αυτό που είπατε μόλις, ο οργανισμός, η πλατφόρμα, η συγκεντρωτική, κεντρική θέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό δεν είναι κρίσιμο. Το κρίσιμο θα είναι οι αρμοδιότητες που θα έχει η μονάδα αυτή. Άρα, τι χρειάζεται ο Γερμανός ε, Μεταφορών μίλησε για, μια, ε, για ένα οργανισμό συμψηφισμού. Εσείς τι ιδέα έχετε για μια πραγματική αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς. Ο κ. Καγέχα, ευχαριστώ αγαπητέ κύριε Κίσικε και ευχαριστώ και τους άξονες φίλους σας που είναι ε, σήμερα εδώ. Είπατε δύο σημαντικά πράγματα. Πρώτο, Χρειαζόμαστε ξεκάθαρη νομοθεσία. Όσο γίνεται πιο ξεκάθαρη νομοθεσία. Διότι είμαστε μια μεγάλη κοινότητα με διαφορετικέ γλώσσε και διαφορετικέ νομικέ παραδόσει κτλ. Άρα η νομοθεσία που εγκρίνουν τα δύο συνομοθετικά όργανα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και να μπορεί να εφαρμόζεται σε όλε τι δικαιοδοσίε. Για τις ε, εκπομπές των αυτοκινήτων πιστεύετε πως οι διαφορές, ε, θα πρέπει να καταλάβετε ότι οι κλιματολογικές διαφορές και οι γεωγραφικές διαφορές που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα στη Σαξονία, στη Φιλανδία, την Ανδαλουσία, διότι και εξής επηρεάζει το πώς συμπεριφέρεται το κάθε αυτοκίνητο. Είναι πάρα πολύ σημαντική λοιπόν η σαφήνεια της νομοθεσία. Δεύτερον, χρειαζόμαστε ομοιόμορφη εφαρμογή. Έχουμε μια αγορά. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε να υπάρχουν ε, διαφορές στην εφαρμογή των νομοθεσιών και τα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται σε μια χώρα να υπόκειται σε διαφορετικές διαδικασίες έγκρισης από ότι σε άλλες χώρες που υπήρχαν, δηλαδή πιο εύκολες ή λιγότερο απαιτητικέ από ό,τι άλλο. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε αυτόν τον κανονισμό για να θεσπίζουμε ότι ένα ένα αυτοκίνητο που έχει εγκριθεί στη μία χώρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο και στις υπόλοιπες. Είναι αλήθεια ότι αυτή η διαφορά ε, στις, ε, ε, στη συμπεριφορά επηρεάζει. Εσείς αναφερθήκατε στην υπόθεση της Fiat. Εξετάζουμε αυτή τη στιγμή το αίτημα της Γερμανίας και της Ιταλίας για να δοθεί αποσαφήνιση σε αυτή την υπόθεση. Και είναι σημαντικό, όπως είπατε, να έχουμε αυτή την εμπειρία. Ε, ε, πρέπει να στηριχθούμε σε εθνικές αρχές ε, έγκρισης, γι' αυτό πρέπει να συνεργαζόμαστε στην τα γι' αυτό δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι κακόπιστα, πρέπει να εργαζόμαστε, α, συνεργαζόμαστε αγαστά όπως απαιτεί και η συνθήκη. Ευχαριστώ, κύριε, ο κύριος Λόπες. Λόπες. Είπατε ότι ανταλλάσσετε πληροφορίες για την ε, λειτουργία των ε, δοκιμών και ότι δεν γνωρίζετε τα συσκευέ αναστολή. Όμω πρέπει κάποια πράγματα να ε, διευκρινιστούν. Γιατί στην υπόθεση των ψυκτικών MAC έγινε τέτοια αίτηση αποσαφήνιση και όχι για την υπόθεση Volkswagen. Είναι απλό. Γιατί για την MAC γνωρίζουμε, έχουμε μάλλον ρητή αναγνώριση μιας επιχείρησης που παραβιάζεται ο κοινοτικό δίκαιο και που έθεσε στην αγορά αυτοκίνητα που δεν σέβονταν την ε, κοινοτική νομοθεσία και το αρμόδιο κράτος μέλος δεν ε, έκανε τη δουλειά του. Είχε δώσει ένα παλιό πιστοποιητικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε από αυτή την εταιρεία. Ενώ εδώ για τη Volkswagen, όταν η Αμερικανική Αρχή μας ενημέρωσε ότι υπήρχε παραβίαση της Αμερικανικής νομοθεσίας, ε, ε, προβήκαμε και εμείς σε, σε ενέργειες. Όμως πόσες φορές συζητήθηκε στην Τεχνική Επιτροπή για τα αυτοκίνητα ε, και ε, πόσο καθυστέρηση υπήρξε σε σχέση με την, με την υπόθεση αυτή. Θα σας έδινα αυτές τις πληροφορίες, αλλά αυτό το ντοσχέ για τις καθυστερήσεις είναι στην ατζέντα της Επιτροπής Αυτοκινήτων, το για τα αυτοκίνητα, σε όλες τις ημερήσιες διατάξεις ε, από το 2014, 1η ε, Απριλίου, 15 Οκτωβρίου, 24 Νοεμβρίου και 18 Δεκεμβρίου, κάθε μήνα δηλαδή, μάλιστα τέθη στην ημερήσια διάταξη στις 26 Ιανουαρίου 2015, 24 Μαρτίου 2015 δεν επετεύχθη η δική πλειοψηφία και στις 19 Μαΐου καταφέραμε, του 2015 καταφέραμε να το εγκρίνουμε. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορέσαμε να το εγκρίνουμε νωρίτερα, πάντως μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι σε κάθε κάθε ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων τη Επιτροπή υπήρχε το θέμα. Μάλιστα. Γίναν σεβαστέ όλε οι προθεσμίε που προβλέπονταν σε σχέση με την ανακοίνωση CARS 2020. Ναι, η πιο σημαντική προθεσμία έγινε σεβαστή, τηρήθηκε, ότι δηλαδή θα τεθεί σε ισχύ από το 2017. Δεν μπορέσαμε να τηρήσουμε την προθεσμία του Σεπτεμβρίου του 2014 γιατί δεν υπήρχε ε, ειδική πλειοψηφία εγκρίθηκε, υπήρξε μάλλον η πλειοψηφία το Μάιο του 2015. Είχαμε μία μικρή καθυστέρηση κάποιων μηνών, αλλά χωρίς να επηρεαστεί η τελική προθεσμία για την έναρξη ισχύω που είναι το 2017. Στις, αναφε... στις απαντήσεις σας λέτε για πιθανές ε, πρωτοβουλίες από πλευράς της Κομισιόν για να αποσυρθούν τα ελαττωματικά αυτοκίνητα. Μπορείτε να μας πείτε ε, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή. Εμείς υποβάλαμε αυτή την πρόταση στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της νομοθεσίας για το type approval, για την έγκριση τύπου, για την οποία μιλούσαμε προηγουμένως. Αυτό που προτείνει η Κομισιόν είναι να έχουμε την ε, αρμοδιότητα που τώρα δεν έχουμε, να μπορούμε να επιβάλλουμε κυρώσεις άμεσα τον κατασκευαστή. Αυτό που μου ζήτησαν, ε, με ρώτησαν ορισμένοι βουλευτές γιατί δεν το κάνατε, γιατί απλώς η νομοθεσία αυτή τη στιγμή δεν μας επιτρέπει κάτι τέτοιο και δεύτερον να μπορεί η Κομισιόν να επανέλθει στην, στον νέο προγραμματισμό και στην μεταρρύθμιση. Ξέρω πως εδώ δημιουργούνται πολλά προβλήματα στην Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς και αγωνίζεστε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχυθούν οι, οι αρμοδιότητες εποπτείας της αγοράς. Εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα ξαναγίνουν τέτοια πράγματα ε, λόγω των ε, ε, ελαττωμάτων της ισχύουσας νομοθεσίας. Ευχαριστώ κύριος Γκίζικε. Ο κύριος Γκίζικε λοιπόν. Δεύτερη σειρά ερωτήσεων από εμένα. Έρχομαι στην συζήτηση που διεξάγει τώρα στη Γερμανία σχετικά με το μέλλον του κινητήρα diesel. Στο μεγάλο συνέδριο των Πρασίνων του Σαββατοκυριακού αποφάσισαν από το 2030 και μετά να μην επιτρέπονται πλέον κινητήρες εσωτερικής καύσεως. Προ δύο εβδομάδων είχαμε εδώ από την κάτω σαξονία των Υπουργών Μεταφορών κάτω Σαξονία υπερψήφισε, ενδιαφέρον αυτό, στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο αυτή την πρωτοβουλία. Εδώ πάντως ο υπουργό είχε άλλο ε, ύφος, άλλο τόνο δηλαδή στις ε, ε, παρατηρήσεις του, στι δηλώσει του και είπε ότι δεν το βρίσκει διαρρεαλιστικό αυτό. Εσείς πώς βλέπετε το μέλλον του κινητήρα Diesel στον χρονικό, μέχρι τον χρονικό ορίζοντα 2030. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως η υπόθεση Volkswagen έθεσε επιτάπητος στο μέλλον του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας, στο μέλλον της τεχνολογίας diesel στην Ευρώπη, αντίθετα με το τι συμβαίνει στις ΗΠΑ. Τα αυτοκίνητα diesel είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της αγοράς, είναι το μισό τη αγορά. Στη ΣΥΠΑ είναι 3-4% αν είναι σωστά τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, αλλά πιστεύω πω η αυτοκινητοβιομηχανία ε, στο μέλλον ε, θα προβεί σε τεχνολογικές καινοτομίες. Η χρήση του ηλεκτρισμού είναι απαραίτητη, το υβριδικό αυτοκίνητο, αλλά πιστεύω πως και στην Ευρώπη είναι αλήθεια ότι οι κινητήρες δίζελ έχουν εξελιχθεί για να αντιμετωπίσουν τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Οι εκπομπές ε, του των οξυδίων του αζότου πρέπει επίσης να ελεγχθούν εντάξει να χρησιμοποιηθεί, να συνεχίσει να χρησιμοποιείται το ντίζελ, αλλά να είναι καθαρό, να τηρούνται οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Ε, ναι, στο ντίζελ, αλλά που πρέπει να χρησιμοποιεί την τεχνολογία, την καινοτομία, ώστε να ε, εντάσσεται στο σεβασμό της οδηγίας. Πάντως, ε, κάτι πολύ σημαντικό θέλω να πω, ότι και η Κομισιόν από πλευρά τη πρέπει να κρατά απόλυτη ουδετερότητα στα τεχνολογικά θέματα. Δεν μπορούμε να προωθήσουμε τη τάδε ή τη δίνα τεχνολογία. Οι κατασκευαστέ και οι αρχέ είναι αυτέ που έχουν αυτή την ε, δυνατότητα. Εμεί ε, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ότι όποια και να αποφασιστεί να είναι η τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσουν, θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφέ ασφαλεία και οι περιβαλλοντικέ προδιαγραφέ επίση. Πάλι ο βουλευτή Γκίζικε. Ευχαριστώ. Ούτε εσείς είστε τεχνικός, ε, νομίζω δηλαδή πως δεν είστε, εγώ πάντως δεν είμαι, ούτε ο μηχανικός λοιπόν. Γι' αυτό θα ήθελα να θέσω υπόψη σας κάτι που είπε ο κύριος Ίντρα, Καθηγητή εξέλιξη μηχανών, ο οποίος είπε ότι η μηχανή εσωτερική καύσης θα αντέξει ακόμα 100 μέχρι 300 χρόνια, ιδίω δε ο ντίζελ, διότι επιτρέπει να εξοικονομούνται ε, καυσαέρια διοξιδίου του άνθρακος. Έτσι λοιπόν, αν ακούσουμε τους τεχνικούς, υπάρχουν εμπειρογνώμονες που λένε ότι μέσα σε 14 χρόνια, με το 2030 δηλαδή, βεβαίως και μέχρι τότε αλλά και για 100 χρόνια ακόμα θα έχουμε κοντά μας τον κινητήρα εσωτερικής καύσεως. Σα συγχαίρω γιατί όντως ανα... ανακαλύψατε ότι δεν είμαι τεχνικός, όντως και το μέλλον θα δείξει. Όμως σε κάθε περίπτωση πιστεύω πως τα αυτοκίνητα diesel που θα δίνουν καλά αποτελέσματα για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα και τηρούν και τα όρια για τα οξύδια του αζότου και υπάρχουν τεχνολογίες που αποδεικνύουν ότι είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Είναι δυνατόν οι κινητήρες να προσαρμοστούν να, να τηρήσουν και τι εκπομπέ οξυδίων του ΑΔΟΤΟ, τότε ε, πιστεύω θα συνεχίσει να εξελίσσεται η... το αντιζελοκίνητο αυτοκίνητο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζωγίνιο. Ο συνάδελφό σα τη προάλλε, στην τελευταία ακρόαση, με άφησε πολύ χαρούμενο γιατί ανέφερε πω η τεχνολογία σε αυτέ τι περιστάσει, με αυτά που διακυβεύονται για τον αριθμό των ανθρώπων ε, που πεθαίνουν πρώιμα, δεν μπορεί να μένει μόνο ένα αόριστο θέμα η τεχνολογία. Η Κομισιόν πρέπει να μείνει ουδέτερη. Όμω ο γενικό διευθυντή για το περιβάλλον μπορεί να μείνει ουδέτερο. Εσείς ήσασταν παράγονο κλειδί στον καθορισμό τη Ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα είστε γενικό Διευθυντής για το περιβάλλον. Αυτό που κατέστε σαφέ ότι ε, ε, πρέπει να χειριστούμε το πρόβλημα συνολικά. Υπήρχαν εκπομπές πάνω από αυτές που εσείς ε, θέλατε. Θα βελτιώσουμε λοιπόν τον τρόπο μέτρησης και το κοινό κέντρο μελετών έκανε πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη. Αλλά δεν έγινε τίποτα όσον αφορά την προέλευση των εκπομπών. Τώρα, όπως γενικός, σαν Γενικός Διευθυντής του Περιβάλλοντος, είπατε ναι, μια ανεπιστολή προς τις πόλεις, ότι είναι σημαντικό να βελτιωθούν τα συστήματα κινητικότητας. Δεν θα έπρεπε να στέλνετε και μια τέτοια επιστολή στις κατασκευαστές που να λέει ότι πρέπει να βελτιώσουν τα τεχνολογικά συστήματα τους ώστε να μειωθούν τον οι Κάπως ανησυχώ, δηλαδή δεν μπορούμε να βασιστούμε στον Γενικό Διευθυντή του Περιβάλλοντος ώστε να υπάρχει περισσότερη ηλεκτρική κινητικότητα και καθαρή κινητικότητα στην Ευρώπη. Ναι, βεβαίω, Και σας διαβεβαιώ ότι ο Γενικός Διευθυντής για το περιβάλλον αυτή τη δουλειά θα κάνω. Θα καταθέσω προτάσεις για καθαρό περιβάλλον. Ε, άλλωστε αυτό ε, έλεγα και στην επιστολή μου με τις απαντήσεις. Βεβαίως εδώ έχω δύο ιδιώτες γιατί δίνω μαρτυρία και ως πρώην Γενικός Διευθυντής για τις επιχειρήσεις. Λοιπόν, για την ερώτηση σχετική με την αυτοκινητοβιομηχανία συμφωνώ ότι θα μείνουν ε, κοντά μας για πολλά ακόμα χρόνια και πρέπει να εξασφαλίσουμε τα δρόμο δυνατόν πιο καθαρά. Άλλαξαν οι κανόνε για τη μέτρηση. Γιατί μόνο αυτοί οι κανόνε, και άλλου είδου ε, κανόνε μπορούν να τα στάνταρ καταμέτρηση, ναι, αλλά από τη στιγμή τη κατασκευή του οχήματο. Ναι, μπορούμε να αλλάξουμε ε, τα στάνταρ, αλλά πρέπει και να από τη στιγμή που θα ορίσουμε τους προσανατολισμούς, δεν πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις Βρυξέλλες, από το τμήμα του περιβάλλοντος, μπορούμε να πούμε στους κατασκευαστές το τι είδος αυτοκίνητα πρέπει να κατασκευάσουν, ούτε καν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο μάλιστα. Βλέπουμε ότι προχωρούν προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα υβριδικά αυτοκίνητα, ε, το βλέπουμε και στις, πόλεις, και στις πόλεις ε, και στις δημόσιες μεταφορές και μέσω των προγραμμάτων για την πρόθεση των καθαρών μέσων ε, κυκλοφορίας για την κυκλική οικονομία και οι καθαρές μεταφορές είναι πολύ σημαντικές που μπορούν όμως να γίνουν σιγά σιγά. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να δουλέψουμε και να προσφέρουμε πρωτευουλίες και και πρέπει να δουλέψουμε για τη βελτίωση του αέρα στις πόλεις. Ναι, αλλά τι, σε 10... Χάσατε δέκα χρόνια. Δέκα χρόνια χαμένα. Κοιτάξτε, όπως είμαι τώρα γενικό Διευθυντής για το Περιβάλλον εδώ και ένα χρόνο, να σας πω ότι είμαι αισιόδοξο. Ε, ε, δεν πήγαν χαμένα τα δέκα χρόνια, όχι. Ο κύριος Γκίζικε πάλι. Ευχαριστώ. Κύριε Καγιάχα, επανέρχομαι στην επιστολή που έχουμε ξανασυζητήσει της 19ης 11 του 2014 από τον κύριο Φάλκενμπεργκ προς εσάς όπου διαλαμβάνει διάφορα περί των ε, τρόπων ε, ε, τροποποίησης των μετρήσεων. Εκεί περιλαμβάνεται ή αναφέρεται και ένα συνημένο, το οποίο δεν σας έφτασε ποτέ ή πάντως σας έφτασε με μια καθυστέρηση των 10 μηνών. Μιλούμε τώρα για βελτιωμένη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μιλούμε για επικοινωνία και βλέπουμε τώρα ότι δέκα μήνες καθυστέρησε ένα συνημένο. Πώς μπορείτε να το εξηγήσετε. Εγώ ίδιος προσπάθησα να βρω μια εξήγηση, όμως δεν την βρήκα ήταν ένα παράρτημα το οποίο προσθέθηκε ένα χρόνο μετά και δεν το έλαβα ποτέ. Ζήτησα και εξηγήσει και όντω πιστεύω πω θα έπρεπε να γίνονται καλύτερα τα πράγματα. Όμω αυτό το παράρτημα δεν το έλαβα ποτέ, προσθέθηκε ένα χρόνο μετά και αυτό είναι πραγματικά ξεθρύνητο. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Επανέρχεται ο Θα πρέπει εγώ να ζητήσω συγγνώμη τώρα απέναντι στου ακροατέ σα διότι στην εισαγωγή σας κύριε Καγέχα μιλήσατε για τα BEMS και την αποτελεσματική εποπτεία και εκτός από τις μετρήσεις RDE καθώς μιλήσατε επίσης και για φορητά μηχανήματα μετρήσεων. Αυτά που μας είπαν όμως οι εμπειρονόμενες εδώ είναι ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκρίσεις μέχρι και 20%. Εν τέλει εμείς θέλουμε τις πραγματικές τιμές και όχι απλά να τις έχουμε, αλλά θέλουμε και καθαρό ατμοσφαιρικό αέρα. Πότε μπορούμε να περιμένουμε τέλος πάντων αξιόπιστες μετρήσεις από αυτά τα συστήματα BEMS. Πιστεύω πως η μελέτη του Κενού Κέντρου Μελετών του 2013 είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί εκεί εξετάζονται τα πλανεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων συστημάτων και από την τεχνική άποψη πιστεύω πως ε, το σύστημα των φορτών συσκευών είναι το καλύτερο. Γιατί το PEMS γιατί θα μας δώσει τις πραγματικές κομπές σε συνθήκες οδήγησης του αυτοκινήτου. Μέσα από αυτήν την τεχνολογία θα μπορέσουμε να μάθουμε ποια είναι η πραγματικότητα των εκπομπών για κάθε αυτοκίνητο. Με το σημερινό σύστημα, με τους τέσσερις αστικούς κύκλους και τον κύκλο εκτός πόλης, Είχαμε πολλές περιπτώσεις που μέναν ακάλυπτες στο εργαστήριο και υπήρχε η πιθανότητα να περάσουν τα αυτοκίνητα το ειδοκιμή και μετά στην πραγματικότητα να έχουν μεγαλύτερες εκπομπές γιατί ο κύκλος ελέγχου δεν ήταν αντιπροσωπευτικός. Όταν εξετάζει κανείς τα πλονεκτήματα του συστήματος PEMS, του φορητού συστήματος, το κοινό κέντρο μελετών, και αυτό τελικά ενέκριναν και τα κράτη ε, το κέντρο μελετών λοιπόν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι θα μας επιτρέψει να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί και θα είναι η Ευρώπη η πρώτη περιοχή του κόσμου που θα θέσει εφαρμογή αυτό το σύστημα. Και το σύστημα αυτό θα είναι ευρωπαϊκό πρότυπο. Μπορεί να μας ακολουθήσουν και άλλοι. Αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, το NEDC το ακολουθεί η Κίνα, η Ινδία, η Κορέα και η Ρωσία. Αν η Ευρώπη προχωρήσει στο PEMS θα θεσπίσουμε παγκόσμιο πρότυπο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό από τη βιομηχανική προοπτική. Ε, αλλά κυρίως από την προοπτική της υγείας των ανθρώπων. Θα καταφέρουμε να μην συμβαίνει αυτό που γινόταν, ότι δηλαδή να υπάρχει υπερβολικές εκπομπές γιατί το τεστ ήταν τελείως ξεπερασμένο. Σαλντιμόζε. Ναι, ευχαριστώ. Είμαι μια από τους τελευταίους μιλητές και θα προσπαθήσω να διατυπώσω και μερικά συμπεράσματα από όσα υπόθηκαν σήμερα. Ε, από ό,τι καταλαβαίνω δηλαδή, θεωρείτε ότι η Επιτροπή δεν έχει διαπράξει κανένα σφάλμα στο παρελθόν και ότι ήταν ευθύνη των κρατών μελών. Τα πάντα. Δεν έχετε όμω αυτή τη στιγμή να εκφράσετε λύπη, να πείτε ότι θα, έχετε, θα είχατε κάνει κάτι διαφορετικό ξέροντα αυτά που ξέρετε τώρα. Σα ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, γιατί δεν ισχυρίζουμε ότι ό,τι κάναμε ήταν σωστό και δεν διαπράξαμε κανένα σφάλμα. Ε, σας είπα ότι αισθάνθηκα ε, κατάπληξη αλλά και οργή όταν ξέσπασε το σκάνδαλο Volkswagen και λυπούμουν, λυπούμουν και λυπάμαι που δεν είχα παραπάνω εξουσίες γιατί η νομοθεσία δεν μας επέτρεπε να προχωρήσουμε περισσότερο. Το σύστημα λειτουργεί με μια διάκριση αρμοδιοτήτων και ευθυνών, τα, η αυτοκινητοβιομηχανία καλείται να, υλοποιεί την, να προσαρμόζεται στην νομοθεσία, τα κρατη να επιτηρούν, η Επιτροπή από μακριά. Και λυπούμε ιδιαίτερως που δεν είχαμε τη δυνατότητα να παρεύουμε. Πολύ θα ήθελα να είχαμε παρέμβει γιατί ε, διακυβεύτηκε η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας. Δεν ε, αισθάνομαι λοιπόν καμία ικανοποίηση ω Ευρωπαίο και ιδιαίτερα ω Γενική Διεύθυνση για τι επιχείρησει του τομέα αυτό. Αλλά ήταν δύσκολο να κάνουμε κάτι περισσότερο δεδομένων των συνθήκων. Και θα ήθελα να σα ρωτήσω όμω, λέει η κυρία Σουαλντεμόζερ, ε, το είπε και ο κύριο Φάλκενμπερκ νωρίτερα, ότι χρειάζεται μια ευρωπαϊκή υπηρεσία που θα έχει μια εποπτεία τη κατάσταση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εποπτεία της αγοράς σε ευχερέστερους όρους, γιατί γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει επαρκής ε, εποπτεία της αγοράς. Γιατί λοιπόν να μην προτείνει η Επιτροπή η υπηρεσία, αφού ξέρουμε ότι είναι μια από τις λύσεις για να αποφευχθούν νέα σκάνδαλα. Είναι πολύ σημαντική η παρατηρή σας. Θα συνεχίσω στο συλλογισμό μου με την απάντηση στην ερώτηση σας. Ένα από τα σφάλματα που διαπράξαμε επίση ήταν ότι περισσότερο ε, εστιάσαμε την προσοχή μας στην τροποποίηση τη νομοθεσία και είχα συναδέλφου που αγωνίζονταν και διαβάζανε και μελετούσαν και προσπαθούσαν να βρουν συμβασιστικέ λύσεις και τροπολογίες και πήγαιναν από την ε, ομάδα για τι εκπομπές ε, στην ομάδα για την αυτοκινητοβιομηχανία που συνομιλούσαν με κράτη-μέλη και το καθεξή. Αλλά εξίσου σημαντικό για να αλλάξουν τα πράγματα είναι η εποπτεία τη αγορά. Ε, σε σχέση με μια υπηρεσία εναλλακτικέ υπάρχουν. Γιατί για την υπηρεσία, ξέρετε, χρειάζεται πολιτική συμφωνία, πολιτική βούληση. Στο παρελθόν, στι μεγάλε κρίσει στι μεταφορέ, διατυπώνονταν από την Επιτροπή προτάσει για υπηρεσία. Μετά το ΕΡΙΚΑ, μετά το Πρεστής, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για, τις μεταφορές, για την ασφάλεια των θαλασσιών μεταφορών, από την κυρία Λογιόλα Τεπαράσου, παραδείγματι, το ίδιο και με την ΕΖΑ. Αλλά αλλά δεν χρειάζεται απαραίτητα. Αυτό που είπατε χρειάζεται ένας ανεξάρτητος μηχανικός εποπτείας. Μπορεί να γίνει από την Επιτροπή, μπορεί να γίνει από μια Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Ναι, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, γιατί ασχολούμαι με την ιστορική χώρα δέκα χρόνια τώρα του Ευρωβουλευτή και είναι τόσο η τομή που βλέπουμε να μην υπάρχει επαρκής εποπτεία της αγοράς από πλευράς των κρατών μελών. Δεν μας προτείνεται λοιπόν ούτε καν υπηρεσία, αλλά ούτε καν συγκεκριμένο στόχο για το βαθμό υλοποίηση αυτής τη εποπτείας αγορά από το κράτη-μέλη έστω. Δεν υπάρχει κάποια μετρήσιμη πρόταση. Ναι, βεβαίω και με την πρόταση για την αναθεώρηση του, της έγκρισης τύπου, έστω και χωρίς υπηρεσία ευρωπαϊκή, έχουμε πολύ Δυνατότητε γιατί δίνουμε και στην Επιτροπή τη δυνατότητα τη διερεύνηση, επιβολή κυρώσεων, ε, επιβολή τη εφαρμογή νομοθεσία, ε, προσφυγέ και όλα αυτά. Έχουμε ένα πολύ γερό μηχανισμό δηλαδή προβλέψει. Και χωρί πάλι υπηρεσία, δεν θα σα ξαφνιάσω φαντάζομαι, ε, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υφιστάμενη υπηρεσία. Έχουμε την Κοπενχάγη. υπηρεσία πρώτη γενναία. συλλέγει στοιχεία, έχει εξουσίε κοινό ερευνητικό κέντρο με την πραγματογνωμοσύνη την τεχνική που διαθέτει μπορεί να διαδραματίσει ρόλο. Περισσότερη πραγματογνωμοσύνη μπορούμε να εξασφαλίσουμε και σε επίπεδο επιτροπή, σε παραδείγματι, για την ασφάλεια των αέριων Έχουμε μια μονάδα επιθεωρητών που επισκέπτονται τα αεροδρόμια, αλλά χρειαζόμαστε πόρου. Με την κατάσταση όπω την αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, αυτά τα καθήκοντα δεν μπορούν να τα αναλάβουν οι υπηρεσίε μα. Ευχαριστώ. Η επόμενη ομιλητρία πρόεδρε δεν έχω καμιά άλλη ερώτηση, έχω καλυφθεί τις προηγούμενες απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Επομένως ακούσουμε τους συζητητές μας. Ο κύριος Σάλβα πρώτα. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καγιέχα για όλες τις λεπτομέρειες που... και τις ευκρινήσεις που μας δώσατε σήμερα. Υπάρχει όμως ε, μια ερώτηση που, ένα θέμα που πολύ με εγκαλεί με βάση τα όσα εξέτασε το Διεθνές ε, Συμβούλιο Καθαρών Μεταφορών, γιατί εκεί λέει ότι είναι 20 πλάσια η υπέρβαση των νόμιμων ορίων. Πώς γίνεται αυτό κύριε Καγιέχα? Και αυτό έχει que aclararlo, porque se ha dicho reiteradamente cómo era posible que superaran 20 veces. El estudio del ICCT se hizo sobre 15 coches, 12 aprobados en la Unión Europea y 3 en Estados Unidos. Los coches que sobrepasaban 20 veces τα αυτοκίνητα που ξεπερνούσαν 20 φορές ήταν τα αμερικανικά, όχι τα ευρωπαϊκά. Τα, τα ευρωπαϊκά Είμαστε σε ένα μέσο όρο τεσσάρων φορών, τετραπλάσιων εκπομπών δηλαδή, που είναι πολύ μεγάλη υπέρβαση, αλλά ε, δεν είναι 20 πλάσια τουλάχιστον. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι λοιπόν. 20 πλάσια εκπομπές είχαν τα αυτοκίνητα που εγκρίθηκαν στην Αμερική, στη ΣΥΠΑ. Και ξέρετε ότι εκεί τα όρια εκπομπών είναι πολύ πιο αυστηρά. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η ένταξη αυτών, ότι μάλλον εντάσσοντας αυτά τα αυτοκίνητα που υπερέβαιναν 20 φορές το όριο, ε, ανέβασε το μέσο όρο. Ανέβηκε ο μέσος όρος. Πάντως είναι αλήθεια ότι αυτά όλα τα αυτοκίνητα ξεπερνούσαν τα όρια στις πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Ε, αυτή η μελέτη διαβιβάστηκε αμέσως στις Εθνικές Αρχές και μάλιστα συζητήθηκε το Μάρτιο του 2014 στην Επιτροπή ε, για των Πραγματικών Εκπομπών για να μπορέσουν τα κρατημέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Πάντως, οι κοσαπλάσεις ήταν εκπομπές από τα αυτοκίνητα που εγκρίθηκαν στη ΣΥΠΑ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν σημαντική αυτή η διευκρίνηση. Γιατί όμως ε, αποκαλύφθηκε αυτό στη ΣΥΜΠΑ. Κοιτάξτε, εντάξει, για το γυροφέρνω με αυτό το θέμα όλη την ώρα. Η ΣΥΠΑ είναι μια χώρα. Εμείς είμαστε 28. Η ΣΥΠΑ έχουν ένα πράγμα που λέγεται ΕΠΑ. Μπορεί να έχουν, μπορούν να έχουν πρόσβαση στους κατασκευαστές και μπορούν να κάνουν έρευνες. Ε, έχουν 300 ε, μηχανικούς που εργάζονται στην ΕΠΑ. Εγώ να είχα 10 μηχανικούς και έκαναν τα πάντα. Ε, νομοθεσία, έλεγχο, παρακολούθηση της, των συζητήσεων και όλα. Είπα, είχαν την υποχρέωση στον παραγωγό να δηλώνουν αυτό το είδος τα λογισμικά. Εμείς εδώ δεν το είχαμε κάνει. Υπάρχει στη ΣΥΠΑ ένα σύστημα αυτοδήλωσης και ένα σύστημα, ένα καθεστώς εταιρικής ευθύνης πραγματικά δρακόντιο. Ενώ εμείς έχουμε τις αρχές, εθνικές αρχές έγκρισης και με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη γίνεται και αμοιβαία αναγνώριση. Υπάρχουν πολλοί και διάφοροι λόγοι στους οποίους οφείλονται όλα αυτά και επανερχόμαστε λίγο σε αυτά που είπαμε. Ότι πρέπει να ενισχύσουμε το ευρωπαϊκό σύστημα, να το ολοκληρώσουμε περισσότερο και να έχουμε πιο ισχυρούς μηχανισμούς υποπτίας. Δεν μπορώ να το πω γιατί θα μου ορμήξει κάποιος ευρωβουλευτής, αλλά πιστεύω πως θα πρέπει να προχωρήσουμε προς μια Ομοσπονδιακή Ευρωπαϊκή Αρχή. Αλλά δεν το λέω, δεν το λέω, είναι προσωπική μου γνώμη, δεν είναι η άποψη της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Κύριε. Λόπε Βερμέχο, ίσως αυτό το τελευταίο είναι το μόνο στο οποίο συμφωνούμε, κύριε Καγέχα μου. Πάντως η αλήθεια είναι εγώ πρώτα τώρα ανησυχώ περισσότερο από ό,τι στην αρχή. Κυρίως γιατί ήταν όλα γνωστά, ε, οι εταιρείε κάνανε ό,τι θέλανε, περάσαν αποφάσεις και με βάση ε, μία κρίση για τις αποφάσεις την καλή πίστη, την κακή πίστη των, ε, των χωρών. Χωρίς πραγματικά να έχει γίνει έλεγχος για το αν σωστά εφαρμοζόταν η νομοθεσία. Οι αποφάσεις όμως αυτές θα πρέπει να είναι οι πιο απλές, γιατί αυτές δίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα και σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον ε, απεφεύχθη το πιο απλό και το πιο εύκολο. νέοι μηχανισμοί, προσαρμογές που δεν λέω ότι δεν είναι απαραίτητα, αλλά αντί να έχουμε αυτό, να έχουμε το πιο απλό, Ήταν το πιο απλό να δούμε αν υπήρχαν παραβιάσεις ή μη τήρηση της νομοθεσίας να διερευνηθούν όλα αυτά τα στοιχεία. Διαφορετικά, αν οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνουμε βασίζονται στην καλή πίστη, πραγματικά κύριε Καγέχα, πολύ πολύ ανησυχώ για το τι θα γίνει. Ό, όχι, εγώ δεν νομίζω πως θα πρέπει να ανησυχείτε καθόλου. Διότι όταν κανείς εργάζεται στο Ευρωκοινοβούλιο και γνωρίζει τις ευρωπαϊκές συνθήκες, γνωρίζει πως βασίζονται στην αμοιβαία αρχή, που είναι θεμελιώδης αρχή της ε, υποχρέωσης συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη και, τις αρχές, και, και τους θεσμούς της Ένωσης. Αυτή είναι η μία θεμελιώδης αρχή. Όταν συνεργάζονται λοιπόν όλοι αυτοί, κράτη-μέλη και θεσμοί, αντιμετωπίζονται τα προβλήματα. Ποτέ δεν θα μπορούμε να έχουμε την ασφάλεια ότι κάποιος δεν παραβιάζει την νομοθεσία. Γίνεται καθημερινά και σε όλα τα πλαίσια, σε όλους τους τομείς. Αυτό που πρέπει να έχουμε είναι δυνατότητες επιβολής κυρώσεων και δυνατότητες ενίσχυσης της νομοθεσίας. Από πλευράς της Κομισιόν εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να εκτελούμε αυτά που μας ζητά το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών κάθε φορά και αυτά που έχουν συμφωνηθεί μέσα σε αυτή τη ε, διαδικασία ΚΑΡΣ 2020, 2020 ήταν να αλλάξουμε το σύστημα. Όμως δεν σταθήκαμε σε αυτό. Έχουμε ταυτόχρονα υποβάλει προτάσεις ώστε να καταφέρουμε να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς εποπτείας. Τη μεταρρύθμιση του type approval που έχετε επιτάπητος και που σας δίνει την ευκαιρία, αν υπάρχει απαρκής πολιτική βούληση, να ενισχύσετε το σύστημα εποπτείας. Αυτό μπορώ να σας πω. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ντέλη, τελευταία. Κύριε Καγιάχα, ε, επικαλυστήκατε νωρίτερα την Αμερικανική νομοθεσία, η οποία όμω είναι λιγότερο αυστηρή από την Ευρωπαϊκή, γιατί δεν κάνει λόγο για την συνήθη χρήση ή κανονική χρήση. Απλώς απαγορεύει τους μηχανισμούς αναστολής. Και όμως, και αυτό είναι που δεν καταλαβαίνω, την επαύριο της έκδοσης δημοσίευσης έκθεσης ISDT, οι Αμερικανοί το 2014 ξεκινάνε μια έρευνα. Εδώ γιατί δεν γίνεται τίποτα. Γιατί εμείς πρέπει να φτάσουμε το Σεπτέμβριο του 2015 για να κινηθεί επιτέλους κάτι. Και εσείς ως Γενικός Διευθυντής της Enterprise, τι σκοπεύετε να κάνετε για την αναπροσαρμογή των αυτοκινήτων. Σε αυτό νομίζω κανείς δεν θέλει να συζητήσει. Αλλά κύριε Καγιαχά, στείλαμε χιλιάδες εργαζομένους μισθωτούς σε αυτή τη βιομηχανία του παρελθόντος που είναι το ντίζελ. Ξέρω ότι θα μου απαντήσετε πως δεν έχουμε κάτι καλύτερο. Έχουμε όμως ένα πλεονέκτημα. Ξέρουμε, έχουμε την τεχνολογία και για τα υβριδικά και για το αέριο, πολλές τεχνολογίες για τα αυτοκίνητα. Γιατί λοιπόν να μην γίνει αυτή η αναμετατροπή. Και να πούμε στην αυτοκινητοβιομηχανία, κοιτάξτε, πέσαμε τα μούτρα στον τοίχο, τώρα πρέπει να κάνουμε όπισθεν. Γιατί τα πρώτα θύματα ήταν οι μισθωτοί. Α σταματήσουμε να λέμε το πρόβλημα Volkswagen, ε, ε, εκβιασμοί για την απασχόληση κτλ. Εάν δεν κοιτάξουμε αυτή την, την ουσία τη υπόθεση, πολύ θα δυσκολευτούμε. Πολλό δε μάλλον που σήμερα γίνεται λόγο για επενδύσει και οι επενδύσει ξέρουμε πολύ καλά που πρέπει να γίνουν. Και αν αύριο ντίζελ δεν υπάρχει και στις δημόσιες μεταφορές και στην αναμετατροπή των οχημάτων υπάρχει το δυναμικό που μπορεί να μας επιτρέψει αυτές τις επενδύσεις. Αυτό το έχετε λάβει υπόψη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντελή και ιδιαίτερος ευχαριστώ για τα μελήματα που εκφράζει αυτή η ερώτηση και τους προβληματισμούς, γιατί τους συμμερίζομαι και εγώ, σε σχέση με τα αυτοκίνητα που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά για το οποίο υπάρχουν προβλήματα. Ο κύριος Βέλα, Επίτροπος Αρμόδιος για το Περιβάλλον, ε, απίφθινε στην κυρία Πιετκόψκα και μάλιστα έδωσε μια ακρόαση στο Κοινοβούλιο, ε, γιατί τον είχε ρωτήσει τι μέτρα θα μπορούσαν να προβλεφθούν. Δεν είναι ευχερήση. Ε, κατάσταση, αλλά και ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, αυτοκίνητα που ξεπερνούν τα όρια και πρέπει να προβλεφθούν λύσεις. Πρόκειται για ένα τομέα στον οποίο, τον, οποίο επεξεργάζεται, στον οποίο επεξεργάζεται λύση επιτροπή. Σε σχέση με καθαρές λύσεις μεταφορών, και εσείς πολύ σωστά αναφερθήκατε στις κοινωνικές συνέπειες. Είναι όντω μεγάλες οι συνέπειες για τους εργαζομένους μας και έχουμε πιστεύω την ευκαιρία με το ανακοινωθέν για τις καθαρές μεταφορές να ε, θεσπίσουμε ένα πλαίσιο συζήτησης. Μιλήσαμε για το ΚΑΡΣ 2020 σήμερα εκτεταμένως. Υπάρχει εντωμεταξύ νέα πρωτοβουλία για την οποία είναι σημαντικό πιστεύω και εσείς να συμμετάσχετε κάποιοι συναδελφοί σας το Gear 2030. Πρέπει όλοι μαζί να φροντίσουμε μαζί με την αυτοκινητοβιομηχανία να βρούμε λύσεις και αηφορίας και βιωσιμότητας. Και πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για να βρούμε λύσεις. Μαζί με τη βιομηχανία, τους εργαζομένους, τους ενδιαφερομένους όλους. Ας κοιτάξουμε λοιπόν μια λύση. Και με αυτά τα ολίγα. Κύριε Καγιάχα, τελειώνουμε, κλείνουμε. Έμαθα ότι έχετε και γενέθλια σήμερα, χρόνια σας πολλά. Μεγάλη μέρα. Ενημερώστε λοιπόν παρακαλώ όποιο θέλει. Η επόμενη συνεδρίαση 24 Νοεμβρίου. Με την κυρία Σεγκολέν Ρουαγιάλα, Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας της Γαλλικής Δημοκρατίας.